Bonjour tout le monde. Nous allons commencer la réunion. Καλημέρα σε όλους. Να ξεκινήσουμε την συνεδρίασή μας, να ξεκινήσουμε με την ημερήσια διάταξη. Υπάρχει μια αλλαγή στην ημερήσια διάταξη. Οι συντονιστές αποφάσισαν να βγάλουν την εμεσία διατάξη στα σημεία 7 και 15 πρωτοβουλίε για προφορική ερώτηση ώστε να ασχοληθούν με το θέμα τη σεξουαλική βία σε τρίτε χώρε και την καταπολέμησή τη βεβαίω, κάτι που προβλεπόταν για τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Όμω, μάθαμε το μεταξύ ότι η Επιτροπή των ε, Δικαιωμάτων των Γυναικών συνέταξε μια προφορική ερώτηση προ το Συμβούλιο και την Επιτροπή <clears throat> για το ίδιο θέμα για την Ολομέλεια του Νοεμβρίου επί τη ευκαιρία της Διεθνούς ημέρας της βίας εις βάρος των γυναικών στις 25 Νοεμβρίου. Αντί λοιπόν να περάσουμε σε, μια, σε έναν ανταγωνισμό για την πρωτοβουλία αυτή, ας προσπαθήσουμε <clears throat> να ευστήσουμε την προσοχή στην αναπτυξιακή διάσταση του όλου ζητήματος. Η Επιτροπή έθεσε ερώτηση προς το Κοινοβούλιο ή μάλλον ζήτησε από το Κοινοβούλιο να διευρυνθεί συζήτηση προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα τα μέλη και οι πολιτικές ομάδες καλούνται να συμμετάσχουν στην όλη συζήτηση κατά την Σύνοδο της Ολομέλειας του Νοεμβρίου και να συμμετάσχουν στη σύνταξη ψηφίσματος που ετοιμάστηκε από την Επιτροπή των Δικαιωμάτων των Γυναικών. Υπάρχουν ενδεχομένω άλλε παρατηρήσει για την ημερήσια διάταξη. Εάν όχι, την εγκρίνουμε. Εγκρίνουμε και τα πρακτικά της συνεδρίασης της 9ης Οκτωβρίου. 19ης μάλλον Οκτωβρίου. Θα τα δείτε στο πακελό σας. Εάν έχετε παρατηρήσεις παρακαλούμε Ενημερώστε τη γραμματεία σχετικά πριν το τέλο τη συνεδρίαση. Αν δεν ληφθούν, παραληφθούν παρατηρήσει, θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται και τα πρακτικά. Θα θυμάστε μάλλον ότι είχαμε προεδρικές εκλογέ στο Αφγανιστάν στις 20 Αυγούστου φέτο. Η Επιτροπή μας αποφάσισε να προσκαλέσει τον ειδικό εκπρόσωπο του ΟΗΕ για το Αφγανιστάν, τον κύριο Καϊάιντε, και επειδή ακυρώθηκαν σε μια πρώτη φάση οι εκλογές στο Αφγανιστάν, δεν προσήλθε, όμως τώρα μας επιβεβαίωσε ότι μπορεί να έλθει για να συζητήσει μαζί μας και ακριβώς αυτό θα συμβεί στις 16 Νοεμβρίου, από τις 5.30 μέχρι τις 7.30. Θα πληροφορηθείτε προσεχώς σε ποια ακριβώς αίθουσα. Ήθελα επίσης εξ ονόματος της Προεδρίας να χαιρετήσω την απόφαση του ΟΗΕ η οποία ενέκρινε την έκθεση Goldstone. 114 ψήφισαν υπέρ, 18 κατά και υπήρξαν και 44 αποχές. Έτσι λοιπόν προσεκλήθησαν και το Ισραήλ και την Παλαιστίνη να διενεργήσουν έρευνες για τις σοβαρότατες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διπράχθησαν κατά την ε, σύραξη στη Γάζα στις αρχές της φετινής χρονιάς, τον πόλεμο της Γάζας. Προσκαλέσαμε τον κύριο Γκόλστον, ο οποίος αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας λοιπόν και ελπίζουμε να μπορέσουμε να τον δούμε κατά τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Η Επιτροπή έχει κάτι να ανακοινώσει. Μάλλον όχι. λάβαμε ερώτηση από τον κύριο Μπέρμαν που αφορά την βοήθεια προς το Σουδάν. Η ερώτηση αυτή μοιράστηκε στα μέλη, δεν θα την αναγνώσω, αλλά θα δώσω ευθύς αμέσω το λόγο στην Επιτροπή που εκπροσωπεί ο κύριος Κρίσλερ. Σας ευχαριστώ. Όπως γνωρίζετε το Σουδάν απεφάσισε να μην κυρώσει την αναθεωρημένη συνθήκη Κοτονού μέχρι τις 30 Ιουνίου 2009 που προβλεπόταν. Η απόφαση αυτή λήφθηκε για να ενθαρρυνθούν οι χώρες και να λάβουν μέτρα για να θέσουν σε εφαρμογή το, την, ε, το πρωτόκολλο της Ρώμης και τα σχετικά ε, άλλα έγγραφα. Η μη κύρωση από το Σουδάν Σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν μπορεί να εφαρμόσει διμερή συμφωνία αναπτύξεως μέσα στα πλαίσια του 10ου ε, Ευρωπαϊκού Ταμείου με το Σουδάν. Και αυτό σημαίνει επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα μπορέσει να διαθέσει τα 300 εκατομμύρια ευρώ τα οποία υποσχέθηκε στο κονσόρτσιουμ ε, του Σουδάν το 2008 και για την περίοδο 2008 έως 2013. Πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα είναι υποχρεωμένη να πάυσει κάθε είδους αναπτυξιακή βοήθεια προς το Σουδάν. Χρηματοδότηση από την κοινότητα θα συνεχίσουν να αυξάνονται και τον επόμενο χρόνο αλλά και το 2011 στη βάση των προηγούμενων υποχρεώσεων από το 9ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αναπτύξεως κυρίως αυτές οι υποχρώσεις δεν επηρεάζονται από την νομική ε, κατάσταση που αντιμετωπίζουμε τώρα. Αυτό θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε τη χρηματοδότηση ε, προγραμμάτων τα οποία συνεχίζονται και έργων επίσης, για παράδειγμα στην εκπαίδευση, υγεία και αφοπλισμό, καθώς και ιδιαίτερα στο νότο του Σουδάν. Δεύτερο, η ευρωπαϊκή κοινότητα ε, αναζητεί τρόπους να διαθέσει Κάποιε χρηματοδοτήσεις τουλάχιστον προς το Σουδάν υπό την ισχύ άλλων μηχανισμών περιλαμβανομένων και από το ε, μηχανισμό σταθερότητας όχι από το Ευρωπαϊκό ε, ε, Όργανο Δημοκρατίας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων για να ενισχυθεί η συνολική Συμφωνία Ειρήνης και εφαρμογή της και ο εκδημοκρατισμός σε ολόκληρο το Σουδάν. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδέχεται να χρησιμοποιήσει υπό συγκεκριμένε προποθέσει και όρου και τον περιφερειακό φάκελο του EDF για θεματικά προγράμματα και στα πλαίσια του DCI. Τρίτο, η ανθρωπιστική βοήθεια θα συνεχιστεί όπως αυτό είναι αναγκαίο, όπου αυτό είναι αναγκαίο, διότι προέρχεται από διαφορετικό μηχανισμό και δεν ε, θίγεται από την απόφαση της κυβέρνησης Του Σουντάν. Τέλος, η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή άρχισε συζήτηση με τις, Ευρωπαϊκές, με τις χώρες μέλη στις Βρυξέλλες για να εξετάσουμε πώς μπορούμε να αποφύγουμε μια δραματική μείωση των χρηματοδοτήσεων υπέρ των πιο ε, ε, ευαίσθητων τροτών τμήματων του πληθυσμού του Σουδάν. Τέλος, η Κομισιόν έχει ήδη κάνει μια πρώτη εκτίμηση των συνεπειών της μη κύρωσης επιτόπου. Εξετάσαμε ιδίω τα πιθανά κενά τα οποία θα προκαλέσει επιτόπου η απόφαση αυτή στους διάφορους τομείς παρέμβασης μας όπως την αγροτική ανάπτυξη και την εκπαίδευση. Και υπενθυμίζω ότι αυτοί οι δύο τομείς πρόκειτο να είναι αυτοί στους οποίους θα δίδεται ιδιαίτερη έμφαση και υπό το δέκατο ε, πρόγραμμα. Αρχίσαμε και μια συζήτηση με τις χώρες μέλη στις αρμόδιες ομάδες εργασίας του Συμβουλίου για το θέμα αυτό. Το ερώτημα εδώ είναι πώς θα αντιδράσουν και οι άλλοι δωρητές και πώς θα μπορέσουν να προσαρμόσουν το προγραμματισμό τους στη νέα κατάσταση που προέκυψε. Και αυτό πάντως το εγχείρημα συνεχίζεται η Κομισιόν αναλαμβάνει πρωτοπόρο ρόλο διότι έχουμε λάβει υποχρεώσει απέναντι στον λαό του Σουδάν και δεν μπορούμε να αποδεσμευτούμε κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο, νομίζουμε, διότι επίκυνται εκλογέ τον Απρίλιο του 2010 στο Σουδάν, καθώ και δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία του Νότιου Σουδάν που προβλέπεται για τον Ιανουάριο του 2011. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για αυτή την απάντηση. Καταγράφουμε και στη μνήμη μας το πρόβλημα του Σουδανέζικου λαού και την έλλειψη 300 εκατομμυρίων βοήθειας εξαιτίας της μη κύρισης. Να καλωσορίσω τον κύριο Φίλιπ Μάιστατ, ο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Είναι μεγάλη μας χαρά να σας έχουμε σήμερα μαζί μας, διότι αυτή η συνεδρίαση τη Επιτροπής μας θα επικεντρωθεί στην χρηματοπιστωτική κρίση και τις επιπτώσεις της αναπτυσσόμενες χώρες. Η Επιτροπή αυτή ασχολείται ιδιαίτερω και με φορολογικά ζητήματα ω εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, γνωρίζετε ότι η τράπεζα αυτή θα μπορούσε να συνδράμει ιδιαίτερα στι αναπτυσσόμενε χώρε αυτή την περίοδο κρίση. Ένα άλλο λόγο που καλωσορίζω την παρουσία σα εδώ είναι ότι η, τράπεζα των, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, υπόκειται στην ενδιάμεση αναθεώρηση των εκτορικών αναθέσεων εργασιών τη, οι οποίε θα υπόκεινται και στη νέα διαδικασία συναπόφαση ε, που φέρνει σε συνεργασία το Συμβούλιο με το Κοινοβούλιο. Γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που μπορούμε να ακούσουμε τη συνεισφορά σα. Κύριε Μάιστατ, πρόεδρε Μάιστατ, έχετε το λόγο για 20 περίπου λεπτά. Merci, Madame la Présidente. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να ξεκινήσουμε μια νέα φάση διαλόγου με την Επιτροπή σας. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχω αυτή τη χαρά να βρισκόμαι στην Επιτροπή σας. Η τελευταία φορά βέβαια ήταν πριν από χρόνια, το 2005. Έκτοτε είχα επαφές με πολλά μέλη της Επιτροπής σας, αλλά είναι η πρώτη φορά από το 2005 που έχω την χαρά να μπορώ να σας συναντήσω διαζώσεις. Νομίζω ότι η στιγμή είναι κατάλληλη, διότι η Επιτροπή σας αναντήρητα θα έχει καθοριστικό ρόλο να διαδραματίσει στις συζητήσεις που θα ξεκινήσουν από το 2010 για τις εξωτερικές εντολές της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Για όσους από εσά δεν γνωρίζουν πολύ καλά πώς εργάζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, να θυμίσω σύντομα ότι αυτή η τράπεζα είναι η Τράπεζα των 100 Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημιουργήθηκε βάσει της συνθήκης της Ρώμης και στόχος της είναι βάσει της συνθήκης να στηρίζει οικονομικά και να επιδιώκει τους στόχους, αυτό που τότε ονομαζόταν η οικονομική κοινότητα της Ευρώπης. Σήμερα αυτοί οι στόχοι ονομάζονται στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε λοιπόν σήμερα 27 μετόχους, τα 27 κράτη-μέλη, και χρησιμοποιούμε τους πόρους, τους πόρους μας που δεν είναι πόροι του προπολογισμού αλλά από την οικονομική αγορά, τη χρηματοπιστωτική αγορά παγκοσμίω. Αυτούς τους πόρους που αντλούμε λοιπόν από τη χρηματοπιστωτική αγορά τους ε, χρησιμοποιούμε για να επιδιώξουμε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βάσει της, ε, λόγω της σημερινής κρίσης μας ζητήθηκε να αυξηθεί ο όγκος των ε, δανείων μας. Από 50 δις ευρώ που ήταν ο ετήσιος όγκος δανειοδότησης της ΕΤΕ και που την έκανε το σημαντικότερο χρηματοπιστωτικό οργανισμό διεθνώς, φέτος θα δανείσουμε 75 δις ευρώ. Όμως, εξορισμού να διευκρινίσω ότι από αυτά τα 75 εκατομμύρια, τα 70 προορίζονται για προγράμματα τα οποία θα διεξαχθούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή πάνω από το 90% των ε, δράσεων δανειοδότησης που οργανώνουμε προορίζονται για σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να παρέμβουμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά εκτός και αν υπάρχει κάποια εντολή. Εντολή η οποία θα μας δοθεί είτε βάσει διεθνούς συνθήκης, είτε από μια απόφαση και ω τώρα τέτοιε αποφάσει ελάμβανε το Συμβούλιο. Εντολή λοιπόν βάσει διεθνού συνθήκη όπω η συνθήκη Κοτονού. Αυτή είναι μια συνθήκη μεταξύ των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των χωρών ΑΚΕ. Βασίστηκε στι συμφωνίε Γιαουντέ και Λομέ και στη συμφωνία Κοτονού ανατέθηκε αποστολή στην ΕΤΕ να διαχειριστεί μια διευκόλυνση οικονομική για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα στις χώρες ΑΚΕ. Αυτή η εντολή ανατίθεται βάσει συνθήκης και μπορεί συγκεκριμένη να θεωρηθεί ως πραγματική αναπτυξιακή εντολή. Πέραν αυτού, λαμβάνουμε από το Συμβούλιο και άλλες εξωτερικές εντολές, όπου το Συμβούλιο καθορίζει ποιο είναι το μέγιστο ποσό του δανείου που μπορούμε να περάσουμε σε μια συγκεκριμένη περιοχή, γιατί τι είδου πρόγραμμα, βάσει ποιων προποθέσεων και αυτό ποικίλει από μια περιοχή του κόσμου σε άλλη. Δεν θα αναπτύξω τώρα όλε τι αναπτυξιακέ εντολέ που υπάρχουν, αλλά ουσιαστικά ο στόχο είναι να δοθεί οικονομική συνεισφορά για την επιδίωξη συγκεκριμένων στόχων. Η τελευταία τέτοια απόφαση ελήφθη το Δεκέμβριο του 2006 για την περίοδο 2007-2013 από το Συμβούλιο και όρισε εκεί το Συμβούλιο ένα ποσό, το θυμίζω εντάχει, η ΕΤΕ μπορεί να δανείσει κατά την περίοδο αυτή 2007-2013 8,6 δις για τις χώρες ε, πριν την ε, προσχώρηση, τις προενταξιακές χώρες, των Δυτικών Βαλκανίων δηλαδή, το ίδιο για τις χώρες εταίρους της Μεσογείου, το ίδιο ποσό, 3,7 δις, 3,7 μάλλον για τους γείτονες των, ε, στα Ανατολικά και τη Ρωσία, 8 περίπου δις για την, Αμερική, για την Λατινική Αμερική και επίσης ποσά για την ε, νοτιο, Νότια Ασία, Νοτιοανατολική Ασία και την Κίνα. Αυτά ήταν περίπου τα ποσά που αναφέρονταν για τη συγκεκριμένη περίοδο. Βέβαια το Συμβούλιο ε, διευκρίνησε σε αυτή την απόφαση ότι μπορούσαμε συγκεκριμένες επενδύσεις να επενδύσουμε σε κάθε περίπτωση. Στην Ανατολή, στα ανατολικά λόγου χάρη τεσσάρων ειδών προγράμματα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν σε τέσσερι συγκεκριμένου τομεί. Σε άλλε περιοχέ περιοριστήκαμε σε προγράμματα που ενδιαφέρουν τι ευρωπαϊκέ εταιρείε. Κάτι που δεν ισχύει παντού. Υπήρχε λοιπόν μεγάλη επικοινομορφία στι προποθέσει τη εντολή. Υπήρξαν δύο νέα στοιχεία βέβαια. Πρώτον, σε αυτή την απόφαση του Δεκεμβρίου 2006 το Συμβούλιο αποφάσισε ότι θα υπάρξει ενδιάμεση αναθεώρηση η οποία θα έπρεπε ουσιαστικά να γίνει το 2010. Το Συμβούλιο αποφάσισε ότι η, απόφαση, η αναθεώρηση αυτή έπρεπε να προετοιμαστεί από ομάδα σοφών ειδικών, μια ομάδα εννέα ατόμων η οποία συστήθηκε και θα προχωρήσει σε ανάλυση, μελέτη των δράσεών μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συντάξει κάποιες συστάσεις το δεύτερο νέο στοιχείο της απόφασης αυτής ήταν μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, διότι το Κοινοβούλιο προσέφυγε κατά της απόφασης του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2009, προσέφυγε θεωρώντας ότι η νομική βάση δεν ήταν η ορθή νομική βάση και ότι η απόφαση για τι εξωτερικέ εντολέ τη ΕΤΕ ήταν αρμοδιότητα όχι μόνο του Συμβουλίου αλλά και του Κοινοβουλίου. Πιο συγκεκριμένα, το Κοινοβούλιο θεωρούσε ότι έπρεπε να αναφερθεί κανείς όχι μόνο στο 181α άρθρο της συνθήκης, αλλά και στο 179 στο βαθμό που υπάρχουν ε, και αναπτυξιακές διαστάσεις στην εξωτερική εντολή αυτή της ε, ΕΤΕ. Οπότε έπρεπε να εφαρμοστεί η δικασία της αναπόφασης. Δικαιώθηκε από το ΔΕΚ το Κοινοβούλιο. Είπε το ΔΕΚ ότι πράγματι ο ορισμός της εξωτερικής εντολής της ΕΤΕ έπρεπε να προκύπτει από την ε, συνεργασία, την διαδικασία της αναπόφασης Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Εφαρμόστηκε λοιπόν αυτό στον επανακαθορισμό της συγκεκριμένη εντολής. Μεταβατικά, το Κοινοβούλιο, πριν τις πρόσφατες εκλογές, θέλησε να ανανεώσει την απόφαση που είχε ληφθεί από το Συμβούλιο, αλλά αυτό έγινε μόνο προσωρινά. Θα πρέπει λοιπόν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, δηλαδή το αργότερο τον Οκτώβριο του 2011, να υπάρξει συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου ώστε να επανακαθοριστεί η εξωτερική εντολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Νομίζω ότι θα είναι μια καλή ευκαιρία αυτή για να έχουμε μια διεξοδική συζήτηση για το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ΕΤΕ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένοντας ε, αυτή τη στιγμή να πω τι κάνουμε ως σήμερα και τι μπορούμε να προσφέρουμε σήμερα. Στι χρηματοδοτήσει εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, μπορούμε να προσφέρουμε την πείρα μα, την εμπειρογνωμοσύνη που έχουμε αναπτύξει εντό Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούμε να προσφέρουμε, να ε, επιτρέψουμε να αξιοποιήσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό θα μας επιτρέψει να δώσουμε την τεχνική μας γνώση σε ορισμένους τομείς. Δεν είμαστε μια συνηθισμένη τράπεζα έχουμε μεταξύ του προσωπικού μας έναν αυξημένο αριθμό μηχανικών λόγου χάρη που σε ορισμένους τομείς έχουν ε, συγκεντρώσει τέτοια εμπειρογνωμοσύνη που είναι σπάνια. Και αυτό θα μας επέτρεπε όχι μόνο να δώσουμε χρηματοδότηση στις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και τεχνική αρρωγή. Να βοηθήσουμε τους διαχειριστές των προγραμμάτων να βελτιώσουν την τεχνική ποιότητα και την οικονομική αποδοτικότητα των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν. Αυτό γίνεται σε τομείς όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, το νερό Υπάρχουν τουλάχιστον τρει τομεί όπου η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει αναπτύξει εμπειρογνωμοσύνη εντό Ευρωπαϊκή Ένωση αρχικά, αλλά που μπορεί πραγματικά να θέσει στην υπηρεσία των αναπτυσσόμενων χωρών. Το δεύτερο στοιχείο που μπορούμε να προσφέρουμε στι δράσει εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η οικονομική εμπειρογνωμοσύνη. Διότι έχουμε αναπτύξει μέσα ιδιαίτερα ποικίλα χρηματοδότηση και ιδιαίτερα ανεπτυγμένα στις δράσεις μας εντό Ένωση. Και αυτά λοιπόν μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωση. Εδώ λίγο πολύ η συνολική εικόνα των δράσεων της ΕΤΕ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας ζητήθηκε εάν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα εξαιτία τη ε, χρηματοπιστωτική κρίση που πλήττει ακόμη περισσότερο τις αναπτυσσόμενες χώρε από ό,τι τις αναπτυγμένες ε, αλλά δεν μπορέσαμε να αποκριθούμε σε αυτή την έκκληση για ένα πολύ απλό λόγο. Οι δυνατότητέ μα να δράσουμε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση περιορίζονται ακριβώ από την εξωτερική εντολή που έχουμε. Εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, μπορέσαμε αισθητά να αυξήσουμε τον όγκο τη δανειοδότηση και προ την κατεύθυνση που μα υποδι... από το Συμβούλιο από 50 δις περάσαμε σε 75 δις δανειοδότησης και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις προτεραιότητες που έχει ορίσει το Συμβούλιο, υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, προτεραιότητα στις περιφέρειες εκτός ε, αναπτυξιακού άξονα. Αυτό λοιπόν μας επέτρεψε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης να αυξήσουμε τον όγκο των επιχειρήσεών μας, των δρασεών μας. Αυτό όμως δεν ισχύει και για τα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι να απορρίψουμε κάποιες χρηματοδοτήσεις ακριβώς διότι προσεγγίζουμε τα όρια του χαρτοφυλακίου που αποφασίστηκαν από το Συμβούλιο. Ωστόσο, καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να συνεισφέρουμε στην καταπολέμηση αυτής της ε, κρίσης. Ε, συμμετέχουμε σε πρωτοβουλίες που έχουν ε, καθορίσει άλλοι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. Για να αναφέρω τρεις πρόσφατες τέτοιες πρωτοβουλίες, αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε στο Microfinance Enhancement Facility που ξεκίνησε το IFC, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η KW που είναι γερμανική φυγατρική προκειμένου να στηρίξουμε την ανάπτυξη των μικροοικονομικών επιχειρήσεων στις χώρες ΑΚΕ. Μια άλλη πρωτοβουλία πρόσφατη στην οποία αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε είναι το Infrastructure Crisis Facility για να στηρίξουμε σχέδια υποδομών, οικοδόμησης υποδομών από ιδιώτες, διότι η χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα για τις υποδομές είναι σημαντικότατο στοιχείο σε περίοδο κρίσης. Και εκεί λοιπόν πήραμε μέρος σε αυτή τη διεθνή πρωτοβουλία και αποφασίσαμε να συνεισφέρουμε ένα δις ευρώ συγχρηματοδότησης στον τομέα των ιδιωτικών υποδομών. Τέλος, Πρόκειται τώρα να αποφασιστεί η συμμετοχή μας στο African Bank Capitalization Fund και πάλι πρωτοβουλία που έλαβε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο στόχο έχει να στηρίξει τα χρηματοπιστωτικά, τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Αφρική. Μια πρόσφατη πρωτοβουλία στην οποία επιθυμούμε να συμμετάσχουμε στο γενικότερο πλαίσιο καταπολέμησης της κρίσης. Στο ίδιο επίπεδο Θέλουμε να αναπτύξουμε αυτό που ονομάζεται mutual reliance, αμοιβαία εξοπιστία, δηλαδή να μπορούμε να βασιστούμε περαιτέρω στο έργο που έχουν φέρει πέρα άλλοι οργανισμοί. Όταν προχωρούμε σε, χρηματοδο... σε συγχρηματοδότηση, διαπιστώνουμε ότι το ίδιο έργο πολλέ φορέ επαναλαμβάνεται από διάφορου οργανισμού που συγχρηματοδοτούν τελικά το ίδιο σχέδιο. Ε, όταν γίνεται μελέτη και ανάλυση και επαλήθευση κάποιων προποθέσεων περιβαλλοντικών και κοινωνικών που πρέπει να πληρούνται, Διερωτόμαστε στη συνέχεια πώς ε, συνήφθη μια σύμβαση, οπότε αυτό πολλές φορές σημαίνει ότι οι πόροι χρησιμοποιούνται ξανά και ξανά για τον ίδιο σκοπό από πολλούς ε, οργανισμούς. Και αυτό δεν έχει απαραίτητα ε, και χαμηλό κόστος για τον δικαιούχο. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να μην υπάρχει επικάλυψη των έργων μα με άλλου οργανισμού, αμοιβαίω κιόλα, και αυτό έχουμε ξεκινήσει να το κάνουμε με πιλωτικά προγράμματα, ιδίω με, με τον Γαλλικό Οργανισμό Ανάπτυξη και τον αντίστοιχο Γερμανικό Οργανισμό. Να προσθέσω ότι στο ίδιο πνεύμα συνεργασία με του ε, οργανισμού και του φορεί έχουμε στη Σύνοδο τη Κοπενχάγη ηγετικό ρόλο αναλάβει για τη σύνταξη μια κοινή δήλωση, joint statement των πολυμερών τραπεζών ε, επενδύσεων και την οποία πρόκειται να παρουσιάσουμε στην Κοπενχάγη για να δείξουμε ότι οι πολυμερείς τράπεζες επενδύσεων μπορούν να συνεισφέρουν ε, σαφέστατα στην ανάπτυξη βάσει και την κατευθύνσεων που θα αποφασιστούν στην Κοπενχάγη. Και σε κάθε περίπτωση με συστηματική συνεργασία μεταξύ των πολυμερών τραπεζών επενδύσεων ώστε να υπάρξει πρόοδο σε αυτό το τομέα. Τέλος, να επισημάνω ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κατέβαλε κάθε προσπάθεια για να υλοποιήσει την αρχή του G20 για τα offshore financial centers, τα εκτός τα offshore, τα οικονομικά κέντρα offshore, κάναμε μια πολύ ενδελεχή μελέτη για το κατά πόσον αυτός ο παράγοντας επένδυσης μπορούσε να, είναι, να έχει την έδρα του offshore και κατόπιν τη συνόδου του G20 δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε περαιτέρω διότι εδώ έχουμε επικεντρωθεί σε ένα κέντρο που βρίσκεται στο μαύρο κατάλογο του ΩΣΑ Προσωπικά διαρωτώ με βέβαια γιατί κάποιες χώρες δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το μαύρο κατάλογο για τη συγκεκριμένη χώρα δεν θα την κατονομάσω. Τέλος πάντων, για τις χώρες αυτές, όταν έχουμε κάποιον δανειολήπτη που βρίσκεται, έχει την έντρα σε αυτή τη χώρα, του ζητούμε να μετακινηθεί σε άλλη δικαιοδοσία. Εκτό τη χώρα αυτή που βρίσκεται στο μαύρο κατάλογο. Ιδού, Πρόεδρε, λίγο πολύ ποιε είναι πρόσφατε δραστηριότητε τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Νομίζω ότι σημαντικό είναι επίση να επισημάνω ότι Κατά τη διάρκεια του 2010 θα έχουμε διάλογο, συζήτηση για το ρόλο τη εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό που εμεί περιμένουμε από την πλευρά μα είναι διευκρινήσει. Να μα διαφωτίσετε. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θέλουν ή δεν θέλουν, συμφωνούν ή δεν συμφωνούν η ΕΤΕ να έχει ρόλο να διαδραματίσει στι αναπτυσσόμενε χώρε. Εάν η απάντηση είναι καταφατική, α μα δώσουν τον τρόπο τα μέσα. Να μας επιτρέψουν δηλαδή να προσλάβουμε το προσωπικό που χρειάζεται για να έρθει πέρα σε ένα τέτοιο αναπτυξιακό έργο και έπειτα να μας επιτρέψουν να υποφεληθούμε από συγκεκριμένου πόρους ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε και παραχωρητικά δάνεια. Διότι η ΕΤΕ, βάσει του καθεστώτος της, δεν μπορεί να επιχορηγήσει τα δικά της δάνεια. Αυτό μας είναι ρητός απαγορευμένο. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε τα επιτόκια της αγοράς. Ωστόσο, για τη χρηματοδότηση κάποιων προγραμμάτων στι αναπτυσσόμενε χώρε, ε, τα επιτόκια αυτά είναι ιδιαίτερα αυξημένα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε παραχωρητικά επιτόκια, κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε παρά μόνον εάν έχουμε χορηγήσει από, από τρίτα μέρη, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από τον προπολογισμό των κατώμελών, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε ανάγκη από τη συνδρομή τρίτων θα είμαι σαφής λοιπόν, εάν στο πέρας των συζητήσεων που θα έχετε με το Συμβούλιο την ερχόμενη χρονιά καταλήξετε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρέπει να διαδραματίσει ένα ρόλο αναπτυξιακής τράπεζας σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, να σα πω ότι ευχαρίστω να δεχτούμε την αποστολή αυτή, αλλά υπό την προπόθεση σε κάθε περίπτωση ότι θα υπάρξει συμφωνία για τα μέσα που μα χρειάζονται, ώστε να φέρουμε πέρα με τον ορθό τρόπο την αποστολή αυτή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Είστε σίγουρα καθοριστικός παράγοντας και για μας. 5 δις ευρώ είναι περισσότερα από όσα διαθέτει και η Αφρικανική Τράπεζα Επενδύσεων. Η Αμερικανική Τράπεζα Επενδύσεων είναι μεσομεντικά τα κονδύλια για την ανάπτυξη. Να δώσω τώρα το λόγο στους συναδέλφους. Ο κύριος Ντέβα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Μάστεντα στην Επιτροπή μας και η συγκυρία της επίσκεψης εδώ είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή στην έναρξη της ε, νέας αυτής ε, θα έλεγα θητείας με την ε, συναπόφαση που αποκτούμε με τη νέα συνθήκη της Λισαβόνας. Με μεγάλη ικανοποίηση σημειώνω πρέπει να πω ότι οι ανώτατοι στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προβληματίζονται να μετατρέψουν την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε μια αναπτυξιακή τράπεζα. Είναι μια συζήτηση που εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα διεξάγεται και χαίρομαι που γίνεται αυτή, λαμβάνεται αυτή η τροπή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε σχέση με τη μονάδα που είναι μια ήπια δύναμη και η ήπια δύναμη σίγουρα συνδέεται και με το ότι ε, χρήματα δίνουμε, δεν είναι θέματα στρατών ε, ή βομβών ε, και χρήματα τα οποία είναι δάνεια και δεν είναι φάπαξ χορηγίες, είναι λοιπόν πιστώσεις και φαίνεται σε σχέση με τον ελεγχόμενο, την ελεγχόμενη επιτυχία που θα θέλαμε να έχουμε υπάρχει αρκετό περιθώριο ενώ δανείζεται χρήμα στον ιδιωτικό τομέα και εκεί έχουμε διαφορετικό ήθος και λειτουργεί και δημιουργεί περισσότερο πλούτο και χρήμα ως ε, αντάλλαγμα. Αυτό λοιπόν εμείς πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Είναι κάτι θα έλεγα και που είναι θαρρυντικό. Η κυρία Σίμερ είναι εδώ. Έχει πολύ έργο επιτελέσει στο παρελθόν. Αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω όμως είναι τούτο. Εσείς λέτε ότι αν και όταν εμπλακεί με συναπόφαση η Ευρωβουλή, θα μπορούσε να αλλάξει αυτή η ισορροπία πραγμάτων των 75 δις επιπλέον έναντι των 5 δις για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Θα υπήρχε η εξουσία από πλευράς μας να βρούμε ως Ευρωβουλή οι υποστηρικτικά κονδύλια, κονδύλια αρρωγής που θα δίναμε και μάλιστα με, θα έλεγα αρνητικά επιτόκια σε σχέση με τις ε, εταιρείε που εποφελούνται οι σε σχέση με μικρότερα επιτόκια από ότι αυτά τα οποία ισχύουν στην αγορά θα έλεγα ότι όλα αυτά τα χρήματα τα οποία δίνουμε στην ευρωπαϊκή, στην δυτική οικονομία, ο λόγος ε, και ο ρόλος ε, του πληθωρισμού σε ε, λίγα χρόνια θα είναι ανησυχητικός. Θα έπρεπε λοιπόν εδώ να πούμε σε σχέση με την, τα υψηλά επιτόκια και σε σχέση με υψηλό ποσοστό πληθωρισμού δεν θα έπρεπε όμως αυτό να είναι επιζήμιο έναντι των αναπτυσσόμενων κρατών αν θα μπορούσαμε να είχαμε τα ελεγχόμενα επιτόκια για αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο, τον λόγο θα λάβει ο κύριος Μπέρμαν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο και ευχαριστώ για την σύντομη αυτή αλλά σαφή εισαγωγή που κάνατε. Μία ερώτηση θα είχα. Εγώ πιστεύω ότι περισσότερο από ποτεδήποτε είναι αναγκαίο η πρόσβαση των αναπτυσσόμενων χωρών να βελτιωθεί, διότι η οικονομική κρίση δεν διευκολύνει τα πράγματα, ιδιαίτερα όσον αφορά τις χώρες που έχουν οικονομικές δυσκολίες. Όσο πιο ευάλωτες είναι αυτές οι χώρες, τόσο πιο δύσκολο είναι για αυτές να έχουν πρόσβαση σε δάνεια και πιστώσεις και να έχουν και εγγυημένε τέτοιε πιστώσει. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα μπορούσε να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο παράλληλα με την Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και άλλου τέτοιου ε, φορεί. Όσοι έχουν λοιπόν τέτοια, τέτοιες μεγάλες δυσκολίες να έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους χρήμα, παράδειγμα γυναίκες, ε, γεωργοί, ε, άτομα με ειδικές ανάγκες, με αναπηρίες, στρέφονται για να καλύψουν τις ανάγκες τους με τέτοιο χρήμα δεν ε, έχουν πρόσβαση στις τράπεζες ε, και δεν έχουν πρόσβαση σε τέτοιο χρήμα. Αυτό το δείχνουν και μελέτες εξάλλου και νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον της ανάπτυξης να διασφαλίσουμε την πρόσβαση αυτών των ατόμων στα, σε κονδύλια και εκπλήσωμαι και θλίβομαι για το ότι δεν ανέλαβε αυτόν τον ρόλο η Ευρώπη μέχρι σήμερα. Το κατανοώ όταν λέτε ότι θα θέλατε και θα χαιρόσαστε να διευρυνθεί η εντολή σας το πλαίσιο της εντολής σας δεν ήταν ιδιαίτερα φιλόδοξο αυτό το πλαίσιο. Χρηματοδοτούμε υποδομές, σίγουρα χρηματοδοτείτε υποδομές, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό. Όμως οι εγγυήσει αυτών των δανείων και πιστώσεων που δεν επιτρέπεται, δεν πρέπει να είναι τόσο υψηλές και τόσο δαπανηρές. Είναι όμως ένας μοχλός για ιδιωτικά κεφάλαια που δεν επενδύουν ε, τόσο ε, πρόθυμα σε κεφάλαια κινδύνου. Δεν γνωρίζει κανείς για παράδειγμα ποια θα είναι η συγκομιδή σε σχέση με τους γεωργούς ή και για τις γυναίκες έχει κανείς την ως ήθιστε αντιμετώπιση εις βάρος τους ε, και είναι, υπάρχουν προσκόμματα και εμπόδια για αυτές. Ακριβώς σε αυτούς λοιπόν τους τομείς πρέπει να, να δραστηριοποιηθούμε και κατανοώ πολύ καλά τα επόμενα χρόνια με αυτή την πρόκληση που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω της δικής μας για παράδειγμα Κοινοβουλευτικής Επιτροπής αλλά και μέσω της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Προϋπολογισμών πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιωθεί ο ρόλος αυτός. 5 δις ετήσια είναι περισσότερα από ό,τι έχει η Αφρικανική Τράπεζα. Όμως είναι πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με τον τζίρο μας και όσον αφορά το ΑΕΠ που είναι πολύ ανώτερο από πλευράς μας. 5 δις λοιπόν είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, δεν είναι σοβαρό ποσότη. Ή θα μπορούσατε να πείτε για τι δυνατότητε τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων. Ή θα έπρεπε να ήδη να εγκαθιδρυθεί μια νέα τράπεζα, παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης. τραπεζα αναπτυξη πειτε μα ποιε είναι οι απόψει σα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εσείς έχετε τον λόγο. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο κύριος Γκέρενς. Πριν από λίγα χρόνια είχαμε το εξής. Η Παγκόσμια Τράπεζα είχε 15 δις χρέη τα οποία διέγραψε όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες. 15 δις δεν είναι μικρό ποσό και παρόλα αυτά έλαβαν την απόφαση στη συνέχεια να κάνουν κάτι σε σχέση με την ε, Παγκόσμια Τράπεζα σε σχέση με τις ε, χώρες μετόχους ε, να υπάρξει η δυνατότητα να συγκρότησης αυτών των κονδυλίων υπήρχε ένα όρος και προϋπόθεση καλύτερη, χρηστότερη διακυβέρνηση και διαχείριση από πλευρά των κρατών. Αυτή η συμφωνία σε σχέση με την Παγκόσμια Τράπεζα και τις ε, αποδέκτριες χώρες ε, καταλήγει σε ακόμα αυστηρότερους όρους και προϋποθέσεις σήμερα και στη σχέση σας με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Βλέπετε σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ε, να κρύβεται κάτι άλλο ή φαντάζεστε κάτι διαφορετικό από αυτά τα οποία έχει προβλέψει η Παγκόσμια Τράπεζα. Η δεύτερη ερώτησή μου είναι εξή σε σχέση με το, αυτό που θα είσαστε πρόθυμοι να ε, εγκρίνετε για τον ιδιωτικό τομέα. Διαπιστώνει κανείς ότι στην Αφρική κάποιες εμπορικές τράπεζες, τουλάχιστον μερικές από αυτές, έχουν χρήμα επειδή τα κονδύλια τα οποία έχουν στη διάθεσή τους δεν δαπανώνται με σωστό ε, και ε, χρηστό τρόπο. Δεν βλέπετε ακριβώς εκεί μια δυνατότητα να υπάρχει για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η ανάγκη υπάρχει, αλλά θα μπορούν να πληρώνονται, να εξοφλούνται αυτά τα δάνεια. Βλέπετε εκεί κάποια δυνατότητα από πλευρά σας. Και μια άλλη ερώτηση. Θα ήθελα να μου πείτε πώς εσείς βλέπετε αυτά τα πράγματα. Διαπιστώνει κανείς ότι τα δάνεια, οι πιστώσεις που εγκρίνονται για την Αφρική είτε είναι θεσμικού χαρακτήρα μεταξύ εμπορικών τραπεζών για παράδειγμα ή ε, σε σχέση με ε, επίσημους αποδέκτες ε, αναπτυξιακής βοήθειας αλλά και σε σχέση με την μικροοικονομία ε, τα επιτόκια είναι πολύ ψηλά διότι υπάρχει αναχρηματοδότηση μέσω των διεθνών κεφαλαιακών αγορών και υπάρχουν επιτόκια τα οποία είναι διπλάσια ή τριπλάσια εκείνων των ποσοστών επιτοκίων που ισχύουν για τις ε, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ε, που λαμβάνουν τέτοια δάνεια. Και τι διαπιστώνει μετά στη, κανείς στη συνέχεια. Ότι και αυτά τα ποσοστά δεν, δεν παρακολύουν την αποπληρωμή. Το αντίθετο, για τα μη μικροδάνεια χαρακτηριστικό είναι ότι τα δάνεια αυτά σε πάνω από 90% αποπληρώνονται. Αυτό είναι αξιοπρόσεκτο, είναι αξιόλογο. Αν νομίζει κανείς ότι ε, χάνονται αυτά, δεν συμβαίνει αυτό στα μικροδάνεια. Γι' αυτό ερώτησή μου, τι σκοπεύετε να κάνετε και ποια επιτόκια θα υιοθετήσετε στην προσπάθεια αυτή και σε, ποιες, σε ποιους οίκους αξιολόγησης θα στραφείτε ώστε η φερεγγιότητα, η αξιολόγηση αυτών των αποδεκτών να μπορέσει να αξιολογηθεί, να αποτιμηθεί αντικειμενικά. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Ευχαριστώ. Merci, Madame la euh, Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντέβα έθεσε εξ αρχής μια σημαντική ερώτηση. Ποιες οι δυνατότητες να αντιμετωπίσουμε την σημερινή κατάσταση και μέσα από τη συζήτηση που θα οργανωθεί και το 2010 μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου και έθεσε τον τύπο, το δάκρυο τον τύπο των ύλων, δηλαδή την, ε, τον περιορισμό που μας θέτει ο προπολογισμό. Γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο να αυξήσουμε συνολικά τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Τώρα για ένα προπολογισμό που είναι το 1% του ΕΠ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, μια, μια οποιαδήποτε αύξηση δεν θα είναι σημαντική μένα, αλλά ξέρουμε ποια είναι και πολιτική πραγματικότητα. Είναι δύσκολο στην πράξη να έχουμε αύξηση του ευρωπαϊκού προπολογισμού και ιδίω για το σταθερό μα ε, χαρτοφυλάκιο, πώ θα προκύπτει τον προπολογισμό. Τώρα, εάν θέλουμε να κάνει περισσότερη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μπορούμε να διακρίνουμε μεταξύ δύο περιπτώσεων. Το τι κάνουμε βάσει εντολή. Οι εντολέ, όπω είπαμε, συνοδεύονται από μέσα που δίδει ο Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Όταν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο αποφασίσουν για την εξωτερική εντολή τη ΕΤΕ, θα αποφασίσουν ταυτόχρονα και ποια υπερκοδότηση των εντολών αυτών. Δηλαδή ότι ο ευρωπαϊκός προπολογισμός καλύπτει το πολιτικό κόστος, τον πολιτικό κίνδυνο που θα αναλάβετε. Αυτό λοιπόν θα έχει ένα συγκεκριμένο κόστος για τον προπολογισμό. Αλλά ένα κόστος που δεν θα είναι και τεράστιο. Ε, έχω μάλιστα την τάση να πω ότι θα είναι και πτωτική η πορεία του. Διότι επειδή δεν κάνουμε και τόσο πολύ έκκληση στην εγγύηση αυτή του ευρωπαϊκού προπολογισμού, στη διασφάλιση του προπολογισμού, αυτή τη στιγμή ίσως έχουμε και πολύ μεγάλο απόθεμα. Εάν λοιπόν αυξήσουμε το χαρτοφυλάκιο των εντολών, θα πρέπει να ξαναδούμε και τη μέθοδο υπολογισμού για την διασφάλιση που μας δίνει ο προπολογισμό. πέραν της εντολής αυτής καθεαυτής υπάρχει δυνατότητα να αποφασίσουμε και να δημιουργήσουμε διευκολύνσεις χρηματοδότησης. Αλλά με ανάληψη του κινδύνου από εμά του ίδιου. Χωρί λοιπόν διασφάλιση από τον, Ευρωπαϊκό, από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Μπορούμε να το κάνουμε, αλλά γι' αυτό πρέπει να έχουμε την ομόφωνη γνώμη των ε, κρατών μελών, όλων των κρατών μελών, βάσει του άρθρου 18 του καθεστώτο του καταστατικού τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Μπορούμε λοιπόν, εφόσον λάβουν ομόφανη απόφαση τα κάτι μέλη τη Ευρωπαϊκή ε, Ένωση, να περάσουμε σε τέτοιε εξωτερικέ δράσει. Υπάρχουν κάποια παραδείγματα, να σα δώσω τέσσερα πρόσφατα. Τα κράτη-μέλη συμφώνησαν ότι μπορούμε να διευκολύνουμε τη χρηματοδότηση προγραμμάτων σε στον ενεργειακό τομέα, εφόσον είναι προγράμματα που θα συνεισέφεραν στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών ή την ασφάλεια της προμήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το χαρτοφυλάκιο αυτό έφτασε τα 3 δις για την ε, περίοδο 2007-2013. 3 δις λοιπόν διαθέσιμη χρηματοδότηση για τα οποία δεν έχουμε τη διασφάλιση από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε οποιοδήποτε πρόγραμμα. Θα πρέπει να είναι προγράμματα τα οποία θα έχουν συγκεκριμένο investment grade, συγκεκριμένο βαθμό επενδυτικό, αλλά ε, έχουμε ένα περιθώριο χρηματοδότηση. Εδώ ένα άλλο παράδειγμα είναι αυτό που ονομάζουμε pre-exception facility, δηλαδή διευκόλυνση προένταξης. Ε, 7,5 δις ευρώ για την περίοδο 2007-2013 ε, συμπλήρωμα στη βοήθεια για τις, για τις χώρες, ε, τις προενταξιακές, τις γείτονες χώρες τις οποίες μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε με ίδιο κίνδυνο χωρίς την συνδρομή του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού. Άλλο παράδειγμα, η διευκόλυνση για την ε, Μεσόγειο. Σε δύο περιπτώσεις τα κάτι μέλη δέχτηκαν να δώσουμε από δύο φορές ένα δις, ένα χαρτοφυλάκιο δανείου ενός δις για τα προγράμματα που μπορούσαν να υλοποιηθούν στη Μεσόγειο με ανάληψη του κινδύνου από εμάς τους ίδιους. Και ένα άλλο, ακόμη πιο πρόσφατο παράδειγμα που δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, αλλά είναι πρόταση που κάναμε προς τα κάτι μέλη, είναι να δημιουργήσουμε μια διευκόλυνση παρόμοια για τους εταίρους μας προς για ένα ποσό 2,5 δις. Για 1,5 δις. Αυτό λοιπόν ε, είναι το ποσό που προβλέψαμε με ένα χαρτοφυλάκιο πολύ περιορισμένο και με τις εγγύησεις που διαθέτουμε και βεβαίως εφόσον μας δοθεί η έγκριση για να κάνουμε περισσότερα αλλά με ανάληψη του κινδύνου από εμά. Και μια άλλη πτυχή, η οποία δεν έχει σχέση με τον προπολογισμό. Ο συσχετισμός που πρέπει να γίνει κατά την άποψή μου μεταξύ των δυνατοτήτων δανειοδότησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των επιχορηγήσεων που μπορεί να προέρχονται είτε από τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση είτε των κρατών των ίδιων. Διότι επαναλαμβάνω ότι είναι δύσκολο στι αναπτυσσόμενε χώρε να χρηματοδοτήσουμε οποιαδήποτε, οποιοδήποτε σχέδιο με τα επιτόκια τη αγορά. Υπάρχουν προγράμματα που είναι κερδοφόρα, οπότε αυτά μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα επιτόκια τη αγορά, αλλά αυτό δεν μπορεί να ισχύει για όλα τα προγράμματα, ιδίω αυτά που έχουν κοινωνικέ διαστάσει. Έχουμε λοιπόν ανάγκη να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε με παραχωρητικά επιτόκια, αλλά για αυτό το σκοπό χρειαζόμαστε επιχορηγήσει. Οπότε αυτό θα έχει αντίκτυπο στον προπολογισμό. Πρέπει λοιπόν να το συζητήσετε. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου των Επενδύσεων και σε συνδυασμό με την Επιτροπή και τα κρατη λόγω χάρη, προβλέψαμε ένα trust fund για τη χρηματοδότηση των υποδομών ε, στις περιφέρειες της Αφρικής. Υποδομές οι οποίες αφορούν πολλές χώρες της Αφρικής ταυτόχρονα και εκεί συνδυάζουμε δάνεια της ΕΤΕ μαζί με επιχορηγήσεις που προέρχονται από το Trust Fund. Το Trust Fund το οποίο τροφοδοτείται από αυτό το ίδιο από τη μια από το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο και από την άλλη από τι οικειοθελεί συνεισφορέ των κρατών μελών. Πρόκειται λοιπόν για μια φόρμουλα πρόσφατη, αλλά η οποία έχει δώσει πολύ καλά αποτελέσματα, διότι εδώ είμαστε πλέον σε θέση να συνδυάσουμε τι δικέ μα χρηματοδοτήσει και την τεχνική μα εμπειρογνωμοσύνη, όπω έλεγα προηγουμένω, ιδίω για τα προγράμματα μεταφορών και ενέργεια, με τι επιχορηγήσει που επιτρέπουν να φτάσουμε σε επιτόκια παραχωρητικά ουσιαστικά. Να κάποιες δυνατότητες λοιπόν οι οποίες είναι υπαρκτές και εντός των φραγμών του προπολογισμού που όλοι γνωρίζουμε. Τώρα για την ερώτηση του κυρίου Μπέρμαν, την πρόσβαση στις πιστώσεις και ιδίως τη διασφάλιση, τις εγγυήσεις. Ταυτόχρονα θα απαντήσω λίγο πολύ και στον κύριο Γκέρνης για τα μικροοικονομικά. Έχουμε εδώ ένα καλό παράδειγμα, διότι παράσχαμε εγγύηση σε τοπικούς τραπεζικούς οργανισμούς που χρηματοδοτούν ακριβώς φορείς μικροοικονομικών. Είναι δυνατό και νόμιμο και εγώ ίδιος επισκέφθηκα μια τέτοια ε, συνάντηση στην, στην ΤΑΚΑ που υπήρχε συνάντηση σε επίπεδο γειτονιάς των ε, φορέων των υπευθύνων και μιλούσαμε εδώ για ποσά ε, που διαχειρίζονταν οι ίδιοι οι Σενεγαλέζοι και χρηματοδοτήσαμε και την Τράπεζα τη Σενεγάλη, αλλά ο κίνδυνο που αναλαμβάναμε ήταν ε, περιορισμένο. Διότι το ποσοστό επιστροφή των ε, δανείων είναι πολύ ψηλό. Επίσης με 50 εκατομμύρια δολάρια συμμετάσχαμε στην διευκόλυνση Microfinance Enhancement Facility, στην ενίσχυση, στη διευκόλυνση ενίσχυσης των οικοπιστώσεων και εδώ Προσφέραμε στήριξη σε φορεί μικροπιστώσεων, οι οποίοι λειτουργούν καλά, αλλά σε, στη φάση αυτή τη κρίση ε, δεν έχουν δυνατότητα να αναχρηματοδοτηθούν. Εδώ λοιπόν χρηματοδοτήσαμε υγιεί φορεί μικροπιστώσεων στην Αφρική. Δεν είναι πανάκια βεβαίω οι μικροπιστώσει, όμω είναι ένα τρόπο να στηρίξουμε την ανάπτυξη αυτού του είδου τη δραστηριότητα. Τώρα, μα ρωτήσατε κύριε Γκέρνη και για τι προποθέσει που θέτουμε. Πολλέ φορέ συμμετέχουμε σε δράσει συγχρηματοδότηση με άλλου οργανισμού, την Διεθνή Τράπεζα, την Αφρικανική Τράπεζα Επενδύσεων και άλλου. Οπότε πρέπει να συμφωνήσουμε και για κοινέ προποθέσει που θα εφαρμόσουμε για τα διάφορα προγράμματα. Θα έλεγα ότι η ΕΤΕ από παράδοση εφαρμόζει προποθέσει που έχουν άμεση σχέση με τη φύση του ίδιου του προγράμματο. Προποθέσει λοιπόν που μα φαίνονται αναγκαίε προκειμένου να διασφαλίσουμε την επιτυχία του προγράμματο δεν θέτουμε τι εξαρχικέ εξαρχή προποθέσει μακροοικονομικού χαρακτήρα. Αυτή ίσω είναι η διαφορετική μα προσέγγιση σε σχέση με την ε, Παγκόσμια Τράπεζα. Οι δικέ μα προποθέσει αφορούν και στοχεύουν κυρίω στην επιτυχία του προγράμματο, που μπορεί να αφορούν και τομεακέ ή μακροοικονομικέ βέβαια διαστάσει, όμω πάντοτε έχοντα υπόψη το τι χαρακτήρα, τι φύση έχει το πρόγραμμα που χρηματοδοτούμε. Τέλο, αναφερθήκατε στο αρκετά ευρύ πρόβλημα των Αφρικανικών τραπεζών, που όπως είπατε έχουν θέμα ρευστότητας και που πολλές φορές χρησιμεύουν για να τροφοδοτήσουν την τοπική οικονομία. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι οι τράπεζες αυτές δεν είναι καλά εξοπλισμένες για να αναλύσουν τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν. Δηλαδή, τίνουν να δανείζουν χωρίς να έχουν επαρκή δυνατότητα ανάλωσης και διαχείρισης του κινδύνου. Πιστεύουμε λοιπόν ότι μια από τις δικές μας συμβολές, τις πιθανές συμβολές μας εδώ, είναι όχι μόνο να χρηματοδοτούμε, αλλά και να προσφέρουμε τεχνική στήριξη για την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης του κινδύνου στις Αφρικανικές τράπεζες. Σας ευχαριστώ. Έχω ακόμη έξι εγγεγραμμένους στον κατάλογο των αγορητών. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ολοκληρώσει μέχρι τις 4 και 10. Διότι ο επόμενο προσκεκλημένο μα έχει μόνο 30 λεπτά, ο κύριο Διούφ. Λοιπόν, σα ζητώ να θέσετε τι ερωτήσει σα σε ένα λεπτό ο καθένα. Το, λόγο έχει ο κύριο Γκερέρο Σαλόμ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, μάλλον. Ευχαριστώ, κύριε ε, ε, Δίκητα. Στην ε, παρουσίαση που κάνατε, μας δώσετε ορισμένες πληροφορίε και αναγνωρίζουμε την αξία του έργου σας. Επίσης κηρύξατε τον πόλεμο στους φορολογικούς παραδείσους. Παρόλο που γνωρίζουμε ότι δεν κηρύξατε τον πόλεμο σε όλους τους φορολογικούς παραδείσους, ορισμένοι διαφεύγουν ακόμη. Αυτά <clears throat> δεν είχε αρχίσει ακόμα η οικονομική κρίση το 2007. Ούτε είχαμε λοιπόν την κρίση, ούτε είχαμε τις ε, διαθώσεις και τις δομές που έχουμε σήμερα. Αυτά τα πράγματα έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Εάν μπορείτε τώρα να βοηθήσετε ώστε η τράπεζα να αποκτήσει ένα νέο πλαίσιο αρμοδιότητων, να ε, έχει στη διαθεσή και περισσότερα χρήματα, αυτό θα ήταν καλό. Και ε, στη βάση θα είναι και, βάση μιας καλύτερης εξωτερικής πολιτικής ανάπτυξης. Ευχαριστώ κύριε Κέλλερ. Τρεις ερωτήσεις. Πρώτα, μιλήσατε για Κοπενχάγη και αλλαγή του κλίματος. Διάβασα ότι στα τελευταία, στα τελευταία 7 χρόνια έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 6,5 δισεκατομμύρια σε μία ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μόνο τα μισά περίπου σε ανανεώσιμες. Γιατί? Γιατί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δίνει τόσο μεγαλύτερη έμφαση σε μία ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ε, χρηματοδότηση και την ενίσχυσή τους δηλαδή. Τώρα για τους ε, διαμεσολαβητές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και εκτός Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή φαίνεται να υπάρχει ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά τι πληροφορίε για το πώ δαπανώνται τα χρήματα μετά. Υπάρχει δηλαδή κάποια έλλειψη διαφάνεια. Διερωτώ με εάν θα αυξήσετε την διαφάνεια για το πώ χρησιμοποιούνται τα χρήματα αυτά από του ε, διαμεσολαβητές αυτούς. Και τρίτη ερώτηση για του φορολογικού παραδείσους. Κατανόησα από αυτά που είπατε ότι υπήρχε πρόβλημα στο παρελθόν, αλλά ότι καταβάλλετε προσπάθειες για να βελτιώσετε την κατάσταση. Πώς γίνεται αυτό. Μέσω των έργων που χρηματοδοτείτε θα υπάρχουν και φορολογικά έσοδα. Και εν πάση περιπτώσει τα όσα γίνονται ήδη θεωρείτε ότι είναι επαρκή. Αρκούμε σε αυτά. Χωρίς μικρόφωνο Thank you, Madam Ο κύριο Κάσμαν. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομο. Ο κύριο Μέιστατ Καλύψει ήδη ορισμένε από τι ερωτήσει που ε, ε, ε να ε, θέσω. Οι επενδύσεις δεν έχουν σχέση μόνο με την κεφαλιακή απόδοση, αλλά και τις μακροχρόνιες αποδόσεις και τη σταθερότητα και την ανάπτυξη. Και είμαι βέβαιος ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συμφωνεί με τους στόχους αυτούς και είμαι βέβαιος ακόμη ότι δίνονται προτιμησιακά επιτόκια σε ορισμένους ε, οφειλέτες μόνο. Και αυτό έχει σχέση με τα έργα ε, στα οποία προσφέρεται χρηματοδότηση. Οι Κινέζοι, για παράδειγμα, δεν έχουν απολύτως κανένα δισταγμό να δανείζουν μεγάλα ποσά χρημάτων και το μακροχρόνιο αποτέλεσμα Ελπίζω ότι δεν θα το αγνοήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ε, ιδίω αυτή, και, αλλά και οι χώρε μέλη. Τώρα για το soft power, την ήπια δύναμη. Έχουμε, εκτός από ήπια δύναμη, έχουμε και νόμους και συνθήκες. Και οι συνθήκες προβλέπουν και κυρώσεις. Και έχουμε και την καινούργια ε, συνθήκη. Γεια σας κύριε Ντέβα. Και τελευταία μου ερώτηση που μου την έδωσε ο κύριος Μπέρμαν. Μπορεί να παίξει ρόλο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στον χώρο των ασφαλιών, δηλαδή για χώρες ή επιχειρήσεις ή και άτομα που θέλουν να μπουν στην, ε, να ασφαλίσουν για παράδειγμα τις οδιές τους ή κάποιες υπηρεσίες που προσφέρουν. Βλέπω κινήσεις της κεφαλής που σημαίνει ότι ίσως δεν πρόκειται να μου δώσετε κανένα απάντηση αλλά σας ενθαρρύνω πάντως σε όσα πράτετε και ορισμένοι από εμά αναγνωρίζουμε ότι έχει και ποικιλία η χρηματοδότησή σας και ότι χρηματοδοτείται ίσω και έργα τα οποία ίσως να μην είναι βραχυπρόθεσμα βιώσιμα, αλλά σίγουρα είναι, αφού όσον αφορά την ανάπτυξη, βιώσιμα πιο μακροχρόνια. Κύριε Τσίμερ, Ευχαριστώ κύριε Μάιστατ που πάλι εδώ ήρθατε στην Επιτροπή μας στην αρχή της κοινοβουλευτικής θητείας για να συζητήσετε μαζί μας το έργο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Με ενδιαφέρει κυρίως κατά πόσον υπάρχουν αποδείξιμες εξελίξεις, δηλαδή εξελίξεις μετρήσιμες από την τελευταία φορά που βρεθήκατε εδώ κοντά μας και ε, πώς αξιολογείτε εσείς οι ίδιοι το έργο σας, κατά πόσον πετύχατε να εντάξετε και τους επιτόπου εταίρους από την αρχή, από τις πρώτες φάσεις των έργων περισσότερο, αλλά επίσης ποιες είναι οι αξιολογήσεις των ε, συνεπειών, των επιπτώσεων των ε, χορηγωμένων δανείων, επίσης σε κοινωνικά θέματα, στα δικαιώματα των γυναικών, στην ε, απασχόληση κλπ. Δηλαδή κατά πόσον επετεύχθησαν αυτά τα πράγματα να επεκταθούν, κατά πόσον μπορέσατε να ενισχύσετε και τις δομές της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κατά πόσον εκτιμάται ότι είναι, όπως εκτιμούν ορισμένοι, ε, είναι ασθενής ακόμα η ΕΤ σε ορισμένες ε, περιφέρειες. Επίσης με ενδιαφέρει ποιες προσδοκίες θέτετε εσείς ο ίδιος απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μας ιδιότερα, ιδιαίτερα, γνωρίζοντας κιόλας ότι με την νέα συνθήκη θα συμμετέχει πολύ περισσότερο το κοινοβούλιο στη λήψη των αποφάσεων. Σε ποιου τομεί θεωρείτε ότι θα μπορούσαμε να συμμετέχουμε περισσότερο. Για παράδειγμα και για την ε, κάλυψη θέσεων του οργανογράμματος και ούτω καθεξής. Εκεί δηλαδή όπου εμείς έχουμε κάποιες προσδοκίες από μια συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά και εσείς σίγουρα κάποια πράγματα μένετε από εμά. Θα ήταν καλό αν μπορέσετε να τοποθετηθείτε και σε αυτά. Και μια τελευταία παρατήρηση που αφορμή μου δίνει ο κ. Κάσμαν για αυτήν, η αναφορά του δηλαδή στην δράση της Κίνας και την διάθεσή της να διαθέσει σημαντικές και μεγάλες πιστώσεις και πολύ γρήγορα. Πρόσφατα νομίζω παραπονεθήκατε, εκφράσατε το παράπονο δηλαδή, ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με τα ίδια κριτήρια όπως οι Κινέζοι. και είχε το νόημα αυτό ότι ίσως θέματα ε, διατήρησης απασχόλησης να μην χρειάζεται να παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο. Ή εξακολουθείτε να θεωρείτε το ίδιο πράγμα ή θεωρείτε ότι ανεξαρτήτως του πώς δρούν οι Κινέζοι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τηρεί και να σέβεται και να προωθεί τις αξίες αυτές. Η κυρία Τεκέιζερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ο κύριος και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορούν να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο σίγουρα στο έργο τους και αυτό θα μου έδινε ιδιαίτερη ικανοποίηση και εμένα τις ίδιες. Τώρα για την απόφαση του Συμβουλίου που αναφέρατε για δανειοδότηση σε περιπτώσεις της, σε χώρες της Μεσογείου. Εδώ μιλήσατε για δάνεια και ήθελα μια επιβεβαίωση. Δάνεια προς το Ισραήλ ήταν αυτά. Το άκουσα αλλά δεν είχα καμία επιβεβαίωση. Και αν αυτό ισχύει τι, για ποσά μιλάμε και πότε ε, εγκρίθηκαν αυτά τα δάνεια. Και για να κλείσουμε να θέσω κι εγώ μια ερώτηση από μένα την ίδια. Μας μιλήσατε για το τραπεζικό εισόδημα, το καθαρό εισόδημα της ΕΤΕ κατά μέσο όρο τα τελευταία πέντε χρόνια. Από τη μια και από την άλλη, επειδή εργάζεστε και βάσει των μαύρων καταλόγων του ΩΣΑ και μετά την συνάντηση τη Σύνοδο του G20 γνωρίζουμε ότι εδώ ε, αυτό δεν υποχρεώνει τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεστε να απαλλαγούν από αυτές τις ε, φορολογικές ελαφρύνσεις από τις οποίες αποφελούνται. Θα εξετάζει λοιπόν πλέον η ΕΤΕ το κατά πόσο οι επιχειρήσεις αυτές ε, σε, αν περιλαμβάνονται στους μαύρους καταλόγους και θα δείτε αν ωφελούνται από εξαιρετικές φορολογικές ελαφρύνσεις οι επιχειρήσεις που χρηματοδοτείτε και θα, θα ζητάτε από τις εταιρείε αυτές να τα, κινηθούν λόγω χάρη όχι από τη, Ζάμπια στον Άγιο Μαυρίκιο. Πρόεδρε, κατάλαβα απολύτως το πνεύμα σας. Θα απαντήσω λοιπόν και εγώ τηλεγραφικά θα με συγχωρήσουν τα μέλη της Επιτροπής, αλλά θα παραμένουμε στη διάθεσή τους για να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες προσεχώς, εάν το επιθυμείτε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Γκερέρο Σαλόμ για τη στήριξή του. Στην κυρία Κέλλερ, σύντομα. Να πω ότι ο κανόνα που έχουμε ορίσει για τον εαυτό μα και ενέκρινε και το Διοικητικό μα Συμβούλιο είναι ότι τουλάχιστον 20% των νέων δυνατοτήτων παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματο που χρηματοδοτούμε 20% θα πρέπει να ε, απευθύνεται στι ανανεώσιμε ε, πηγέ ενέργεια. Και αυτό το σεβαστήκαμε την τελευταία δεκαετία και είμαι έτοιμο να σα δώσω και αριθμητικά στοιχεία. 20% λοιπόν τουλάχιστον βάσει ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Για την διαφάνεια στήριξη μεσαίων επιχειρήσεων. Οι νέε συμβάσει που προσφέρουμε από το 2008 διασφαλίζουν αυτή τη διαφάνεια πολύ καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Εφόσον στι νέε συμβάσει. Υπάρχει γραπτή ρητή δέσμευση της ενδιάμεσης ε, τράπεζας για τα ελάχιστα πλεονεκτήματα που πρόκειται να μεταφέρει στην μικρή δικαιούχο επιχείρηση είτε ως προς τα επιτόκια είτε ως προς την οριμότητα του δανείου και έπειτα υπάρχει η δέσμευση της ενδιάμεσης τράπεζας να πληροφορεί ε, ξεχωριστά κάθε μικρή επιχείρηση για το πλεονέκτημα που θα αποσπά χάρη στην παρέμβαση της ΕΤΕ. Αυτό υπό διάφορες μορφές. Μια αγγλική τράπεζα δίνει επιταγή λόγω χάρη στη μικρή επιχείρηση και αυτό είναι το οικονομικό της ωφέλιμα που παίρνει από την παρέμβαση της ΕΤΕ. Μια γαλλική τράπεζα στέλνει επιστολή στον καθένα από τους δικαιούχους. Σε κάθε περίπτωση απαιτούμε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια για την μεταβίβαση των πληροφορημάτων. Και έπειτα για τις συμβάσεις τις καινούριε προβλέπεται η δυνατότητα της ΕΤΕ να οργανώσει έλεγχο για την διάμεση τράπεζα για να είμαστε βέβαιοι ότι οι προποθέσεις αυτές γίνονται σεβαστές. Σε ό,τι αφορά τώρα τους φορολογικούς παραδείσους. Σας είπα ότι αναθεωρήσαμε την πολιτική μας βάση των αποφάσεων του G20 και θα έλεγα ότι ως προς αυτό έχουμε προλάβει και τις υπόλοιπους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Είμαστε στην πρωτοπορία. Ίσως πήγαμε πολύ μακριά ζητώντας την ε, μετακίνηση σε άλλη δικαιοδοσία πριν ε, εγκρίνουμε δάνειο. Αληθεύει, Πρόεδρε, ότι παραμένουμε πιστοί στους καταλόγους του οσα δεν τους ε, ορίζουμε εμείς τους καταλόγους των φορολογικών παραδείσων. Ίσως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να αναλάβει την πρωτοβουλία να συντάξει τέτοιους καταλόγους ώστε να είναι πληρέστεροι από τη σημερινή κατάλογη του ΩΣΑ. Σημείωσα πάντως τις παρατηρήσεις του κυρίου Κάσμαν και νομίζω ότι έχει δίκιο να τονίζει ότι θα πρέπει να είμαστε διερωτικοί στη θέση των στόχων μας. Για τις ε, ασφάλειες, αυτό είναι εκτός του καταστατικού μας. Δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε λοιπόν δράσεις ασφάλισης και όπως και η ατζίμερ ε, έθεσε ερώτηση για, τις, τα δάνεια από τις κινέζικες τράπεζες. Είναι ένα φαινόμενο που αυξάνεται συνεχώς, ε, παίρνει αυξητικές διαστάσεις στην Αφρική σε περιπτώσεις όπου επί χρόνια δεν ειδωτούσαμε συγκεκριμένους δικαιούχους, την τελευταία στιγμή μας αντικαθιστά. Μας αντικαθιστά μια κινέζικη τράπεζα που θέτει πολύ λιγότερες προποθέσει τελικά. Βέβαια, πέραν αυτού, συνεχίζω να πιστεύω ότι εάν θέλουμε να φέρουμε πέρα στην αποστολή μας, πρέπει να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε να απαιτούμε το σεβασμό συγκεκριμένων προποθέσεων και κοινωνικών και περιβαλλοντικών. Ιδάλλως, δεν θα είμαστε σοβαρή τράπεζα. Είμαστε τράπεζα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να προσπιζόμαστε τι ευρωπαϊκέ αξίε. Είμαι λοιπόν υπέρ τη διατήρηση των προποθέσεων αυτών. Ε, σε ό,τι αφορά ιδίω το σεβασμό των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προδιαγραφών. Ακόμη και αν οι συνέπειε σε κάποιε περιπτώσει είναι ότι οι κυβερνήσει προτιμούν να συνάψουν σχέσει οικονομικέ και συναλλαγέ με κοινωνικέ τράπεζε. Ένα παράδειγμα από τις πρόσφατες συζητήσει μας όπου επιτελέσαμε πρόοδο ήταν αυτό που αφορά την ανάλυση προγραμμάτων για τον αντίκτυπο, περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Αναπτύξαμε μια νέα μεθοδολογία το οποίο ονομάζουμε περιβαλλοντικό και κοινωνικό ε, πλαίσιο μελετών επιπτώσεων αυτό θα μας διασφαλίσει για τις μελλοντικέ μας πολιτικές να έχουμε μια πληρέστερη μελέτη και πιο διεξοδική ανάλυση. Βεβαίω υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμη για να ολοκληρωμένο το πλαίσιο αυτό, αλλά αυτό μας παραπέμπει και σε παρελθούσες συζητήσει μας για τέτοιου είδους προγράμματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το προσωπικό, είναι σαφέ ότι για να γίνει σωστά η δουλειά μα χρηματοδότηση δηλαδή προγραμμάτων σε αναπτυσσόμενε χώρε, πρέπει να έχουμε πολύ περισσότερο ε, άτομα. Για να σα δώσω μια ιδέα για τι σημερινέ μα διαστάσει. Είπα ότι δανείζουμε 75 δι ευρώ φέτο, 5 ε, μόνον εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Λιγότερο από το 10% λοιπόν. Όμω, ω προ το προσωπικό μα, η αναλογία, και θα μιλήσω τώρα για το προσωπικό που ε, ασχολείται με αυτά τα προγράμματα, είναι, η αναλογία είναι 2 τρίτα, 1 τρίτο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αναλογικά ήδη προσλαμβάνουμε πολύ περισσότερα άτομα για τι επιχειρήσει εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση από ότι εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντω αυτό δεν αρκεί. Είμαι ο πρώτο που αναγνωρίζω ότι ιδιαίτερω ε, δυσκολευόμαστε σε κάποιου τομεί, κυρίω στον τομέα τη παρακολούθηση. Σα είπα ότι έχουμε επιτελέσει πραγματική πρόοδο στην, ε, των προτέρων ανάλυση των προγραμμάτων, όμω απομένουν πολλά βήματα πρόοδου να γίνουν στην παρακολούθηση, στο monitoring, για να ε, παληθεύουμε το κατά πόσο έγιναν σεβαστέ οι προποθέσει που θέσαμε. Ένα από τα μέσα που διαθέτουμε είναι προφανώ να έχουμε εξωτερικά, εξωτερικούς συνεργάτες εξωτερικά γραφεία. Έχουμε πλέον σήμερα κάποια τέτοια γραφεία και έχουμε σκοπό να συνεχίσουμε στα πλαίσια βεβαίω των προπολογισμών που οι μέτοχοί μα θα μα παραχωρήσουν. Αλλά έχουμε σκοπό να προβλέψουμε τη δημιουργία και άλλων τέτοιων εξωτερικών γραφείων. Τέλο, και αν μου το επιτρέπετε, Πρόεδρε, ένα τελευταίο λεπτάκι στον αντιπρόεδρο μου που βρίσκεται στην αίθουσα και είναι πιο καλός γνώστης των θεμάτων της Μεσογείου να του δώσω το λόγο για να σας απαντήσει για την Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να πω ότι για τη Μεσόγειο δανείζουμε περίπου 1,5 δις ευρώ ετησίως και από αυτό το 1,5 δις ευρώ το ετήσιο που μα κάνει τον πρώτο χρηματοδότη αυτή τη περιοχή. Λιγότερα από τα 200 δι πηγαίνουν στο Ισραήλ και 200 εκατομμύρια πηγαίνουν στο Ισραήλ και αυτό θα αφορά και τις δύο επόμενες ε, δράσεις μας, κοινέ δράσεις Ισραηλινο-Παλαιστινιακές για τον τομέα του, της ηλεκτρικής ενέργειας και του capital risk. Διότι οι ομάδες και από τις δύο πλευρές συνεργάζονται μαζί μας, και των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών. Και την τελευταία σας ερώτηση, Πρόεδρε, την οποία δεν απάντησα, για το ετήσιο κέρδος μας, περίπου 1,5 δι, δις, και εδώ υπολογίζουμε να έχουμε, ότι πρέπει να έχουμε κέρδος για, δύο λόγους. Πρώτον, διότι πρέπει τακτικά να αυξάνουμε το κεφάλαιό μα. Το καταστατικό μα λέγεται ότι το σύνολο των τρεχών των δανείων μα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 250% του κεφαλαίου μα. Οπότε, όταν αυξάνουμε τι δράσει μα, πρέπει, όταν θέλουμε να κάνουμε περισσότερα για να ανοιχτήσουμε την κρίση, πρέπει να αυξήσουμε και το όριο. Πρέπει να ζητήσουμε από του μετόχου μα, τα κράτη-μέλη, αύξηση του κεφαλαίου και η απάντηση, η τυπική απάντηση είναι να μα λένε εντάξει, αλλά δεν πρέπει να μα κοστίσει τίποτα. Δεν πρέπει να επιβαρύνει αυτό τον προπολογισμό των κατομελών. Ήμουν στη συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών και μα είπαν στην ΕΤΕ μπορείτε να αυξήσετε βεβαίω τον προπολογισμό τη ΕΤΕ, αλλά δεν θέλουμε να κοστίσει ούτε ένα φράγκο. Λέγαμε κάποτε, τώρα πια λέμε ούτε ένα ευρώ. Στον προπολογισμό των 100 μιλάμε λοιπόν για αποθεματικά τα οποία μπορεί να είναι ανεπαρκή, αλλά πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι θα διασφαλίσουμε την μελλοντική αύξηση των ε, δράσεών μα. Και βεβαίω αυτό σημαίνει ότι και τα κράτη-μέλη μπορούν να αναλάβουν μεγαλύτερο κίνδυνο για να χρηματοδοτήσουν ή να συγχρηματοδοτήσουν προγράμματα, όπω τώρα δεν χρηματοδοτούσαν χωρί τη δική μας την παρέμβαση. Αλλά εδώ πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένε προμήθειε. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε συγκεκριμένο εισόδημα ετησίω για να μπορέσουμε να καλύψουμε και τι προμήθειε. Αυτό λοιπόν ήδη συμβαίνει έχουμε ένα εισόδημα περίπου 1,5 δις ευρώ. σε τη φορά το τελευταίο τελευταίο σας ερώτημα, ας σκεφτούμε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Σε ορισμένε υποθέσει ε, με τις οποίες ασχολήθηκα δεν είχαμε την εντύπωση ότι η χρηματοδότηση από την ΕΤΕ μείωσε τους ή επηρέασε τους πόρους ε, του κράτους ε, που υλοποιείται το πρόγραμμα. Για, να, για τις επενδύσεις ενός προγράμματος Κάποια αφρικανικά κράτη προβλέπουν σημαντικές ε, φοροαπαλλαγές. Ε, δικαίως ή αδίκως, αλλά αυτό είναι δικαίωμα του αυτοκυριαρχού κράτους. Κάποιες φορές είναι πολύ γενναιόδοροι. Πρέπει να το παραδεχτούμε, αλλά κάποιες φορές έχουμε αντιδράσει κιόλας, ιδίω για κάποιες παραχωρητικές συμβάσεις, όπου αρνηθήκαμε και πρέπει να έχουμε υπόψη ότι στα προγράμματα των ορυχείων ε, συγχρηματοδοτούμε συνήθως 15% του αρχικού ποσού που μας ζητάτε και σε κάποιες περιπτώσεις αρνηθήκαμε ολοσχερώς την ε, ε, χρηματοδότηση γιατί θεωρούσαμε ότι ήταν λεόντιος η παραχωρητική σύμβαση. Το κράτος ελάμβανε τελικά πολύ λίγα εισοδήματα σε σχέση με το κέρδος που θα προέκυπτε από την ε, παραχωρητική σύμβαση. Όμω, σε ό,τι αφορά τι φοροαπαλλαγέ, αυτό έχει να κάνει με την αυτοδιάθεση του κάθε κράτου μέλου και την, ε, την κυριαρχία που διαθέτει. Κάποιε φορέ βρίσκουμε κι εμεί ότι είναι υπερβολικά γενναιόδοροι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να λάβει το λόγο. Τότε θα συνεχίσουμε με την ημερησία διάταξή μας. Ευχαριστώ τον ε, κύριο Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την έλευσή του εδώ και για την διάβγεια της ε, παρουσίασης του θέματος.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 Comment allez-vous you. Vous allez bien Good to see you. You're, you're, you're, you're just uh, next to your president. Mr. Peterson is uh, Swedish. Swedish, okay, thank you. It's now my pleasure. Με μεγάλη μου χαρά απευθύνω το καλώς ορίσατε στον κύριο Ζακ Ντιούφ, Γενικό Διευθυντή του ΦΑΟ, δηλαδή του Οργανισμού Επιστημισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών. καλώ ήρθατε στην Επιτροπή μα, σα προσκαλέσαμε στην ακροασή μα για τι συνέπειε τη οικονομική κρίση, στην επιστηστική ασφάλεια στις αναπτυσσόμενε χώρες. Επειδή όμως, ε, προσκαλέσει αύριο, επειδή όμω είστε ε, αύριο υποχρεωμένοι να λάβετε το αεροπλάνο, ε, θα ε, είχατε την καλοσύνη να έρθετε να μας δείτε σήμερα. Πολύ ωραία, σας δίνω μέσω το λόγο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι για μένα μεγάλη τιμή και προνόμιο να μπορώ σήμερα να απευθυνθώ στην ε, Επιτροπή σας. Ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω για την ε, ευγενική σας πρόσκληση. Οι οικονομίες του κόσμου ολόκληρου γνωρίζουν ύφεση και κάμψη. Κανένα κράτος δεν έχει αποφύγει κρίση και όπως συνήθως οι χώρες που είναι πλέον φτωχές και οι πληθυσμοί που γνωρίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες υποφέρουν περισσότερο. Το 2009 πάνω από ένα, δις, ε, ένα δισεκατομμύριο άτομα, δηλαδή ένα έκτο του παγκόσμιου πληθυσμού, υποφέρουν από πείνα. 105 εκατομμύρια περισσότερο από ό,τι πέρυσι. Η διεθνής επισητιστική κρίση προκλήθηκε από την απότομη αύξηση των τροφίμων, των βασικών ε, τροφίμων, η οποία έπληξε ιδιαιτέρως ε, εκατομμύρια ε, φτωχών ατόμων. Και παρά την κάμψη των, διεθνών, των τιμών διεθνώς τον περασμένο Ιούλιο, οι τιμές των βασικών τροφίμων παραμένουν σήμερα ιδιαίτερα αυξημένε στις αγορές των αναπτυσσόμενων χωρών εσωτερικά. Είναι ανώτερες οι τιμές αυτές από το 20% σε πραγματικούς όρους από ό,τι ήταν πριν την κρίση του 2006. Επιπλέον, οι γεωργοί ε, πλήγησαν από την αύξηση του κόστους ε, των, ε, των βοηθητικών ουσιών 176% για τα λιπάσματα 75% για τις ζωοτροφές και 70% για, τα, ε, για τις η εμπορευματοποίηση επίσης ε, των προϊόντων τους ε, υπέστη το κόστος της αύξησης των τιμών στις μεταφορές επειδή αυξήθηκαν και οι τιμές των καυσίμων. Κατά δεύτερον, η οικονομική κρίση ε, πλήττει ολόκληρο τον πλανήτη πλέον κατά τρόπο συγχρόνως μάλλον. Σε τέτοιε συνθήκες οι χώρες δεν μπορούν πλέον να ανατρέξουν στα κλασικά εργαλεία ή μέσα όπως η νομισματική υποτίμηση ή το δάνειο ε, για να αντιμετωπίσουν την κρίση. Επιπλέον, βάσει του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι ξένες επενδύσεις οι άμεσες ξένε επενδύσεις θα μειωθούν κατά 32% το 2009. Οι μετακινήσεις κονδυλίων προς τους ε, μεταναστεύοντες, από τους μεταναστεύοντες ε, εργαζομένους που ήταν της τάξης των 300 δις ε, Αμερικανών δολαρίων το 2008 μπορεί να γνωρίσουν πτώση 5 8% το 2009. Η ξένη βοήθεια προς τις 71 πλέον φτωχές χώρες θα μειωθεί κατά 25%. Και για να ολοκληρώσουμε αυτή τη ζωφερή εικόνα, ο όγκος των διεθνών συναλλαγών θα υποχωρήσει κατά 5 9% και οι τιμές των εξαγόμενων προϊόντων από τις αναπτυσσόμενες χώρες θα, μειωθούν κατά, θα μειωθεί κατά 15 26% το 2009. Τα φτωχά νοικοκυριά καταναλώνουν τώρα λιγότερο θρεπτικά τρόφιμα και αναγκάζονται να πολλούν τα μέσα που διέθεταν για την παραγωγή ή να απαρνηθούν την ε, υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση που τους ε, αναλογούσε. Κυρίε και κύριοι, κυρία Πρόεδρε, οι διευθυντικοί παράγοντε που προκάλεσαν την επιστημιστική κρίση του 2007 και 2008 συνεχίζουν να υπάρχουν. Η γεωργική παραγωγικότητα των φτωχών χωρών ε, και το έλλειμμα τροφίμων είναι σημαντικό. Δηλαδή η δημογραφική αύξηση έχει αυξηθεί, ενώ η πρόσβαση στις, ε, στα λοιπάσματα στη σημερινή εποχή, καθώ και στο νερό ή την καλλιέργεια των εδαφών ε, είναι σημαντικά προβλήματα. Οι πλημμύρε και οι ξηρασίε επίση έχουν ξεπεράσει τον ιστορικό όρο. Η σημερινή κατάσταση λοιπόν, η επισητιστική ανασφάλεια και τα αποτελέσματα τη αμέλεια έχουν οδηγήσει στην ε, επιδείνωση της γεωργίας στις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ ε, Χάνουν το 70% του μέσου αυτού που του εξασφάλιζε την επιβίωση οι φτωχότεροι κάτοικοι του πλανήτη. Η δημόσια βοήθεια για την ανάπτυξη που αφιερώνεται στην Γεωργία από 8 δι ε, Αμερικάνικα δολάρια το 1984 πέρασε σε 3,4 δι Αμερικάνικα δολάρια το 2004. Δηλαδή πραγματική μείωση 58% και το μερίδιο της γεωργίας ε, από την κρατική αναπτυξιακή βοήθεια μειώθηκε 17% από το 1980 σε 3,8% το 2006. Τώρα φτάνει το 5% στη σημερινή φάση. Η μόνιμη λύση θα ήταν να αυξήσουμε την παραγωγή και την παραγωγικότητα της γεωργίας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Για αυτόν τον σκοπό θα πρέπει να αυξήσουμε και τις επενδύσεις στον γεωργικό τομέα. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τις γεωργικές υποδομές των χωρών αυτών, ιδίω τον έλεγχο του νερού, την ε, άρδευση, τις, ε, τους, γεωργικούς, τους δρόμους της υπαίθρου, τις δυνατότητες αποθήκευσης, ε, τους λιμένες, τι υπηρεσίε μικροπιστώσεων κτλ. Η γεωργία των αντισώμενων χωρών χρειάζεται 44 δις αμερικάνικα δολάρια ετησίως για την, ε, από την κρατική αναπτυξιακή βοήθεια για επενδύσεις προκειμένου να ωφεληθούν οι μικροί παραγωγοί. Το ποσό αυτό όμως είναι πολύ περιορισμένο σε σχέση με τα 365 δις αμερικανικά δολάρια που δίνονται στους γεωργικούς παραγωγούς των χωρών του ΟΣΑ που δόθηκαν το 2008 και σε σχέση με τα 1.340 δις αμερικανικά δολάρια που δαπανώνται ετησίως στον κόσμο για τους εξοπλισμούς. Η διεθνής επισητιστική κρίση επέτρεψε ωστόσο την επιστροφή της γεωργίας ε, μεταξύ των πρώτων προτεραιοτήτων στην διεθνή ατζέντα. Για πρώτη φορά η πρωτοβουλία για την επισκεπτική ασφάλεια της συνόδου του G8 της ε, Λακίλα το περασμένο Ιούλιο, στην οποία είχα την τιμή να συμμετάσχω, έδωσε έμφαση στην γεωργική ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και προ όφελο των μικρών παραγωγών των αναπτυσσόμενων χωρών. Η δέσμευση που ανελήθη σε αυτήν ε, την σύνοδο ήταν να κινητοποιηθούν 20 δισαμερικανικά δολάρια μέσα σε μία τριετία για την γεωργία και την επισητιστική ασφάλεια και αυτό ήταν ένα ενθαρρυντικό μήνυμα προκειμένου βέβαια αυτή τη φορά να υλοποιηθεί στην πράξη και με ταχύτητα. Εγώ συνηγόρησα επί σειρά ετών, χωρίς πολλά αποτελέσματα, υπέρ των επενδύσεων στην μικρή γεωργία των φτωχών χωρών, προκειμένου να βρούμε μια βιώσιμη λύση στο πρόβλημα της επιστητικής ανασφάλειας. Ε, είμαι λοιπόν ιδιαίτερα ικανοποιημένος που σήμερα οι θύνοντες του G8 ε, συμμερίζονται αυτήν την άποψη. Θα πρέπει επίσης να βελτιώσουμε το σύστημα διακυβέρνησης της διεθνούς επιστημιστικής ασφάλειας. Από αυτή την άποψη, η αναθεώρηση της Επιτροπής για την Διεθνή Επισητιστική Ασφάλεια της ΦΑΟ, όπως είχε εγκριθεί ε, ομοφόνος τον περασμένο μήνα από τα κράτη-μέλη, για να γίνει πιο αποτελεσματική, είναι ένα σημαντικό βήμα. Μέσα σε μια εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι εργασίε του Παγκόσμια Συνόδου των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων για την επισητιστική ασφάλεια. Ελπίζω ότι αυτή η Σύνοδο θα καταφέρει να... μια ευρεία συνένεση για την απάλληψη, την πλήρη και ταχεία απάλληψη τη ε, εξάλληψη τη πείνα τη στον κόσμο. Οι χώρε τη Λατινική Αμερική και τη Καραϊβική έχουν ορίσει καταληκτική ημερομηνία το 2025. Το να αυξηθεί το μερίδιο τη γεωργία μεταξύ τη συνολική αναπτυξιακή βοήθεια, φτάνοντα στα επίπεδα μάλιστα το 1980, είναι κάτι το αναγκαίο. Όπω και το να υλοποιήσουμε μια πραγματικά αποτελεσματική διακυβέρνηση και διαχείριση τη διεθνού επιστημιστική ασφάλεια. Πρόσφατα, η ΘΑΟ έφερε ει πέρα δραστηριότητε στα πλαίσια τη πρωτοβουλία κατά τη ε, διόγκωση των τιμών των τροφίμων, πρωτοβουλία που ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2007 για να βοηθήσουμε του φτωχού γεωργού των αναπτυσσόμενων χωρών να έχουν πρόσβαση στα σύγχρονα μέσα, των οποίων, ε, τα σύγχρονα μέσα παραγωγή, των οποίων τιμέ αυξήθηκαν περισσότερο από ό,τι των τροφίμων. Ε, ο οργανισμό μα κινητοποίησε περισσότερα, περίπου μάλλον 400 εκατομμύρια δολάρια από του ίδιου πόρου του και τα ε, αποθεματικά τη. Η συμβολή 285 εκατομμυρίων δολαρίων ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της διευκόλυνσης, της επιστημιστικής διευκόλυνσης αποτέλεσε ένα σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας. Θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω την βαθιά με ευγνωμοσύνη προς την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και προς τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη γενοδορία τους. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα σημαντικότατος εταίρος της ΦΑΟ εξαιτία τη τεχνική συνδρομή και τη οικονομική συνδρομή που προσφέρει στι αναπτυσσόμενε χώρε στου τομεί τη γεωργία και τη ανάπτυξη τη υπαίθρου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πρωτοπόρος εταίρος της ΦΑΟ με μια συνεισφορά που το 2009 έφτασε τα 297 εκατομμύρια αμερικανικά δολάρια συμβάλλοντας έτσι στου εκτός στους εκτός προπολογισμού πόρους του οργανισμού μας. Ο ΙΦΑΟ λοιπόν ε, επιθυμεί και εύχεται να ενισχυθεί έτσι περαιτέρω η συνεργασία αυτή, η στενή συνεργασία που έχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα. Κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Σα ευχαριστώ κύριε Γενική Γραμματέ. Όπως είπα πριν έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Προτείνω λοιπόν να περιοριστούμε σε μία ερώτηση ανά πολιτική ομάδα, ώστε ο Γενικός Διευθυντής να μπορέσει να απαντήσει κιόλας. Να μου επιτρέψετε να αρχίσω με τον κύριο Γκέρενς που είναι ο μόνος ε, παρόν από την πολιτική του ομάδα αν από τη συνεδρίε, θα είχατε κερδίσει χρόνο, κυρία Πρόεδρε. Μια ερώτηση προ τον Γενικό Γραμματέα τη ΦΑΟ σε ό,τι αφορά τον τρόπο που θα μπορούσατε να επηρεάσετε την διακυβέρνηση αυτή, όπω την ονομάσατε, την επισητιστική. Συναντήθηκα με τον κύριο Λαμή πριν από κάποια χρόνια και συζητήσαμε για το αν θα έπρεπε να προτιμήσουμε υψηλές τιμές για τα τρόφιμα ή χαμηλές. Η αυξημένε τιμέ σημαίνει ότι ενθαρρύνουμε την παραγωγή, ενώ οι χαμηλέ ότι ενθαρρύνουμε του παρα... τους να παράγουν κι άλλο. Το θέμα λοιπόν είναι διεθνώ πώ θα χειριστούμε το θέμα αυτό και ο προβληματισμό μα δεν ήταν πώ θα χειριστεί το θέμα ο Διεθνή Οργανισμό Εμπορίου που πίεζε τι τιμέ προκειμένου να μειωθούν, αλλά το τι θα κάνει η Παγκόσμια Τράπεζα. Συνολικά λοιπόν, όλοι μαζί οι φορεί που επηρεάζουν τη διεθνή επιστημιστική διακυβέρνηση, ποια είναι η θέση και το βάρο τη ΦΑΟ σε αυτές τις ε, διαπραγματεύσεις και η Επιτροπή Παρακολούθησης των Εμπορικών Διαπραγματεύσεων. Νομίζω ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι μέλος ε, στην Επιτροπή αυτή και η Παγκόσμια Τράπεζα το ίδιο. Πού είναι λοιπόν η θέση της ΦΑΟ σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Ο κύριος Μπέρμαν από τους σοσιαλιστές après concertation Μετά από συνεννόηση επί της ουσίας μεταξύ μας, κύριε Ντιούφ, θα ήθελα να σας ρωτήσω τα εξής. Έχετε την εντύπωση ότι μετά την ε, επισητιστική αυτή κρίση γνωρίζουμε σήμερα αντιστροφή των ε, προεπαρχουσών τάσεων για τις επενδύσεις τον κόσμο της υπαίθρου, τη Γεωργία δηλαδή, και τις ε, περιοχές της υπαίθρου στις αναπτυσσόμενες χώρες. Εσείς ο ίδιος το είπατε, η Παγκόσμια Τράπεζα ε, γνωρίζουν την ανάγκη να χρηματοδοτηθεί η γεωργία. Η δυνατότητα αυτοπαραγωγής των αναπτυσσόμενων χωρών είναι σημαντική. Να έχουν τα τρόφιμα που τους χρειάζονται δηλαδή. Γνωρίζουμε σήμερα μια πραγματική αντιστροφή των ε, τάσεων, κάτι τέτοιο το διαπιστώνετε κι εσείς. Και ως προς αυτό τα κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδιαίτερως τιμούν και σέβονται τις υποσχέσεις που έχουν αναλάβει, τις οικονομικές τους υποσχέσεις. Ευχαριστώ. Εγώ θα λάβω το λόγο εξ ονόματο των Πρασίνων. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε Γενική Γραμματέα, εάν η ΦΑΟ έχει προβλέψει κάποιον κώδικα συμπεριφορά για την μακροπρόθεσμη κατανομή ή την αγορά αρωτρέων γιών. Και έχετε διεξαγάγει μελέτες για τη δυνατότητα να περιοριστεί η κερδοσκοπία για τις απαραίτητες πρώτες ύλες για τον, ανθρώπι, για τον ανθρώπινο επισητισμό είτε από, από περιπτώσεις ψευδοσυμβάσεων είτε από, με άλλα μέσα και τώρα κυρία Στίφλερ ναι, με μια σύντομη ερώτηση. Η ΦΑΟ είναι βασικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών με ένα δις ευρώ. Ακούσαμε ποια κονδύλα κινητοποιήθηκαν στα πλαίσια της διευκόλυνσης της επισητιστικής. Πώς προβλέπετε λοιπόν, πώς αποτιμάτε τη μέχρι τώρα πρόοδο της διευκόλυνσης αυτής και πιστεύετε ότι το εργαλείο αυτό θα συμβάλλει σημαντικά ώστε να αυξηθεί η παραγωγή τροφίμων, ιδίω για τους μικρούς ε, καλλιεργητές της χώρας προτεραιότητας. Και ο κύριος Ντέβα, τελευταίος παρεμβαίνουν. Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το νερό για τον εγώ. Εργάζεστε στο ΦΑΟ για να εξετάσετε την έλλειψη ύδατος που αντιμετωπίζετε. Πρόσφατα υπάρχει και έκθεση ότι σε σχέση με τους παγετώνες που λιώνουν και σε σχέση με τον πραγμαπούτρα, τον Κίτρινο Ποταμό και θα έχουν λιγότερο νερό για άρδευση Κάνοντας λόγο για τρόφιμα και γεωργία, δεν μπορούμε να τα αποσυνδέσουμε. Υπάρχει ανάγκη για το νερό. Πώς το βλέπετε αυτό. Ευχαριστώ. Κύριε Γενική Γραμμα... Ε, Διευθυντά, τον λόγο. Χωρίς μικρόφωνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να απαντήσω σύντομα, διότι δεν έχω πολύ χρόνο, για την επιστημιστική διακυβέρνηση. Είναι σήμερα ένα από τα μείζωνα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν πολλοί εταίροι εδώ. Οι εταίροι που χρηματοδοτούν τη γεωργία και την ανάπτυξη. Εδώ είχαμε τα σοβαρότερα προβλήματα. Διότι περάσαμε το 17% αναπτυξιακής βοήθειας που πήγαινε στη γεωργία τη δεκαετία του και είχε επιτρέψει να γίνουν επενδύσεις για την πράσινη επανάσταση στην Ανασία και την, Αμερική, τη Λατινική Αμερική και έπειτα είχαμε δραστική μείωση, 3,8% σήμερα φτάσαμε. Ή μάλλον από το 3,8% πρόσφατα περάσαμε στο 5% σήμερα. Είναι σοβαρό. Και εδώ αυτό αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι στο 1 το αναπτυξιακό ταμείο υπήρχε 4,5% πόρων που απευθύνονταν στη Γεωργία. Είναι ένα πρόβλημα γενικότερο των τραπεζών και των βοηθειών των πολυμερών. Δεύτερη σειρά εταίρων, δεύτερη κατηγορία εταίρων, αυτοί που παρεμβαίνουν στο κομμάτι του εμπορίου. Ιδίω ο ΠΟΕ, αλλά και οι περιφερειακές συμφωνίε που διέπουν το εμπόριο. Κοινέ αγροτικές πολιτικέ και το καθεξή. Εδώ έχουμε δράσεις ε, που έχουν να κάνουν και με τους δασμούς, τελωνιακούς δεσμούς, τεχνικούς φραγμούς στο εμπόριο έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ούτω καθεξής. Τρίτη κατηγορία εταίρων, παραγόντων εδώ, οι ε, εταιρικές σχέσεις για την αναπτυξιακή βοήθεια που επηρεάζουν και τα επισητιστικά Πρόκειται για οικονομικές βοήθειες, πρόκειται για βοήθειες χειροπιαστές, εξαρτάται από το γίνονται και οι αγορές. Υπάρχουν εξειδικευμένοι οργανισμοί για τη χρηματοδότηση της γεωργίας, όπως φαίνεται, αλλά η πόρη της είναι περιορισμένη από το παγκόσμιο Τράπεζα και σε σχέση με τις αναπτυξιακές τράπεζες οι οποίε παρεμβαίνουν και αυτέ στην όλη διαδικασία. Και σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν προφανώ και κυβερνήσει. Κυβερνήσει με τι αποφάσει του για τον προπολογισμό του, τον εθνικό του προπολογισμό και για την πολιτική που θα ακολουθήσουν, α πούμε, στη Γεωργία. Όλα αυτά μαζί πρέπει κανεί να τα συνδυάσει, να τα εξετάσει από κοινού για να καταλάβει τι συμβαίνει και να εξετάσει τι συμβαίνει ω προ την επισητιστική ασφάλεια διεθνώ, ε, να προβλέψει τι τάσει θα διαμορφωθούν στο μέλλον και να προβλέψει λύσει σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, τι μη κυβερνητικέ οργανώσει και τι ενώσει παραγωγών. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στα πλαίσια τη μεταρρύθμιση ε, τη Επιτροπή τη Διεθνού Επιστημιστική Ασφάλεια για να αξιοποιήσουμε καλύτερα την παρουσία όλων αυτών των εταίρων και να συζητήσουμε καλύτερα τι καταστάσει όπω τη σημερινή. Τόσα εκατομμύρια άτομα που υποφέρουν από πείνα στον κόσμο, 10% αύξηση παραγωγή τροφίμων ε, και 9 δις δις ε, αμερικάνικα, ε, μάλλον άτομα, άτομα στον κόσμο, πληθυσμό στον πλανήτη. Θα πρέπει λοιπόν να διπλασιάσουμε την παραγωγή τροφίμων στι αναπτυσσόμενε χώρε ω τότε. Σε ό,τι αφορά τώρα την αντιστροφή των τάσεων, πρέπει να πω ότι για τις επενδύσεις υπάρχουν κάποιες μικρές αλλαγές. Αλλά δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί από την κρίση του 2007 έως 2008 έχουμε φτάσει μόνο στο 2009. Δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερες προβλέψεις, αλλά υπάρχουν κάποιες θετικέ τάσεις. Μια τάση ανανέωσης, ανάκαμψης των επενδύσεων για τη Γεωργία. Τώρα, η ερώτηση για την αγορά και την ε, κατανομή των γεών. Θα γνωρίζετε ότι ήμουν από τους πρώτους που επεσήμαναν το πρόβλημα στη διεθνή κοινότητα με άρθρο στην Μόντ, που μεταφράστηκε και στη Financial Times. Από τις υπηρεσίες μας έγινε διεξήχθη μελέτη με συνεργασία και άλλων εταίρων όπως το ΦΙΝΤΑ για να δούμε πώς μπορούσε να οργανωθεί κάτι τέτοιο στην πράξη. Τα αποτελέσματα ήταν ανησυχητικά. Έχουμε λοιπόν αρχίσει να επεξεργαζόμαστε σε συνεργασία με την Ιαπωνία και άλλες χώρες για να φτάσουμε σε έναν κώδικα συμπεριφοράς σε ό,τι αφορά τις γεωργικές επενδύσεις στις χώρες του τρίτου κόσμου. Διότι από τη μια οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι αναγκαίες αλλά και χρήσιμες εάν θέλουμε να διπλασιάσουμε την παραγωγή τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Πρέπει όμως να βεβαιωθούμε ότι αυτό θα γίνει στα πλαίσια ανταλλαγών που δεν θα είναι παράνομες ή δεν θα επιτρέψουν την κερδοσκοπία. Κάποιοι δεν θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τη θεσμική αδυναμία, την ανθρώπινη αδυναμία κάποιων ε, χωρών. Για την κερδοσκοπία στις αγορές τροφίμων, τις γεωργικές αγορές, ναι, τη μελετήσαμε σε συνεργασία με άλλους εταίρους, όμως ως σήμερα δεν εξήβραμε καμία λύση διότι μιλάμε για αγορές χρηματιστηριακές πια. Στο Σικάγο γίνονται τέτοιου είδους κερδοσκοπικές ε, δράσεις. Ε, μετακινούνται κονδύλια προς τον τομέα των ακινήτων ή άλλους τομείς και Είδαμε σε περίοδους κρίσης ε, τέτοια επενδύσεις να γίνονται προς το γεωργικό τομέα. Με την διεθνή κρίση επίσης πάλι υπάρχει μετακίνηση προς άλλες κατευθύνσεις. Δεν μπορούμε λοιπόν να τα εμποδίσουμε όλα αυτά, ούτε να είμαστε αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Για το δις ευρώ, η ΦΑΟ προς στιγμήν υλοποιεί, μάλλον χρησιμοποιεί 280 δις ε, εκατομμύρια μάλλον δολάρια, 280 εκατομμύρια δολάρια που μπορούμε να εκταμιεύσουμε και μας ικανοποιούν ιδιαίτερα οι συνθήκες υπό τις οποίες συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή. Διότι για πρώτη φορά είχαμε αυτό που πάντοτε ζητούσαμε, δηλαδή κονδύλια προσανατολισμένα προς την συνδρομή των γεωργών των φτωχών χωρών. Εκεί που υπάρχει αυτό το δις ατόμων που πεινούν, που χρειάζονται να παράγουν καλύτερα με λιπάσματα, με ζωοτροφές σε μια πρώτη φάση και σε μια δεύτερη φάση με την απαραίτητη συνδρομή για να μπορέσουν τα εθνικά τους παραγωγικά συστήματα παραγωγή σπόρων, πιστοποίηση σπόρων, ε, βελτίωση των ποικιλιών που καλλιεργούνται στα ερευνητικά τους κέντρα, να τα υλοποιήσουν όλα αυτά. Αυτό το κάνουμε λοιπόν και με τα λοιπάσματα αλλά θέλουμε να περάσουμε και στη φάση της σύνθεσης λιπασμάτων στις χώρες καλλιέργειας και εκμετάλλευσης των εδαφών. Σε μια τρίτη φάση, εάν χρειαστεί, μπορεί να έχουμε και παραγωγή των λιπασμάτων εκεί. Σε χώρες που διαθέτουν ε, πετρελαϊκά κοιτάσματα, διηληστήρια ή κοιτάσματα σε φωσφορούχες ενώσεις ή άλλες λοιπασματικέ ουσίε. Πάντω, ελπίζουμε ότι θα υπάρξει ενοποίηση όλων αυτών των προσπαθειών. Ε, όχι μόνο διεύρυνση, αλλά και ενίσχυση σε ό,τι αφορά τι δεσμεύσει που ελήφθησαν στην Ιλακύλα. Ε, για να κινητοποιήσουμε 22 δι δολάρια σε μια τριετία, 2009, 2010, 2011 και ένα μέρος αυτής της συμβολής προφανώς θα προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζουμε λοιπόν ότι η πείρα που θα αποκομίσουμε και η παρακολούθηση των μέχρι τώρα προσπαθειών μας μαζί με μελέτες επιπτώσεων για κάθε ένα από τα προγράμματα ελπίζουμε ότι όλα αυτά θα προσφέρουν και στους δικαιούχους, δηλαδή στους ίδιους τους γεωργούς, τους εισαγωγείς, όλα αυτά τα δεδομένα θα επιτρέψουν να ενισχύσουμε και να διευρύνουμε αυτού του είδους τις δράσει που νομίζω ότι είναι οι μόνες που καταλήγουν σε αηφορά αποτελέσματα για το θέμα του νερού. Προφανώς το νερό είναι πηγή τη ζωής. Για τους ανθρώπους, για τα ζώα ή για τι καλλιέργειε. Για τα στήρα. Λοιπόν, μια από τι πρώτε μας προτεραιότητε είναι να ενθαρρύνουμε την ε, χρήση καθαρού νερού, Ιδίω στην Αφρική, όπου μόνος, ε, μόνο 7% των αρωτρέων γεών αρδεύονται έναντι του 30% στην Ασία. Και στην υποσαχάρη Αφρική είναι 4% μόνον. Δηλαδή 96% της γης εξαρτάται από τι βροχοπτώσει, από την καλλιέργεια δηλαδή, εξαρτάται από τι βροχοπτώσει. Και υπόκειται στη, στα φαινόμενα των κλιματικών αλλαγών και τις ακραίες μεταβολές του καιρού. Επιπλέον, θα γνωρίζετε ότι οι κλιματικές αλλαγές θα δυσχεράνουν περισσότερο το πώς ε, τα αρχικά αποθέματα νερού ε, και αυτό λέω και των ξηρασιών και αυτό θα δημιουργήσει και σοβαρά πολιτικά προβλήματα. 40% του πόσιμου ύδατος ε, στον κόσμο βρίσκεται εκτός συνόρων. Αυτό δημιουργεί λοιπόν τεράστιους ανταγωνισμούς σε διεθνή κλίμακα. Αυτά όλα θα οξυνθούν με την αύξηση του πληθυσμού δηλαδή τα 9,2 δις ε, κατοίκων που υπολογίζουμε μέχρι το 2015. Σας ευχαριστούμε, Γενική Διευθυντά, για τις ε, παρατηρήσεις σας. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Καλή σας ε, υπομονή και κουράγιο για την τόσο σημαντική σας δράση. Να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στη Μοζαμβίκη. Okay. 28 Οκτωβρίου φέτος είχαμε τρεις ε, σειρές εκλογών ταυτόχρονα στη Μοζαμβίκη και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αποστείλει παρατηρητές. Η κυρία Όλ ήταν ε, η υπεύθυνη των παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο κύριος Πέντα ήταν υπεύθυνο των παρατηρητών από πλευρά Κοινοβουλίου. Σήμερα λοιπόν θα θέλαμε την αποτίμηση της κυρίας Φιώνα Χολ που έχει αποστείλει την προκατακτική της έκθεση διότι η έκθεση αυτή καθεαυτή θα δημοσιευτεί μετά από ένα δίμηνο. Δυστυχώς η κυρία Χολ ζητά συγγνώμη από όλους μας διότι είναι ασθενής. Δεν θα έχουμε τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας. Όμως μαζί μας είναι ο κύριος Κριστιαν Πρέντα. Περιμένοντας λοιπόν την οριστική έκθεση, την έκθεση στην οριστική της μορφή, να δώσω το λόγο στον κύριο Κριστιαν Πρέντα για να μας παρουσιάσει τις προκατακτικές του παρατηρήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε πολύ σύντομα να παρουσιάσω τα λιγοστά συμπεράσματα μου από την επίσκεψη της αντιπροσωπείας μας που αποτελούσαν πολλά μέλη του Κοινοβουλίου. Συγκεκριμένα ήμασταν επτά. Ο κύριος Φερνάντες, ο κύριος Μπόντο από το ΕΛΚ, ο κύριος Τυρολιά και ο κύριος Μορέιρα και ο κύριος Αλβάρες από τους σοσιαλδημοκράτες, τους σοσιαλιστές και δημοκράτες μάλλον. Ο κύριος Πόρτας από την ΚΟΕ. Παρατηρήσαμε λοιπόν την διεξαγωγή των εκλογών στη Μοζαμπίκη και όπως είπατε και εσείς, οι εκλογές έλαβαν χώρα την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου. Ο κύριος Μπέρμαν, που θα ερχόταν μαζί μας και θα προείδρευε της ομάδας μας, αναγκάστηκε να συμμετάσχει σε άλλη επίσκεψη για τις εκλογές στο Αφγανιστάν τελευταία στιγμή, οπότε αντικαταστάθηκε από τον κύριο Άλβες, όπως σας είπα, λέει Παόλο Άλβες. Είχαμε τρεις γύρους εκλογών για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, για το Κοινοβούλιο και εκλογές για τις τοπικές βουλές. Η αντιπροσωπεία μας την ημέρα των εκλογών μετέβη σε διάφορα εκλογικά κέντρα και τα επτά μέλη της αντιπροσωπείας χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Μία έμεινε στο Μαπούτο, την πρωτεύουσα, μία δεύτερη παρατήρησε τι έγινε στα προάστια της πρωτεύουσα και μια τρίτη πήγε στην Πέιρα, τη δεύτερη πόλη της χώρας. Στην Πέιρα, διότι ο δήμαρχος αυτής της μεγάλης πόλης ήταν ένας από τους βασικούς υποψήφιους για τις προεδρικές εκλογές. Ιδρυτής κόμματος, το Δημοκρατικό Κίνημα της Μοζαμπίκης και μέλος του Ρενάμου. ένα από τα δύο βασικά κόμματα που αναμετρήθηκαν στις εκλογές. Εκτός μικροφώνου ο το βράδυ εκείνης της ημέρας ξανασυναντηθήκαμε σε διάφορα εκλογικά κέντρα για να καταμετρήσουμε τις ψήφους. Ήταν μια διαδικασία αρκετά χρονοβόρα, κράτησε και πολύ και κάποιες φορές ήταν και πολύ περίπλοκη. Η καταμέτρηση 200-300 δελτίων κράταγαν 6-7 ώρες, διότι έπρεπε να λάβουμε τεράστιες προφυλάξεις για την καταμέτρηση. Υπήρχαν πάρα πολλοί περιορισμοί. Σε γενικέ γραμμέ, αυτό που εμεί διαπιστώσαμε επί τόπου για τη διεξαγωγή των εκλογών στα εκλογικά κέντρα ήταν ένα κλίμα ήρεμο, εμπιστοσύνη. Οι πρόσωποι των βασικών κομμάτων ήταν πάντοτε παρόντε. Και ήταν καλή η διοργάνωση. Ακόμη και αν η συμμετοχή ήταν ε, κατώτερη από τις προηγούμενες εκλογές. Υπήρχαν σε κάποιες περιπτώσεις και ωραίες αναμονής, αλλά αυτή ήταν η εξαίρεση. Πριν τις εκλογές συναντηθήκαμε με τους βασικούς ε, υποψηφίους για τις προεδρικές εκλογές, τους τρεις υποψηφίους του Φρέλιμο, του Ρενάμο και του MDM ο πρόεδρος Κουεμπούζα ήταν ε, υποψήφιος του Φελιμό, ο κύριος Νακάμα για το Ρεναμό και ο κύριος Σιμάγκο για το MDM. Συναντηθήκαμε επίσης και με τους παρατηρητές που ήταν μέλη της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την αγίδα της κυρίας Χολ και με άλλους παρατηρητές εθνικούς όπως πρέσβης ε, χωρών ε, δωρητριών και τον πρόεδρο της ε, Εθνικής Εκλογικής Επιτροπής. Αποσπάσαμε λοιπόν πολλέ πληροφορίε για την διεξαγωγή, την διοργάνωση μάλλον των εκλογών, για, τις νομικούς, για του κανόνε τη νομοθεσία, για την διάσταση των μέσων μαζική ενημέρωση. Όλα αυτά τα καλύπτει η ενδιάμεση έκθεση στο preliminary statement, στην προκαταρκτική δήλωση που υπέβαλε η κυρία Φιώνα Χολ Στις 30 Νοεμβρίου λέει ο μιλητή, ίσως εννοεί Οκτωβρίου. Ευχαριστούμε λοιπόν την κυρία Χολ και τους συνεργάτες της, τους ε, παλιούς αυτούς συνεργάτε τη, που βρέθηκαν επίσης στη χώρα αυτή από εβδομάδες ε, νωρίτερα για να παρακολουθήσουν τις τεχνικές διοργάνωσης των εκλογών. Δύο στοιχεία να τονίσουμε. Το πρώτο, κάπω ε, ευαίσθητο σημείο, διότι βρεθήκαμε ενώπιν μια κατάσταση μα έφερε σε δύσκολη θέση. Κάποια μέλη τη αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου δεν συμφωνούσαν καθόλου με τα συμπεράσματα τη αποστολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση που βρέθηκε στη Μοζαμβίκη επί σειρά εβδομάδων και ανέλησε τι διάφορε πτυχέ νομοθετικέ, επικοινωνιακέ των υποψηφιωτήτων, Δεν συμφωνούσαν λοιπόν με την προκαταρκτική αυτή δήλωση της κυρίας Χόλ. Όπως ε, δημορφώθηκε αμέσως μετά τις εκλογές. Αλλά βάσει της πείρας που συγκεντρώθηκε επί σειρά εβδομάδων, όπως είπα. Έτσι λοιπόν, κατά τις συζητήσεις μας, ευθύς εξ αρχής, τα μέλη της αντιπροσωπείας δεν συμφώνησαν, δεν υπήρχε συνένεση για την έκθεση της αποστολής συνολικά. Έτσι, η έκθεση αυτή, η προκαταρκτική δήλωση δεν στηρίχθηκε. Δεν στηρίχθηκε από τα μέλη της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας, που ωστόσο συμμετείχε στην ευρύτερη αποστολή επίσκεψης της Ένωσης. Αυτό δημιούργησε λιγάκι, όχι εντάσεις, αλλά κάποια μικρή συγκίνηση και εν τέλει χρειάστηκε να συμβιβαστούμε η κυρία Φιώνα Χολ παρουσίασε τα συμπεράσματα του ή άλλω τη επίσκεψη και σε ό,τι αφορά την κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία περιοριστήκαμε στο να σχολιάσουμε και να αποτιμήσουμε μόνο την ημέρα της διεξαγωγής των εκλογών και τονίζουμε, όπως έκανα εγώ στην κοινή συνέντευξη τύπου, υπογραμμίσαμε δύο σημαντικές πτυχές το γεγονό ότι κατά τη διάρκεια τη ημέρα τη διεξαγωγή των εκλογών οι κάτοικοι τη Μοζαμβίκη εκφράστηκαν ελεύθερα, δεν υπήρξαν περιορισμοί ούτε φραγμοί ε, κατά τη ελευθερία έκφραση τη ψήφου του. Και επίση σημειώσαμε τη συμμετοχή ιδιαίτερα των νέων στην εκλογική διαδικασία και μάλιστα των γυναικών, όχι μόνο στι εκλογέ και τη διεξαγωγή τους, αλλά και στα εκλογικά κέντρα, όπου πολλές φορές ήταν ε, συμμετέχουσες και πρόεδροι των εφορευτικών επιτροπών. Ιδού, λοιπόν, ε, πρόεδρε, τα της δημοσίευσης της έκθεσης που ακόμη δεν είναι πλήρης. Παραμένει, βέβαια, ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι αποστολές που βρίσκονταν στη χώρα από, την από εβδομάδες, από περισσότερο καιρό δηλαδή, είναι ο συνδετικός κρίκος, είναι το σημείο αναφοράς για τις μικρότερες αποστολές, τις ολιγάριθμες μέλη αποστολές, όπως η κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία που πήγαν εκεί για την ημέρα των εκλογών, αλλά αποτελούν μέρος της ευρύτερης αντιπροσωπείας τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ υπάρχουν και άλλα μέλη. Ο κύριο Τυρολιά είναι εδώ. Να ευχαριστήσουμε τη Γραμματεία για τη συνεργασία τη. Είμαστε και άλλοι εδώ πάντω και παραμένουμε στη διάθεσή σα εφόσον έχετε ερωτήσει. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Η Επιτροπή. Θέλετε το λόγο για αυτή την επίσκεψη στην Μοζαμβίκη. Όχι. Ναι. Είμαι ο κύριο Νορμό ε, και νομίζω ότι η κυρία Χολ κανονικά θα έπρεπε να είναι εδώ για να λάβει το λόγο και να απαντήσει σε ε, ερωτήσει εφόσον υπάρχουν. Δεν είμαι ο αρμόδιο. <coughs> κύριε Ντέβα, ε, ευχαριστώ πρώτα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπρέντα για την έξοχη ανάπτυξη του θέματος. Έχω συμμετάσχει σε πολλές παρατηρήσεις εκλογών. Έχω μία απλή ερώτηση. Οι ευρωβουλευτές σε πόσα εκλογικά τμήματα μετέβησαν. και πόσα εκλογικά τμήματα, σε πόσα εκλογικά τμήματα παρατήρησαν τις εκλογές οι μακρόχρονοι παρατηρητές την ημέρα των εκλογών. Κύριε Κάσμαν, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μπορώ και να απαντήσω στον κύριο Ντέβα. 782 σε 84 οι, οι παρατηρητές και οι βαρχιπρόθεσμοι και οι μακροπρόθεσμοι. Και υπάρχει ε, ε, ένα μείγμα και γι' αυτό κάνω και μια ερώτηση ως πρώην επικεφαλής ε, αποστολής παρατηρήσεως ε, πρόκειται για μια χώρα που παρατηρήθηκε για περισσότερο από λίγες μέρες και πρώτων εκλογών και στη διάρκεια των εκλογών. Και πάντως οι αποστολές παρατήρησης εκλογών είναι πολύ σημαντικές και κυρίως για το τμήμα εκείνο που είναι η μακροχρόνια παρατήρηση, η μακρού χρόνου μάλλον παρατήρηση για την συλλογή πληροφοριών, την ανάπτυξη σχέσεων με τις ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις, με τις εκλογικές αρχές κτλ. Και επίσης την παρακολούθηση των μέσων ενημέρωσης. Διάβασα το προκαταρκτικό, την προκαταρκτική δήλωση που τη βρίσκω εξαιρετική και είναι βασισμένη στο νέο πρότυπο που νομίζω ότι εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και η ερώτησή μου, επειδή δεν περιλαμβάνεται στην ίδια τη δήλωση, λέει ότι ήταν επαρκή τα μέτρα διαφάνειας σε σχέση με τι σε σχέση με την ίδια την ψηφοφορία ή σε κάποιο επίπεδο άνω των εκλογικών τμήματων. Και για να μπορέσει να γίνει μια μακροχρονότερη ε, ανάλυση των αποτελεσμάτων αυτών των, παρατηρη... εκλογών, των, ε, των παρατηρήσεων, νομίζω θα ήταν καλό Πάντως σίγουρα στην προκατακτική δήλωση καλά θα είναι να μπαίνει και ο αναπληρωτής επικεφαλής της ε, ε, αποστολής παρατήρησης εκλογών και οι, εκείνοι που αποτελούν τον πυρήνα και οι οποίοι θα είναι ίδιοι για τα πέντε χρόνια της θητείας είτε το πουλ είναι μεγαλύτερο είτε είναι πιο στενό και όταν γίνει πολύ στενό τότε ίσως θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Δεν αναφέρομαι σε προβλήματα που ενδεχομένω να ε, αντιμετώπισα εγώ, αλλά καμιά φορά πηγαίνει κανείς με μια προκατηλημένη άποψη και τότε ε, μπορεί να τίθεται σε εμφιβολία και ολόκληρη η προσπάθεια της ε, αποστολής παρατήρησης εκλογών. Ο κύριος Κάτσμαρεκ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να ε, πω για αυτή την έκθεση ότι συμφωνώ με τον κύριο Κάσμαν ότι οι μακροπρόθεσμοι παρατηρητές έχουν ιδιαίτερη σημασία. Ένα θέμα είναι εδώ το οποίο με ανησυχεί κάπως σε σχέση με αυτή την τοποθέτηση, την αρχική δήλωση. Οι αναφορές σε σχέση με τα ηλεκτρονικά μέσα ε, σε σχέση με πριν από τις εκλογές 44 45% λέγεται του χρόνου εχμής των μεγαλύτερων τηλεοπτικών σταθμών είχαν δοθεί στο κυβερνητικό κόμμα ενώ το υπόλοιπο χρονικό κομμάτι ήταν αφιερωμένο στα υπόλοιπα κόμματα και εδώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη μια ισορροπημένη ε, προσφορά. Ας το πούμε όμως ειλικρινά. Αν είχαμε μια τέτοια κατάσταση στην Ευρώπη σε ένα από τα κράτη-μέλη, αν το κυβερνόν κόμμα χρησιμοποιούσε 45% του χρόνου εχμής ε, σε ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και λέγαμε ότι αυτό θα ήταν ισορροπημένη προσέγγιση, ε, θα είμαστε φρενοβλαβείς να ισχυριζόμαστε κάτι τέτοιο. Εδώ λοιπόν υπάρχουν διπλά μέτρα και σταθμά για την Αφρική. 45% για το κυβερνών κόμμα θεωρείται εύλογο. Τι γίνεται εδώ. Ίσως θα πρέπει απλά τα αντικειμενικά γεγονότα να παρουσιάζονται χωρίς να ε, ακολουθούνται από σχόλια όπως αυτό του ότι ήταν ισορροπημένη αυτή λέει η παρουσίαση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Φρέντα. Θέλετε να παρέμβετε για ένα σχόλιο. Euh, ναι, πολύ σύντομα με τις ελάχιστες πληροφορίες που διαθέτω βέβαια να πω δύο λόγια τα μέλη της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου, τα μέλη, οι βουλευτές, όπως προείπα, συμπεριλήφθησαν στη μεγαλύτερη ομάδα των παρατηρητών, γι' αυτό και η δήλωση. Συνολικά τα μέλη της αποστολής του Κοινοβουλίου μετέβησαν σε περίπου 60, 70 μάλλον, εκλογικά κέντρα, από τα 780 εκλογικά κέντρα που συνολικά επισκέφτηκαν οι υπόλοιποι παρατηρητές, παρατηρητές όλοι μαζί. Εντάξει, ήταν ε, σίγουρα μειοψηφία, 131 ήταν τα μέλη της αποστολής, ήμασταν 7, ε, καλύψαμε ένα μικρό μέρος στις τρεις βασικές περιφερειές που σας ανέφερα. Πρωτεύουσα, προάστια της πρωτεύουσας και Μπέιρα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις διάφορες πτυχές της διεξαγωγής των εκλογών αναφέρονται κατά τρόπο μεθοδικότατο στην έκθεση που υπέβαλε η κυρία Χολ. Υπήρξαν προβλήματα διαφάνειας ε, ως προς τη διαδικασία που ε, εφαρμόστηκε για την ε, καταγραφή λόγου χάρη των υποψηφιωτήτων. Αυτό που έκανε εντύπωση στους παρατηρητές, στους επιτόπιους παρατηρητές, ήταν τεράστιος αριθμός υποψηφίων που δεν μπορούσαν να εγγραφούν, τους αρνήτο η συμμετοχή. Μάλλον τους αρνήθηκαν τη συμμετοχή. Ε, αυτό είναι θέμα της εκλογικής αρχής. Σημαίνει ότι ο νόμος ο εκλογικός κατασκευάστηκε με τρόπο σοβαρό μεν, αλλά ως ε, κώδικας ορθολογικός που έπρεπε να εφαρμοστεί κατά γράμμα. Σε λοιπόν ε, η υποψηφιότητα απορρίφθηκε έλεγαν ότι Μα ζητούν να είμαστε σοβαροί, είμαστε κι εμεί σοβαροί, ετοιμάζουμε ένα πολύ καλά διαρθρωμένο κείμενο και βάσει το κείμενο αυτού μα απορρίπτουν την υποψηφιότητα. Εκεί όμω δεν μπορούσε κανεί να προβάλλει αντιρρήσει εφόσον όλα έγιναν σεβαστά κατά τρόπο πολύ αυστηρό. Έπειτα από την πλευρά του κόμματο του κυρίου Νταβίση Μάγκο, το δημοκρατικό κίνημα τη Μοζαμβίκη, το MDM, υπήρξε δυσαρέσκεια και εκφράστηκε η δυσαρέσκεια αυτή και για αυτή την περίπτωση της απόρριψης ε, των ψηφιοτήτων και για εκφοβισμούς από το κυβερνών κόμμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το τοπίο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ε, ο κύριος Κάσμαν παρατήρησε κάτι που και εδώ έχει σημειωθεί, ότι το κυβερνών κόμμα είχε περίπου 46,5% Ενώ 54-55% είχαν τα υπόλοιπα κόμματα όλα μαζί. Η Μοζαμβίκη είναι μια χώρα όπου δυσπόζει το φρέλιμο ως κόμμα. Έχει σοβαρή κοινοβουλευτική παρουσία, οπότε και με την ε, λογική των αναλογιών που ακολουθήσαμε και εμείς φαινόταν ε, το αποτέλεσμα να είναι ρεαλιστικό. Και βάσει των εκτιμήσεων ε, που είχαμε. Βέβαια τα πραγματικά αποτελέσματα δεν παρουσιάζονται εδώ, αλλά γενικώ υπάρχει πραγματικά μια πρωτοκαθεδρία του κόμματο Φρέλιμο με τον κύριο Γκουεμπούζα, Αρμάντο Γκουεμπούζα, ο οποίο ξεπέρασε το 70% των ψήφων. Είδου, νομίζω ότι κατά τα άλλα η έκθεση της κυρίας Φιώνα Χολ είναι σαφέστατη. Για άλλη μια φορά να, ευχαριστήσω για το, να την ευχαριστήσω για το εξαιρετικό της έργο επιτόπου και όλα τα μέλη της αποστολής. Ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε τώρα στο τελευταίο μας. Α, όχι, ξέχασα, ξέχασα. Ένα... Κύριε Κάσμαν. Uh, miss... όχι, δεν με ξεχάσατε ακριβώς. Ανα έκανα μια ερώτηση που νομίζω ότι απευθυνόταν προς την Κομισιόν. Εάν δηλαδή θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα σχετικά με την συμπερίληψη στην της προκαταρκτική ε, δήλωση και στο τέλος ε, το όνομα του αναπληρωτήου ε, επικεφαλής της αποστολής ή και του λεγόμενου core team της ομάδας πυρήνα δηλαδή. Ναι, δεν βλέπω να είναι και τεράστιο το πρόβλημα. Ορισμένοι επικεφαλής αποστολών παρατηρητήσεων μπορεί να μην είναι σύμφωνοι αλλά έχουμε, ε, όπως για παράδειγμα ε, σε παρατηρήσεις στο Αφγανιστάν, δεν βάζουμε το όνομα για λόγους ασφαλείας, αλλά ε, κατά τα άλλα, ναι, και μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό. Όπως είπα όμως, θα πρέπει να το αποφασίσει η ίδια επικεφαλής της αποστολής. Πολύ σύντομα κυρία Πρόεδρε, πάλι ο Δεν θεωρώ ότι πρέπει ε, ο ίδιος η ίδια η επικεφαλής της παρατηρήσεως να ε, αποφασίσει, γιατί πρόκειται χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων, τα οποία χρησιμοποιούνται και με πολύ καλό τρόπο, μάλιστα στην περίπτωση αυτή. Χρειαζόμαστε λοιπόν απόλυτη διαφάνεια. Ο πιο απλός τρόπος είναι να μπει το όνομα του ε, αναπληρωτή και, το, και της ομάδας πυρήνα σε ένα παράρτημα. Ελπίζω ότι αυτό θα το δεχτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, υπέρ της διαφάνειας. Και θα είναι και σύμφωνη με τον κανονισμό 1049 του 2001 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα. Καλά. Προχωρούμε λοιπόν τότε στο επόμενο ε, θέμα της σημερινής διάταξης που προβλέπεται να διαρκέσει μια μισή ώρα γιατί είναι και πολύ σημαντικό. Όσοι ημών ε, θα αποχωρήσετε τις ευθούσεις στη διάρκεια της συζήτησης του θέματος αυτού, να ξέρετε ότι και η αυριανή μέρα είναι πολύ σημαντική και να είστε παρόσες και παρόντες. Θα εξετάσουμε τώρα την συνοχή, συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ και την, αναπτυ... και την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια ΣΥΝ. αυτό θα, ε, το θέμα θα εγγράφεται στη μέση διατάξη και για τους επόμενους μήνες. Όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροφή, Επιτροπή στις 17 Σεπτεμβρίου εξέδωσε ανακοίνωση βασισμένη στην έκθεση Βιάνο για την συνοχή της πολιτικής της ανάπτυξης όπου ζήτησε μια συνολική προσέγγιση της ε, Ένωσης στην αναπτυξιακή βοήθεια και μια νέα ε, αντίληψη και την αναζήτηση νέων πηγών για την ε, επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια ΣΥΝ. Αυτά πρέπει να αναλυθούν από κάθε σκοπιά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται από την κυρία Φράνσουα Μωρό, που είναι επικεφαλής ε, τμήματος στην Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και επίσης την συνοδεύουν δύο ε, εμπειρογνώμονες, Ανδρέα Μαξιμοβιτς και Νίλς Κάιζερ. που είναι Program Officer του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την ε, διαχείριση ε, των θεμάτων αυτών. Θα ήθελα πρώτα να δώσω το λόγο στον εισηγητή, στην εισηγήτρια μάλλον, την κυρία Κέλλερ, Φραντσίσκα Κέλλερ, για να παρουσιάσει τα βασικά θέματα του ε, κυρίως εγγράφου που αποτελεί, τη βάση της συζητήσεως και μετά θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στους εμπειρογνώμονες. Για 7 λεπτά κυρία ε, Κέλλερ. Ευχαριστώ πολύ και θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Η συνοχή της πολιτικής είναι η συστηματική προώθηση της αμοιβαία εφαρμογής πολιτικών δράσεων μέσα από διάφορες υπηρεσίες και οργανισμούς με συνέργειες ώστε οι στόχοι να μπορούν να επιτευχθούν. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλίζουμε ότι καμιά πολιτική δεν θα αντιβαίνει τον στόχο της ανάπτυξης και σε σχέση με τον κυριότερο στόχο, ο κυριότερος στόχος για την πολιτική αυτή είναι η, η εκρίζωση της φτώχειας. Ωστόσο και πολλοί άλλοι πολιτικοί τομείς πολλές φορές αντιβαίνουν στον κυριότερο αυτό στόχο ε, κρίζωσης της φτώχειας. Έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό το πρόβλημα και είμαστε δεσμευμένοι για να υπάρχει συνοχή και συνεκτικότητα όσον αφορά την πολιτική μας ε, για την ανάπτυξη και λαμβάνοντας υπόψη εντονότερα αυτό το στοιχείο και με, τις ε, εκθέσεις, με την έκθεση ίδιας πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από πρόσφατες ανακοινώσεις της Επιτροπής το ίδιο δείχνει η έκθεση αυτή και η ανακοίνωση είναι ευπρόσδεκτες. Όμως ε, εδώ θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής σε πολλές πλευρές ε, είναι υπερβολικά θετική χωρίς ε, να αναφέρει συγκεκριμένα στοιχεία γενικόλογη και η δέσμευση της Επιτροπής αυτή τη στιγμή δεν ε, ακολουθείτε σε σχέση με κυρώσεις ε, όσον αφορά την πολιτική αυτή και δεν υπάρχει διαδικασία καταχώρησης ε, παραπώνων από πλευράς του πληθυσμού ή όσων εμπλέκονται σε αυτές τις διαδικασίες. Είναι πολύ περιορισμένο αν θέλετε το εύρος του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός για το πώς θα μπορούσε σε μια ευρύτερη περίοδο να ακολουθηθεί μια τέτοια πολιτική πέρα από την θητεία μιας κυβέρνησης. Έτσι λοιπόν θα πρέπει αυτό να θεωρήσουμε ότι είναι ζωτική σημασία για να μπορέσει να επιτευχθεί. Θα ήθελα να τονίσω κάποια παραδείγματα για μη συνεκτικότητα που μπορούν να βρεθούν στην ενέργεια, στην ε, ε, πνευματική ιδιοκτησία, όσον αφορά το εμπόριο επίσης, ε, όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές πολύ λίγα πρόσθετα κονδύλια προβλέπονται για την προσαρμογή και την αντιμετώπιση αυτών των κλιματικών αλλαγών στα αναπτυσσόμενα ε, κράτη. Γίνεται πολύ λίγη, λίγος λόγος ε, για τις ε, χρήσεις γης και την αντιμετώπιση της αποψήλωσης των δασών και τον ανταγωνισμό για την παραγωγή τροφίμων. Αρκετά παραδείγματα δείχνουν ότι η προαγωγή βιοκαυσίμων έχει αρνητικές επιπτώσεις σε σχέση με τις αναπτυσσόμενες χώρες και το περιβάλλον περιβάλλον ε, Και σε σχέση με την παραγωγή της ε, ε, τροφίμων σε σχέση με τον ανταγωνισμό έναντι βιοκαυσίμων, καθώς επίσης βλέπουμε ότι η κατάσταση επιδεινώνεται. Τεράστιες εκτάσεις τροπικών δασών καταστρέφονται για τέτοιου είδους παραγωγές βασίζονται τα περισσότερα προγράμματα σε ορυκτές πηγές ενέργειας και έτσι αυτό δεν είναι το πιο θετικό. Επίσης τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα πρέπει εδώ μεγάλο μέρος να δούμε των εκπομπών ρήπων πώς θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν θεωρηθεί ως μία από τις κυριότερες προτεραιότητες. Τα μέτρα αυτά δείχνουν μία σαφή τάση των συμφερόντων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Οι αναπτυσσόμενες χώρε όχι μόνο δεν έχουν πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες ιατρική και νέα μέσα, αλλά περιορίζονται και από εγγενείς λόγου. Όσον αφορά την αυτάρκεια τροφίμων, η πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν ολέτριες επιπτώσεις ε, στις δομές ε, των αναπτυσσόμενων χωρών. Εξαγωγή κυριότερων γεωργικών προϊόντων ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση καταστρέφουν αγορές στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και έχουμε εδώ από πλευράς διαφορετικών παραγόντων συγκρουσιακή πολιτική με τους κυριότερους αναπτυξιακούς στόχους. Ιδιαίτερα στο εμπόριο που βλέπουμε υψηλό επίπεδο μη συνεκτικότητας στις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης Έχουμε εδώ και, την, ε, και πρότυπα εμπορικών σχέσεων που προάγουν τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων εις βάρος των αναπτυσσόμενων χωρών. Ε, πρόσβαση στις ε, αγορές ε, για τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι περιορισμένη. Έχουμε επίσης και ταχύτητα τους ρυθμούς ε, απελευθέρωσης που επιδεινώνουν την κατάσταση. Δεν έχουμε σαφή αποτίμηση των επιπτώσεων αυτών των πολιτικών από πλευρά μας όσον αφορά την ανάπτυξη. Και δεν αναφέρεται καθόλου στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτό το θέμα, καθώς επίσης είχαν σημειωθεί πολύ σημαντικές επιπτώσεις από αυτό διασυνδέσεις μεταξύ των διαφορετικών στόχων αγνοούνται όσον αφορά τις πολιτικές που ακολουθούνται. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα αντιμετωπίσετε αυτές τις μη συνεκτικές μορφές, τις μη συμβατές μορφές με την ε, ε, συνολική στοχοθέτηση. Είχαν παρουσιαστεί αυτά από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμφωνούμε ότι η αρρωγή δεν είναι επαρκής και πρέπει πρόσθετα κονδύλια και πρόσθετες ε, μέθοδοι να εξευρεθούν βρεθούν για να βοηθηθούν τα αναπτυσσόμενα κράτη. Όμως εδώ βλέπουμε ότι πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε δράση για να επιτευχθεί το ποσοστό που αφιερώνεται στην ανάπτυξη και δεν πρέπει εδώ να υπάρχει στρεβλή εξέλιξη. Επιπρόσθετα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κονδύλια για άλλους στόχους και δεν είναι δυνατόν να ακολουθούν άλλοι πολιτικοί. Ο έλεγχος των κονδυλίων πολλές φορές ε, οι πιο φτωχοί δεν επωφελούνται από τα κονδύλια που διατίθενται. Μπορούμε να ε, ενθαρρύνουμε τέτοιου είδους ε, ροές, όμως δεν υπάρχει διασφάλιση των επιπτώσεων. Ούτε μπορεί κανείς να αποδείξει ότι ο κυριότερος στόχος ήταν πάντα η ανάπτυξη. Και αυτό το θέμα πραγματικά θα πρέπει να συζητηθεί και να μην απουσιάζει και να δούμε κατά πόσον αυτό ε, εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο. Γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ γενικόλογη και αφηρημένη η ε, δράση και πρέπει να υπάρξουν πολλές αποσαφηνήσεις. Αυτό θέλουμε να αποσαφηνιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, πώς είναι δυνατόν να δούμε ότι η πολιτική μας για την ανάπτυξη θα είναι πιο συνεκτική, θα ακολουθεί τους στόχους που έχουμε θέσει ενώπιον μας. Είναι σαφές πώς και με ποια κριτήρια αυτές οι προτεραιότητες επελέγησαν και τι γίνεται σχετικά. Γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω αρκετά πράγματα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω ότι θα μπορέσετε να απαντήσετε στο τέλος αυτές τις ερωτήσεις. Πρώτον, σε σχέση πάλι με αυτές τις πέντε προτεραιότητες, πώς επελέγησαν αυτές οι προτεραιότητες, με ποια κριτήρια και γιατί είναι πέντε αυτές οι προτεραιότητες και πώς οι εμπλεκόμενοι από, τα από τις αναπτυσσόμενες χώρες εμπλέκονται και επιλέγονται σε σχέση με αυτές τις πέντε προτεραιότητες και τι γίνεται με τις άλλες ασυμβατότητες όσο αφορά το, εμπόριο, την γεωργία, την αλληλεία, την γεωργία σε σχέση με αυτές τις πέντε προτεραιότητες. Δεύτερη ερώτηση γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει συμπεριλάβει καμία αναφορά σε σχέση με την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί δεν λάβατε υπόψη τα αποτελέσματα της τελευταίας μας έκθεσης σε σχέση με την πρόσφατη ανακοίνωσή σας και ποια είναι η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα αιτήματα που διατυπώθηκαν από την τελευταία έκθεση. Για παράδειγμα όσον αφορά τα δάση και τις πωλήσει ξυλίας από τα τροπικά δάση. Μετά ποια είναι τα κριτήρια στην ε, πολιτική για την ανάπτυξη ανάπτυξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την επιλογή πολιτικών ε, και την ε, επίπτωση που θα έχουν αυτές οι πολιτικές στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι αναπτυσσόμενες χώρες και τα συμφέροντά τους δεν θα πρέπει να αποκλείονται από τις, ε, την πολιτική για την ανάπτυξη και την αποτίμηση των δράσεών μας. Πώς μπορεί να διασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα διασφαλίζεται μεγαλύτερη συμμετοχή των αναπτυσσόμενων χωρών και η βέλτιστη πολιτική και δείκτες απουσιάζουν. Πώς με μετρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πολιτική για την ανάπτυξη. Βλέπουμε ότι τέτοιοι δείκτες αξιολόγησης της πολιτικής για την ανάπτυξη απουσιάζουν εδώ. Παρότι αναγνωρίζεται η σημασία της πολιτικής για την ανάπτυξη δεν υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα για την, μέσα για την μέτρηση αυτής της πολιτικής. Τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να γίνει για να μπορέσει να υλοποιηθεί η πολιτική για την ανάπτυξη. Και φυσικά η τελευταία ερώτηση αφορά όλους μας ε, που είμαστε σε αυτή την Επιτροπή Ανάπτυξης ε, μακροπρόθεσμο εγχείρημα για μας. Πώς μπορούμε να κατοχυρώσουμε και να βελτιώσουμε την πολιτική ανάπτυξη στην Ευρωβουλή σε σχέση με την Επιτροπή μας ε, και από τις δράσεις της Ευρωβουλής μέσα στο πλαίσιο των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω πολλές ερωτήσεις βλέπουμε ότι είναι πολύ γενικόλογα και αφηρημένα τα όσα αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν είναι σαφές το τι εννοείται με αυτή τη νέα προσέγγιση. Τι γίνεται με αυτή τη ε, νέα αναπτυξιακή πολιτική, ε, ενισχυμένη ε, αναπτυξιακή πολιτική και τι θα συνεισφέρει για την ανάπτυξη. Θα ήμουν ευγνώμων αν απαντούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ. Εξ ονόμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κέλλερ για την ε, πολύ σαφή παρασίαση του θέματος. Πάντως ίσως είναι από την αρχή χρήσιμο να διασαφίσω ότι η ανακοίνωση δεν αποτελεί κανένα είδου σύνοψη της εκθέσεως. Πρόκειται για δύο ξεχωριστά διαφορετικά έγγραφα. Και βέβαια η έκθεση περιλαμβάνει πολύ περισσότερα επί παντός θέματος και επί των θεμάτων που διαλαμβάνονται στο έγγραφο εργασίας της κυρίας Κέλλερ και ασφαλώς τουλάχιστον εν μέρη προσφέρουμε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας. Η ανακοίνωση λοιπόν πρέπει να θεωρηθεί ξεχωριστά από την έκθεση. Η έκθεση όπως και το 271 διαρθρώνεται γύρω από 12 τομείς πολιτικής όπου δραστηριοποιήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και ανέλαβε το 2005 συγκεκριμένες δεσμεύσεις, για παράδειγμα αληθική πολιτική, πολιτική ενέργειας, αγροτική πολιτική, αυτά τα πράγματα ε, συζητούνται στο έγγραφο. Η έκθεση νομίζω ίσω είναι κάπως πιο ισορροπημένη από όσο αφήνει να εννοηθεί η παρουσίαση της κυρίας Κέλλερ. Η έκθεση νομίζω προσπαθεί να προβεί σε μια αξιολόγηση και των θετικών και των αρνητικών πτυχών της πρόοδου ή έλλειψης πρόοδου για τα θέματα αυτά μέσα στην Ένωση. Κάθε ένα από τα κεφάλαια πολιτικής τελειώνει με ένα τμήμα το οποίο εμείς επιγράφουμε ως εκκρεμή θέματα. Είναι δηλαδή τα θέματα εκείνα τα οποία έχουμε εντοπίσει ότι δηλαδή χρειάζονται πολύ περισσότερη δουλειά. Άρα νομίζω ότι είναι ισορροπημένο το εγγραφό μας από την άποψη αυτή. Σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση, αυτή προχωρεί πολύ περισσότερο από την απλή ιδέα, έννοια των 12 τομέων πολιτικής. Και υπάρχουν δύο απλά μηνύματα μετά από πενταετή εμπειρία εργασίας επί της ε, ε, ατζέντα της ECD στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και στο Συμβούλιο και στις χώρες μέλη, αλλά και όπου αυτό είναι δυνατό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε λοιπόν δύο μηνύματα, όπως είπα. Πρώτα, να ληφθεί μια πιο δραστήρια προσέγγιση, proactive. Όταν αντιμετωπίζει κανείς ε, παγκόσμιες προτεραιότητες στην πολιτική ανάπτυξη, πιστεύουμε ότι η Ένωση πρέπει να αναπτύξει μια προσέγγιση πιο προσανατολισμένη στα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, η παγκόσμια ασφάλεια προμήθειας τροφίμων. Αυτό, αυτή δεν ταυτίζεται με την αγροτική πολιτική. Εάν κανείς θέλει λοιπόν, να δραστηριοποιηθεί ενεργητικά μέσα στην διάσταση αυτή που ανέφερα προηγουμένως, σε όλες τις πολιτικές, δηλαδή της Ένωσης κτλ. προς την κατεύθυνση της ασφάλειας τροφίμων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το εμπόριο, η γεωργική πολιτική, ορισμένα θέματα, ορισμένε πολιτικές για το περιβάλλον και το κλίμα, θέματα πολιτικής της ενέργειας και αναφέρομαι εδώ ειδικότερα στα βιολογικά καύσιμα. Άρα, ε, μία από τις παγκόσμιες προκλήσεις δεν ισούτε δεν ταυτίζεται με ένα τομέα πολιτικής. Άρα οι πέντε παγκόσμιες προκλήσεις καλύπτουν ίσως μάλιστα και πολύ περισσότερους τομείς από αυτούς 12 τομείς ε, πολιτικής που ε, εμείς διαλαμβάνουμε στην έκθεση. Δεύτερο βασικό μήνυμα στην ανακοίνωσή μας είναι ότι οι οικονομικές ροές εκτός από την αναπτυξιακή βοήθεια είναι και αυτές σημαντικές για την ανάπτυξη και ίσως και μια φορά και πιο σημαντικές από την ΕΒΑ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον όγκο των κονδυλίων. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εμείς αγνοούμε την ε, ε, οικονομική βοήθεια ανάπτυξης. Ασφαλώς όχι. Αλλά αυτό που λέμε είναι ότι αυτή η βοήθεια, η βοήθεια δεν είναι ευαρκής και ότι πρέπει πράγματι να καταβάλουμε προσπάθειες ώστε να αυξηθούν τα ωφέλη και όλων αυτών των άλλων χρηματοδοτικών ροών, είτε δημοσίων είτε ιδιωτικών, προς και για την ανάπτυξη, είτε σε ένα συγκεκριμένο τομέα πολιτικής, είτε σε κάποιον άλλο. Το ερώτημα είναι πώς αυτές οι ροές που είναι μη ΕΒΑ μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικές. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το κάνουμε με τους μηχανισμούς του PCD που περιλαμβάνουμε εμείς στην έκθεσή μας, κάτι το οποίο λοιπόν μπορούμε να κάνουμε και μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα με αυτά. Παραδείγματα για παράδειγμα στον χώρο της μετανάστευσης όταν προσπαθούμε να λάβουμε κάποια μέτρα, κάποιες πρωτοβουλίες και όταν λέω εμείς εννοούμε εννοώ είτε το ευρωπαϊκό επίπεδο είτε τις χώρες μέλη για παράδειγμα μείωση ε, του κόστου των ε, εμβασμάτων προς τις πατρίδες των μεταναστών. Στον τομέα της ασφάλειας όταν καταβάλουμε προσπάθειες να κάνουμε παρεμβάσεις στην ασφάλεια είτε μη στρατιωτικού είτε στρατιωτικού χαρακτήρα και που να είναι πιο συμβατές με τους στόχους της ανάπτυξης, πάλι βελτιώνουμε τα αποτελέσματα υπέρ της ανάπτυξης. Αυτό εννοούμε όταν λέμε ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλοι οι μοχλοί των μηχανισμών που προσφέρονται ώστε να αυξηθεί το αποτέλεσμα. Η χρηματοδότηση για το κεφάλαιο βεβαίω είναι άλλο σημαντικό τομέα όπου πρέπει να εξασφαλιστεί η συνοχή με την ανάπτυξη και αυτό πρέπει να αποτελέσει και πολιτική προτεραιότητα. Οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωσή μας προέρχονται ευθέως από τις αξιολογήσει που έχουμε κάνει στην εκθεσή μας το 2007 για το PCD και η άλλη πιο πρόσφατη του περασμένου Σεπτεμβρίου. Βοήθεια και δάνεια δεν αρκούν. Αυτό ε, λέμε ως πρώτο συμπέρασμα και νομίζω ότι και στο έγγραφο εργασία σας το αναγνωρίζετε. Πολιτικές άλλες εκτός της πολιτικής ανάπτυξης παίζουν σημαντικό ρόλο για την ενίσχυση των, της πρόοδου των αναπτυσσόμενων χωρών. Αλλά η PCD υπό την έννοια αυτή δεν μπορεί παρά να είναι μια συμπλήρωση της αναπτυξιακής βοήθειας. Δεν πρόκειται να αντικαταστήσει την ε, ΕΒΑ, την ε, βοήθεια ανάπτυξης. Και αυτά μεταξύ των δύο ανακοινώσεων 2005-2009. Δεύτερον, η BCD είναι δύσκολη διαδικασία, περίπλοκη, η οποία ε, απαιτεί τη συμμετοχή πολλών φορέων, θεσμικών φορέων, αλλά και πέρα των θεσμικών φορέων και ιδιωτικών φορέων και της ε, οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Και είναι ανάγκη αυτή η έννοια να χρησιμοποιηθεί με πιο αποτελεσματικό τρόπο και με πιο ενεργό τρόπο. Και γι' αυτό κάναμε την πρόταση για την επόμενη διετία, τριετία να αναπτύξουμε ένα πραγματικό πρόγραμμα εργασιών που δεν είχαμε μέχρι τώρα, όπου να μπορούμε να λαμβάνουμε πρωτοβουλίες για την άσκηση πολιτικών για να βοηθηθεί να ενισχυθεί η PCT. Αυτό είναι το νόημα των ε, βασικών αυτών μηνυμάτων της ανακοίνωσής μας. Now, Όπως προανέφερα, η ανακοίνωση δεν είναι καθόλου μια περίληψη της έκθεσης. Τώρα και σε σχέση με τις ε, αναφορές ε, τομεακά, σε σχέση με το εμπόριο για την έκθεση 20 σελίδες αφιερώνονται στο εμπόριο στην έκθεση όπου αναφέρουμε την πρόοδο ή έλλειψη προόδου σε σχέση με την επίτευξη των στόχων όπου αναλύουμε τις διαβουλεύσεις και τις διαπραγματεύσεις όπου συζητούμε τον ρόλο της βοήθειας που μπορεί να συνεπάγεται το εμπόριο για την ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες ευκαιρίες εμπορικές κτλ. όπου συζητούμε την περιφερειακή ολοκλήρωση και τις συνιστώσει του εμπορίου όσον αφορά την γεωργική πολιτική. Όσον αφορά τι πρώτε ύλε, αυτό είναι ένας νέος τομέας εργασίας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καθώς γνωρίζετε έχει προσαρμόσει την, σε σχέση με την ανακοίνωση νωρίτερα εφέτος αυτά τα θέματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε και μια ομάδα επαϊόντων που θα διασφαλίζει ότι η συνιστόσα της ανάπτυξης θα αναφέρεται και θα λαμβάνετε υπόψη θέματα που σύντομα αναφέρονται σε σχέση με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να δούμε πώς μπορούμε να ταυτοποιήσουμε και να εντοπίσουμε και να συμφωνήσουμε σε ένα σύνολο μέτρων δράσεων για να βελτιωθεί η διαχείριση και διακυβέρνηση όσον αφορά την αναπτυξική πολιτική. Και στο τέλος νομίζω για την αλληλεία η έκθεση δίνει κάποιες απαντήσεις στα, στα ερωτήματα που διατυπώσατε. Υπάρχουν εδώ θέματα κλειδιά και σίγουρα θα συνεχίσουμε να προσέχουμε αυτά τα θέματα στην ανάπτυξη των δράσεών μας. Κάθε μία από τις πολιτικές αλληλείας και τις συμβάσεις, ε, συμφωνίες αλληλείας ε, εξετάζεται και όλα αυτά θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται ως μέσα και ως μηχανισμοί, εργαλεία για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την αναπτυξιακή πολιτική αλλά η αλληλεία και έδωσα το παράδειγμα της ε, επάρκειας και ασφάλειας τροφίμων για να αναφέρω ότι είναι μια κύρια προτεραιότητα το, σε σχέση με το θέμα αυτό δεν θα εξετάζουμε μόνο μια πολιτική αποκλειστικά η αλληλεία για τις χώρες αυτές που αναφέρουμε έχει θεμελιώδη ρόλο όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας τροφίμων και αυτό το λέω για να αναφέρω ότι τα θέματα πολιτικών που θα εξετάσουμε για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων, τα θέματα αυτά είναι πολύ ευρύτερα σε φάσμα. Όσον αφορά την παράνομη ε, ξύλευση, την παράνομη αποψήλωση δασών ε, και η ε, πώληση τροπικής ξυλίας και τα θέματα των εκπομπών ρήπων, όλα αυτά στην έκθεσή μας αφορούν και τη συνιστόσα των ενεργειακών θεμάτων και το περιβάλλον και φυσικά η ξυλία θα συνεχίσει να έχει υψηλή προτεραιότητα στην ημερήσια διαταξή μας. Τώρα, για την χρηματοδότηση χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση δεν ήταν ένας από τους τομείς ε, των 12 πολιτικών όπου συνολικά ανέλαβε το 2005 υποχρεώσεις για την πολιτική για την ανάπτυξη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά είναι μια υποεξέλιξη αυτή η μερίσια διάταξη, ενρευστό και γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι το θέμα της, ε, της καταπολέμησης ε, των παράνομων ροών κεφαλαίων, της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και των φορολογικών οάσεων για να μπορεί να διασφαλιστεί ότι από τέτοια δράση θα απορρέουν περισσότερα ωφέλη. Εξετάζουμε την εξέλιξη και ανάπτυξη των πολιτικών μας και των προτάσεών μας που θα διατυπωθούν ε, νωρίς το 2010 κατά το τέλος ε, του πρώτου τριμήνου το 2010 πιθανότατα και αποτελεί μέρος ε, του σχεδίου του προγράμματός μας ε, για τις εργασίες μας. Για τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας τους επιλέξαμε αυτά τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας τους ως ένα θέμα ενδυνάμει σημαντικό για την πολιτική ανάπτυξη. Αυτό σίγουρα είναι ένα από τα θέματα κλειδιά για την προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας και της μετάθεσης μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. Επίσης έχουν τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τη σημασία τους για τα θέματα των κλιματικών αλλαγών και για την ασφάλεια τροφίμων και ε, διασφάλιση επάρκειας. Και ενώ έχουμε αναλάβει ήδη κάποιες προσπάθειες ε, για να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τους αναπτυξιακούς στόχους σε σχέση με συμφωνίες TRIPS για παράδειγμα, είμαστε πισμένοι ότι πολλά περισσότερα θα μπορούσαν να γίνουν, πολλά περισσότερα για να βελτιωθούν οι τρόποι και οι μέθοδοι με, τις με, ε, της, ε, τη δυνατότητα βελτίωσης ε, της απόδοσής μας. Αυτά έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη για ένα ευρύτερο φάσμα πολιτικών. Για τις κλιματικές αλλαγές είναι μια κύρια πολιτική προτεραιότητα και όπως ε, αναφέρθηκε πιο πριν η συνεκτικότητα και η συνοχή με τους στόχους ανάπτυξης πρέπει να έχει ύψιστη προτεραιότητα στο μέλλον. Υπάρχουν πολλά τα οποία εν δυνάμει μπορούν να καλυφθούν, βιοκαύσιμα για παράδειγμα αναφέρατε πολλά άλλα θέματα σε σχέση με τις κλιματικές αλλαγές και την ανάπτυξη που θα μπορούσαν να καλυφθούν και που πιστεύουμε ότι πρέπει να τύχουν υψηλή προτεραιότητα. Συνοψίζοντας, η πρόθεσή μας σίγουρα δεν ήταν να στενέψουμε, τον, να περιορίσουμε τον αριθμό πολιτικών ή το φάσμα πολιτικών σε σχέση με την ανάπτυξη. Πρώτα απ' όλα οι δεσμεύσει για τη στοχοθέτηση και για την πολιτική μα παραμένουν οι δεσμεύσει αυτέ. Παραμένουν σημεία αναφορά την στοχοθέτησή μας μέσα στο πολιτικό αυτό έγγραφό μας. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να είμαστε πιο δραστήριοι και αποτελεσματικοί στις δράσεις μας. Όχι μόνο ακολουθώντας κάποιες πρωτοβουλίες από πλευράς άλλων τομέων και βλέποντας πώς μπορεί να επιτευχθεί η ανάπτυξη, αλλά και αναλαμβάνοντας αμεσότερα πρωτοβουλίες και δράση που θα έχουν και θα καλύπτουν μια ε, σημαντική συνιστόσα για την ανάπτυξη. Το να καταστεί αυτό το έργο για την πολιτική ανάπτυξη πιο πολιτικό στον χαρακτήρα του είναι ακαθόδες και δύσκολο. Αυτό σημαίνει να εργάζεται κανείς πάντα στα περιθώρια των δυνατοτήτων, των οικονομικών δυνατοτήτων για την ανάπτυξη. Διότι ε, κανονικά εστιαζόμαστε, εστιάζονται όλοι σε ε, άλλους στόχους. Εργαζόμαστε λοιπόν ε, στο περιθώριο και τα άκρα της ημερησίας διάταξης ε, διότι οι ε, ε, στόχοι σε σχέση με τους στόχους της χιλιετίας δεν είναι πάντα οι ίδιοι και δεν είναι πάντα μόνο αναπτυξιακοί και λοιπόν πρέπει με τη βάση αυτή και την εμπειρία μας να δούμε και ένα εύρος χρόνου μεγαλύτερο από την πενταετία και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, να είμαστε σε ένα υψηλότερο, ανώτερο επίπεδο πολιτικής εμπλοκής ε, στις δράσεις που θα ακολουθούμε για την ανάπτυξη. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να εργαστούμε σε θέματα που θα έχουν υψηλή πολιτική προτεραιότητα από πλευρά των κρατών μελών και των ε, θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, αναφερόμενοι σε σχέση με τα δύο σημεία τα οποία έχετε παρέμβει, είχατε ένα τέταρτο και έχετε νομίζω καλύψει αυτόν τον χρόνο. Ευχαριστώ. Τώρα έχετε εσείς τον λόγο για 10 λεπτά παρακαλώ. Yeah, okay. Thank you very much. Um, Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ που είμαστε εδώ και που μας δίνετε την δυνατότητα να παρουσιάσουμε την αντιέκθεση, αντέκθεσή μας ε, όσον αφορά την ε, ε, πολιτική προσπάθεια. Υποβάλλουμε αυτή την έκθεση αλλά και θα εξετάσουμε και κάποιες πτυχές της ανακοίνωσης διότι θεωρούμε ότι είναι σημαντικά αυτά τα θέματα για εκείνους που δεν γνωρίζουν, η Concord είναι η ε, ένωση ε, των δραστηριοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε 18 πλατφόρμες, 1.600 ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Όλες αυτές υποστηρίζουν από εκατομμύρια πολίτες πανευρωπαϊκά έχουμε κύριο, κυριότερο προβληματισμό και δράσεις από πλευρά των κρατών μελών και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών συμπεριλαμβάνοντας και την αναβάθμιση της ποιότητας του αναπτυξιακού έργου. Πιστεύουμε ότι η σωστή προσέγγιση και η ένταξη των γυναικών στο, στην αναπτυξιακή προσπάθεια και των δικαιωμάτων των γυναικών έχει τεράστια σημασία. Και η επόμενη αυτή διαφάνεια θέλει να το υπογραμμίσει αυτό και να το καταστήσει ανάγκη. Και Πολλοί από εσά γνωρίζουν βέβαια την ε, οργάνωσή μας, άλλοι όμως όχι. Και γι' αυτό θα ήθελα σύντομα να κάνω λόγο για αυτή την έκθεση την οποία συντάξαμε για να προαγάγουμε την πολιτική συνοχής και συνεκτικότητα στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε σχέση με αυτά έχω κάποια θέματα που θέλω να αναφέρω. Δεν είναι πάντα πολύ εύκολο να εγγραφούν αυτά τα θέματα στην ημερησία διάταξη και εμεί θέλουμε να αντιδράσουμε σε σχέση με την έκθεση αυτή και να προτείνουμε στι συστάσει μα κάποια πράγματα. Και να αναφέρουμε και κάποιε σημαντικέ ασυμβατότητε. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να πούμε γιατί είναι σημαντική η αναπτυξιακή προσπάθεια. Μέχρι ότου θα έχουν καθοριστεί όλα τα άλλα θέματα και θα έχουν ρυθμιστεί μέσα στο πλαίσιο τη πολιτική για την ανάπτυξη, καθώ επίση και τα άλλα θέματα, κατά πολέμηση φορολογικών οάσεων και η βοήθεια προ τι αναπτυσσόμενε χώρε θα είναι στο να δίνει κανεί να ρίχνει χρήματα σε ένα πίθο των Δαναίδων. Και πρέπει να δούμε ότι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα δίνονται αυτά τα χρήματα και θα γίνονται αυτέ οι δράσει πρέπει να είναι ε, καλά ρυθμισμένο και να αποφεύγεται αυτή η ε, ε, κονδυλίων. Και υπάρχουν πολλά θέματα, τα ίδια ερωτήματα τα οποία εμείς οι ίδιοι ρωτούσαμε και θέταμε επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Φυσικά δεν καταλήγουμε όλοι στα ίδια συμπεράσματα, διότι εμείς δεν θεωρούμε ότι η βοήθεια για την ανάπτυξη πρέπει να καταργηθεί, αλλά πρέπει το σύστημα να καταστεί εύρυθμο μέσα στο οποίο η βοήθεια αυτή λειτουργεί. Ένας τρίτος λόγος ε, για τον οποίο είναι σημαντικό αυτό, αν η οικονομική κρίση μας έμαθε κάτι, έδειξε τις ελλείψεις ενός προτύπου για ανάπτυξη χωρίς να λαμβάνεται καθόλου υπόψη ε, ο μηχανισμός ανακατανομής πλούτου. Δηλαδή τα κοινωνικά δικαιώματα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα κοινωνικά θέματα τα οποία πρέπει να καλύπτονται. Ένας τελευταίο λόγος για τον οποίο είναι σημαντική η πολιτική για την ανάπτυξη είναι επειδή εμεί ε, θέλουμε αυτό που οι φίλοι μα ε, θέλουμε να πετύχουν στι αναπτυσσόμενε χώρε, Να μην εξαρτώνται πλέον από την βοήθεια, να πάρουν τη μοίρα του και το πεπρωμένο του στα χέρια του να καταστούν αυτάρκη και ανεξάρτητα. Μία από τι προτάσει μα σε σχέση με την ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια και πιστεύουμε ότι η συνοχή και συνεκτικότητα είναι να διασφαλίζουμε ότι οι εξωτερικέ δράσει τη ε, Ένωση δεν, δεν θα αντιβαίνουν και δεν θα τορπιλίζουν του κυριότερου στόχου. Πιστεύουμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία μια ε, συνολική προοπτική είναι σημαντική διότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι αποδέκτες πρέπει να είναι οι κριτές αν η πολιτική που δίνουμε για την ανάπτυξη έχει αποτέλεσματα ή όχι. Εκείνοι θα πρέπει να κρίνουν. Θα πρέπει να διατυπωθούν τα ερωτήματα ώστε να μετρηθούν τα αποτελέσματα. Αποτελέσματα βάσει επιδόσεων. Θέλουμε να δούμε αποτιμήσεις βάσει αποτελεσμάτων. Ε, πιστεύουμε στη σωστή ε, ε, εύρυθμη προσέγγιση. Όταν έχουμε δεσμεύσεις πρέπει να είμαστε συνεπείς συνεπεί και να υλοποιούμε αυτέ τι δεσμεύσει ε, και τι υποσχέσει μα. Πρέπει να δούμε επίση τι συνδεδεμένε αλληλεξαρτώμενε πτυχέ αυτών των δράσεων. Δεν είναι μόνο η, η εξέταση τη ανάπτυξη και του εμπορίου ή τη ε, ανάπτυξη και τη μετανάστευση, αλλά πρέπει να δούμε το τρίγωνο αυτό εμπόριο, ανάπτυξη και μετανάστευση. Και πρέπει αρκετά νέα θέματα, παρότι δεν είναι νέα, απόλυτα καινούρια. Για παράδειγμα, τα θέματα ε, φοροδιαφυγής ε, και ε, τα θέματα καταπολέμησης φορολογικών οάσεων είναι καινούρια υπό αυτό το πρίσμα επειδή πρέπει να ενταχθούν σε ένα σφαιρικότερο πλέσμα. Τι έχουμε στην εκθεσή μας. Εντοπίζουμε τρεις λόγους για την απουσία προόδου στην ε, πολιτική ανάπτυξη και υποβάλλουμε συστάσεις πώς μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα πιστεύουμε ότι η, αναπτυξή, η αναπτυξιακή στόχη ήταν ε, ε, επουσιοδέστερη όσον αφορά άλλες προτεραιότητες. Πολλές φορές πιστεύουμε ότι λάθος προτεραιότητες ε, τίθενται και εδώ πολλές φορές ε, υπάρχει και το θέμα πολιτικών που ακολουθούνται που δεν είναι οι ορθότερες. Είναι ένα παράδειγμα πολιτικής ε, που θέτει λανθασμένες προτεραιότητες όχι μόνο για την ανάπτυξη αλλά επίσης και για την ευημερία των ίδιων των Ευρωπαίων πολιτών που εμπλέκεται άμεσα. Πιστεύουμε εδώ λοιπόν ότι η διασύνδεση, η αλληλεξάρτηση είναι σημαντική. Βλέπουμε αυτή την αλληλεξάρτηση και την αλληλοδιασύνδεση μεταξύ πέντε πολιτικών ανάπτυξης. κλιματικέ μεταβολέ, εμπόριο, γεωργία, μετανάστευση καθώ επίση και οικονομία και οικονομικές σχέσεις. Προτού κανείς πει, α, επιλέξατε πέντε ε, ε κατηγορίες, πέντε άξονες ε, και αυτό λόγω ε, ε απουσίας κονδυλίων διαφορετικά θα είχατε επιλέξει περισσότερους. Πρέπει να δούμε την αλληλοδιασύνδεση. Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Σουηδία. Επίσης, σας ζητώ να εξετάσετε αυτή την έκθεση. Θέλω να τονίσω όμως και να υπογραμμίσω κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, κάποια αριθμητικά μεγέθη και στοιχεία. 200 εκατομμύρια εκατομμύρια. Θα έχουμε εκατομμύρια περιβαλλοντικούς μετανάστες ε, και παρόλα αυτά από πλευράς των ε, ευρωπαϊκών πολιτικών ακολουθούμε μια πολιτική αναχέτησης. Εκείνοι όμως που φεύγουν από τις χώρες τους λόγω των κλιματικών ε, μεταβολών θα συνεχίσουν να έρχονται στις χώρες μας. Για το 2006 το Καμερούν σταμάτησε να εισάγει, να, να εισάγει κατεψυγμένα κοτόπουλα. κάθε φορά βλέπουμε ότι η εισαγωγή παραγωγή αυτή εξαφανίζει θέσεις απασχόλησης ε, και στην ε, μεταποίηση αλλά και στη συσκευασία. Τι έκανε λοιπόν το Καμερούν, απέκλεισε το κρέας των πουλερικών ε, σε σχέση με τις εμπορικές αυτές εισαγωγές. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση στις διαπραγματεύσεις που κάνει επιμένει και λέει ότι θα πρέπει να ισχύσουν αυτές οι εισαγωγές για το Καμερούν. Το Καμερούν δεν θα μπορέσει όμως να επομιστεί αυτή την υποχρέωση. Και το δράμα το οποίο βλέπουμε σε σχέση με τα γαλακτοκομικά ατομικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανένα δεν λέει ότι δεν έχει δικαίωμα να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το οποίο έκανε, άσχετα αν αυτό είναι το σωστό ή όχι. Πρέπει να δούμε όμω, ε, να βρούμε τρόπου ε, να μην είναι η, υπο... η πολιτική μα αντιπαραγωγική και υποκριτική. Για παράδειγμα, σε σχέση με τα βιοκαύσιμα, για παράδειγμα, σε σχέση με τι στρεματικέ αποδόσει ε, στην Τανζανία και σε άλλε χώρε, πολλοί εγκαταλείπουν τι καλλιέργειέ του για να καλλιεργήσουν καλλιεργηθούν βιοκαύσιμα. Έτσι κινδυνεύει η παραγωγή τροφίμων λόγω της παραγωγής βιοκαυσίμων και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό. Επίσης γνωρίζουμε ότι υπάρχουν παράνομες ροές 1-3 εκατομμύριο ευρώ σε σχέση με τις αναπτυσσόμενες χώρες που καθιστούν τα 50 δις τα οποία διαθέτουμε εμείς για την αναπτυξιακή μας πολιτική μια σταγόνα μόνο στον ωκεανό καθώς επίσης και για το αν θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συντάσει τον δικό της κατάλογο. Ναι, θα έπρεπε να συντάσει τον δικό της κατάλογο και να ζητήσει από τα ίδια της τα κράτη-μέλη να αναλάβουν δράση και να διασφαλίσουν ότι η οδηγία για τη διαφάνεια που έχει ε, υιοθετηθεί θα εφαρμοστεί και θα έχει τις αναγκαίες επιπτώσεις. Αναφέραμε σε σχέση και με τα μείζωνα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, ε, ονόματι της ανάπτυξης. Όλα αυτά είναι είναι αναδυόμενα θέματα τα οποία θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και να προσέχουμε. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει και εδώ ε, σε σχέση με τις προτάσεις που πρέπει να διατυπώσουμε στην έκθεση στη σελίδα 7 υπάρχουν ε, πολυάριθμες προτάσεις. Εμείς ε, συμφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να υπάρξει μια συντονισμένη προσπάθεια για να πάνε τα πράγματα σωστά. Αλλά πρώτα απ' όλα μπορούμε να τα κάνουμε τα πράγματα μόνο εμένοντας και επιμένοντας στις σωστές δράσεις. Να διασφαλίσουμε ότι οι μηχανισμοί και τα μέσα που έχουμε τώρα θα εφαρμόζονται σωστά. Να δούμε για παράδειγμα τι γίνεται σε σχέση με μια γενική διεύθυνση, να δούμε τι τελευταίε συστάσει αυτή τη ίδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή ω προ αυτά τα θέματα. Πρέπει να είναι δεσμευτικέ ε, οι υποχρεώσει μα, οι δεσμεύσει μα. Αν κανεί ε, δεν ε, τι λαμβάνει υπόψη όταν έρχεται η ώρα να εφαρμοστούν οι πολιτικέ, τότε είναι περιττό να εξετάζονται. Πρέπει να έχουμε ένα μηχανισμό καταχώρηση παραπώνων. Και σε σχέση με, την, με έναν ombudsman, με έναν συνήγορο του πολίτη για τέτοιου είδους παράπονα. Και στο τέλος τέλος όλες αυτές οι αποτιμήσεις πρέπει να βασίζονται σε αξιόπιστα τεκμήρια και στοιχεία. Ένας τρόπος με τον οποίο αυτή η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανάπτυξης θα μπορούσε να βοηθήσει είναι η διεξαγωγή ακροάσεων. Από με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Επιτροπή ε, Παγκοσμίου Εμπορίου είναι κάτι το οποίο μπορούμε να εξετάσουμε στη συνέχεια. Και μια συνολική πανευρωπαϊκή προσέγγιση. Στην ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εργάζεται για την πολιτική ανάπτυξη σαν ένα τμήμα του συνόλου των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προάγονται πολιτικές που θα είναι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα σε αυτές θα εντάσσεται και η πολιτική την ανάπτυξη. Εδώ έχουμε και κάποιες ε, ε, παρατηρήσεις να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, εμείς ε, θεωρούμε ότι ίσως θα πρέπει να εργαζόμαστε πιο αποτελεσματικά και πιο έντονα. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει σε σχέση με την ολιστική προσέγγιση, συνολική σφαιρική προσέγγιση. Εμείς ως ε, αρμόδιοι για τα θέματα ανάπτυξης ε, ανησυχούμε για την ε, παρέκκληση της προσοχής από θέματα ανάπτυξης και στρέβλωση των πολιτικών που θα ακολουθηθούν. Ακόμα και όταν για παράδειγμα η αλληλοσυνάρτηση όλων αυτών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων στην ανακοίνωση αναφέρονται μόνο οι θετικές πτυχές και ξέρουμε όμως ότι αυτή τη στιγμή η Κίνα και η Ινδία προσφεύγουν εις βάρος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ΠΟΕ για την πρόσβαση σε, ιατρικά, σε ιατρικά σκευάσματα, σε φάρμακα κτλ. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Απλά και μόνο σε σχέση με την ε, ε, διοχέτευση κονδυλίων δεν είναι α, πάντα επαρκής. Διατυπώνω την, την εξής προέρχεται όλη αυτή η προσέγγιση. Από την Γενική ε, Σύνοδο που προερχεται ολη προαχθεί από την γενικη συνοδο που ειχε προαχθει απο την ιταλια για μια προσέγγιση αναχώρα. Και αναφέρεται και στα συμπεράσματα του 2009 στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποστήριξη προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η αναπτυξιακή πολιτική, ενισχυμένη αναπτυξιακή πολιτική είναι κάτι καινούργιο από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνεται λόγος για κάποια νέα θέματα, για την χρήση των ε, κονδυλίων για να μπορέσει να υπάρξει μοχλικό αποτέλεσμα. Επιτρέψτε μου πολύ σύντομα να πω γιατί ανησυχούμε για αυτήν την πρόταση. Πρώτα απ' όλα θεωρούμε ότι δίνει το απόλυτα λαθασμένο ε, μήνυμα την πιο λάθος χρονική στιγμή σε σχέση με τις, ε, το ΦΑΟ για παράδειγμα γνωρίζουμε ότι μειώνονται τα κονδύλια, μειώνονται οι δράσεις ε, και η ανάπτυξη μειώνεται και συρρυκνώνεται. Ξέρουμε ότι η αναπτυξιακή υποστήριξη είναι το μόνο το οποίο μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους οι αναπτυσσόμενες χώρες. Ξέρουμε ότι είναι η μόνη προβλέψιμη χώρα ε, πηγή βοήθειας και εσόδων για αυτές τις χώρες. Θέλουμε λοιπόν να πούμε ότι η ενισχυμένη αυτή ε, πολιτική που μας ε, παρεκκλίνει από την ε, πολιτική ανάπτυξη είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Επίσης σε σχέση με τη συζήτηση που είχε γίνει είχαμε ανταλλαγή απόψε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολλές φορές προσπάθησαν να μας καθησυχάσουν και να μας πούν θα τηρήσουμε, θα τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας και θα είμαστε συνεπείς προς τις υποχρεώσεις αυτές. Αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Όταν μου λέει κάποιος εμένα δεν ξέρω για σας ότι θα είμαστε ρεαλιστές όμως αυτό με κάνει να ανησυχώ. Και για όσου από εσά δεν έχουν προσέξει και δεν έχουν διαβάσει αυτή την ανακοίνωση όπως πολλοί από εμά, θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε μια πρόταση που λέει θα χρησιμοποιήσουμε την προσέγγιση ODA Plus για τις συζητήσεις και αναθεώρηση των πολιτικών μας, ιδιαίτερα την δομή της εξωτερικής, των εξωτερικών μας δαπανών. Αυτή είναι η μία και μόνη πρόταση που μας δημιουργεί τις μεγαλύτερες ανησυχίες και τίθεται στο τέλος του κεφαλαίου με τελείως θα έλεγα αυλαβή τρόπο. Θα μπορούσε κανείς ε, να το διαβάσει ίσως και να το ερμηνεύσει και με θετικό τρόπο. Όμως αυτή είναι μία μόνη πρόταση που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ εκεί που έχει τοποθετηθεί. Επίσης πιστεύουμε ότι αυτό μας οδηγεί στην, ε, ε, στο ερώτημα της πολιτικής μορφής της βοήθειας και για το μέλλον η αρχιτεκτονική που θα υιοθετηθεί για αυτό το σκοπό και που δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια θα είναι ενέχει τον κίνδυνο να υπάρχει παρέκκληση από την αρχική στοχοθέτηση για την ανάπτυξη. Και εδώ ουσιαστικά διαφορετικές ερμηνείες υπάρχουν και θα μπορούσαν να υπάρξουν για την Ένωση και για την ODA+. Plus, ODA Θέλουμε να ανοίξουμε αυτό το κυβότιο της, το κουτί της Πανδώρας, ξεκινώντας έτσι μια τέτοια συζήτηση για, την, ε, για τις δεσμεύσεις για την ανάπτυξη. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω λέγοντας ότι κατανοούμε το πολιτικό πλαίσιο και την πολιτική συγκυρία. Ξέρουμε ότι δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια συνάντηση με τον Ντέβιντο Σάλιβαν από την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και σε σχέση με την απουσία του εμπορίου στην ανακοίνωση είπε ότι αυτό ήθιστε και πολλές φορές συμβαίνει. Δηλαδή έχει συναντήσει και αυτό δεν είναι ο τρόπο με τον οποίο εμεί θα θέλαμε να καλυφθούν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι εύκολο πράγμα το θέμα τη ανάπτυξη. Επίση, αντιλαμβανόμαστε ότι το ODA έχει υποστεί επικρίσεις. Θέλουμε όμω να διασφαλίσουμε θα υπάρξει πολιτική υποστήριξη για την ανάπτυξη και πολιτική υποστήριξη για το εμπόριο. Και το Ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι είναι δεσμευμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση για το εμπόριο και την ανάπτυξη. Εδώ θα πρέπει να πιέσουμε τι κυβερνήσει μας λοιπόν για να υπομισθούν τις υποχρεώσεις τους και να είναι συνεπεί προς αυτές. Ευχαριστώ. The floor is for Mr. Kaiser. Κύριε Κάιζερ, 10 λεπτά. Α, να συνεχίσω εγώ τότε. Εξ ονόματος της οργάνωσής μου, πρώτα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κυρία Πρόεδρε και ίσως μπορώ να συμπληρώσω τις παρουσιάσεις που έγιναν ήδη. Αν θέλετε μπορείτε να βλέπετε τις διαφάνειες ε, στην οθόνη εργάζομαι για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης, ε, ε, Πολιτικών Ανάπτυξης και ο στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των απολυπτριών χωρών. Θα σας παρουσιάσω τέσσερα πράγματα. Την έρευνα που κάνουμε, ορισμένες από τις δυσκολίες ανακρούεται ένας εθνικός ύμνος αλλά δεν ξέρουμε από πού είναι. Το τηλέφωνο του κ. Μαρτίνες. Η πρόοδος που έχει γίνει μέχρι τώρα για την ε, πρόθεση της PCT την προηγούμενη εβδομάδα έλαβα ένα σχέδιο των, ε, ε, των συμπερασμάτων για την επόμενη Δευτέρα, για το, το Συμβουλίο δηλαδή, και ε, συμμεριζόμαστε ορισμένα πράγματα. Τέλος, τι έχει κάνει το κοινοβούλιο για να προωθήσει την PCD. Από την 1η Δεκεμβρίου και μετά θα ενισχυθεί η νομική μας βάση για την πρόθεση της PCD στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την μείωση της ε, φτώχειας που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πλέον το στοιχείο αυτό σε όλους τους τομείς πολιτικής και η αξιολογή της αποτελεσματικότητας είναι δύσκολη βέβαια διότι δεν υπάρχουν ε, συγκεκριμένοι στόχοι δεν ξέρουμε δηλαδή αν θα κρίνεται ότι το μπουκάλι είναι μισογεμάτο ή μισοάδιο αν είναι το σωστό ε, μπουκάλι τι υγρό περιέχει και το καθεξής το μόνο που ξέρουμε είναι ότι έχουμε την υποχρέωση, έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να κάνουμε μια προσπάθεια και ότι στη βάση αυτή μπορούν να εκφραστούν διάφορες γνώμες για το αν είναι επιτυχημένες οι προσπάθειες αυτές, ή αν είναι ανεπαρκείς, αν είναι αρκετά συνεκτικές ή ε, πολιτικές. Και αυτό καθιστά δύσκολο, δύσκολη και την έρευνα στον τομέα αυτό. Και δεν ξέρουμε και τι σημαίνει ακριβώς η επαρκής απόδοση. Έχουμε κάνει δύο αξιολογήσεις στο παρελθόν. Πρώτον για να εξετάσουμε ποιοι μηχανισμοί έχουν υιοθετηθεί από τις χώρες μέλη για να προωθηθεί η PCD αλλά και το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν. Δεύτερο, πρόσφατα κάναμε κάποια έρευνα που εξέτασε τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών πολιτικών στην πείνα και στην φτώχεια στον κόσμο και θα περιληφθούν στην φετινή έκθεση της EUPCD και στην τελευταία αυτή μελέτη διαπιστώσαμε ότι είναι δύσκολο να εξηγήσουμε στον κόσμο στις αναπτυσσόμενες χώρες τι ακριβώς εννοούμε όταν μιλούμε για τους στόχους ε, αυτή είναι σαφής δεν αντιλαμβάνονται όμως ε, τα περί νομικής βάσης και τις σχετικές ε, με την πολιτική αυτή συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δύσκολο είναι επίσης όταν διεξάγεται έρευνα να διαπιστωθεί κάποιο αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση της φτώχειας από τις ευρωπαϊκές προσπάθειες, γιατί αυτές συνήθως εντάσσονται μέσα στις διεθνείς Τώρα, οι γιατροί από τη Ζάμπια έρχονται να εργαστούν στην Ευρώπη επειδή ε, αυτό αποτελεί το αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών πολιτικών ή επειδή πρέπει να περιμένουν δύο χρόνια εκεί για να ε, προσληφθούν. Τέλος πάντων, ε, πρέπει να παίξουν ένα ρόλο και οι αναπτυσσόμενες χώρες στις μελέτες αυτές. Στο έργο μας βρήκαμε ότι μπορούμε να μιλήσουμε για τριών ειδών μηχανισμούς, για ρητές δηλώσεις πολιτικής για μηχανισμού συντονισμού για δυνατότητες ε, συνάντησης όπως ε, Inter-Service Communication ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις σχέσεις με την PCD, τις αλληλονημερώσεις σε παλαιότερη αξιολόγηση που χρηματοδοτήθηκε από διάφορε χώρε μέλη, είδαμε ότι οι προσπάθειες αυτές παραμένουν ακόμα στο πειραματικό επίπεδο και είναι ανώριμες. Ορισμένες επίσης από τις πολιτικές δεσμεύσεις που έχουν αληφθεί είναι αμφισβητήσιμες και ορισμένες από τις κυβερνήσεις των χωρών μελών δεν αντιλαμβάνονται τι είδους προσπάθεια απαιτείται για να προωθηθεί επατεραισματικά η PCD. Αρκούν για παράδειγμα τέσσερα άτομα σε ένα Υπουργείο Εξωτερικών που να ασχολούνται με τα θέματα αυτά όταν έχουν 12 τομείς για να εργαστούν. Επομένω, ένα δημόσιο υπάλληλο ανά τέσσερι τομεί. Ορισμένε χώρε μέλη δεν έχουν καν αναπτύξει μια ξεκάθαρη πολιτική για την PCD. Υπάρχουν λοιπόν πολλέ ε, και μεγάλε διαφορέ απόδοση των προσπαθειών αυτών και μέσα στι χώρε μέλη. Πώ να εξασφαλιστεί τώρα η συμμετοχή πλέον παραγόντων στι προσπάθειε αυτέ. Συχνά ένα μηχανισμό PCD θεωρείται ότι αποτελεί μια πρωτοβουλία μια συγκεκριμένη κυβέρνηση. Και όταν αντικατασταθεί αυτή η κυβέρνηση στην εξουσία, δεν συνεχίζεται η προσπάθεια. Δεν είναι βέβαιο δηλαδή αν θα συνεχίσει να προωθεί το μηχανισμό PCD με τον ίδιο ρυθμό ή αν θα υπάρξει κάτι καινούριο κτλ. Όταν διεξάγαμε την μελέτη, Είπαμε ότι ίσως χρειάζονται και 20 χρόνια μέχρι ότου ε, δημιουργηθεί κάποιος κώδικας για την εφαρμογή της PCT. Ε, e ε, έλλειψη και χρηματοδοτική υποστήριξης. Εκεί λοιπόν γίνεται η λιγότερη δουλειά και ίσως είναι και το μεγαλύτερο θέμα διότι αν θέλετε να προωθήσετε το PCD πρέπει να υπάρξει και συνεργασία και με άλλα υπουργεία. να μεταβείτε και αλλού δηλαδή και σε άλλα υπουργεία για να πείσετε περί της αξίας της PCD. όταν δηλαδή αξιωματούχοι αρμόδιοι για θέματα ανάπτυξη πηγαίνουν στο Υπουργείο Οικονομικών, ε, καλούνται να συνεργαστούν με ειδικού στον τομέα του. Οι διπλωμάτε, για παράδειγμα, που πρέπει ταυτόχρονα να ασχολούνται με πολλά και διαφορετικά θέματα. Άρα χρειάζονται καλή υποστήριξη έρευνα προ την κατεύθυνση αυτή. Έρευνα για την υψηλή σημαίνει ότι πρέπει να ξεφεύγουμε και από τη μελέτη συγκεκριμένων επεισοδίων. Είναι δύσκολο αυτό να εξεταστεί η της σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Έρχομαι στα συμπεράσματα. Προηγουμένως άλλοι μίλησαν για τους πέντε ευρύτερους τομείς. Τώρα στα συμπεράσματα του ε, Συμβουλίου, το οποίο δέχεται την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αντιμετωπίσει συνολικότερα την PCD. Αυτά βασίζονται και σε μια προηγούμενη έκθεση που αναφερόταν ότι υπάρχει ανάγκη να γίνει μεγαλύτερη, να πολύ μεγαλύτερε επενδύσει, ε, πολύ μεγαλύτερη επένδυση μάλλον στον διάλογο με τι αναπτυσσόμενε χώρε. Και μάλιστα τώρα όταν, ε, όπου οι χώρες εκεί για πρώτη φορά χρησιμοποίησαν το άρθρο 12 της Συμφωνίας Κοτονού και ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, εξετάσει, να εξηγήσει τις νέες πολιτικές τις ίδιες και από τότε που υπογράφηκε η συνθήκη Κοτονού δεν έχουν κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας που διαθέτουν η Εύα δεν αναφέρεται στο σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου όπως το λέω και στη διαφάνειά μου σήμερα που τα εξέτασα τα συμπεράσματα αυτά βρίσκονται ακόμα στα χέρια της μόνιμης αντιπροσωπείας, των μόνιμων αντιπροσωπιών δηλαδή, αλλά μάλλον αυτή την τελική μορφή θα λάβουν, άρα δεν γίνεται συζήτηση στο Συμβούλιο στα συμπεράσματα δηλαδή για την ΕΒΑΣΥΝ. Θα περιμένουν μάλλον να δουν τι θα ε, αποφασίσει η Κοπενχάγη και ίσως μετά να συζητήσουν τα σχετικά στο Παρίσι, μάλλον και όχι στις Βρυξέλλες, Και επειδή η Κοπενχάγη ίσως επηρεάσει σημαντικά το τι εννοούμε ως ε, Ευρωπαϊκή Βοήθεια Ανάπτυξη ΣΥΝ, ενώ οι περισσότερες συζητήσεις για τους ορισμούς της ΕΒΑ στρέφονταν γύρω από τους φόβους ορισμένους ότι, ορισμένων ότι τώρα θα μπουν και άλλα θέματα, ενώ περισσότερο θα κινηθεί γύρω από τις αλλαγές του κλίματος. Το Συμβούλιο πάντως δέχτηκε τους πέντε τομείς από την ανακοίνωση Επιτροπής άλλαξε έναν μόνο για την διανοητική ιδιοκτησία τον πρώτο και, αποφάσισε να, και προτείνει μάλλον να αποκληθεί εμπόριο και επίσης θέματα, να ενταχθούν εκεί και θέματα φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής. Τέλος, και μια προσπάθεια αναβολής κατά κάποιο τρόπο που λέει ότι το σχέδιο δράσης το σχέδιο εργασιών δηλαδή της PCT θα αναβληθεί για το 2010 θα πρέπει ε, να προβλέπει συγκεκριμένες κατευθύνσεις θα πρέπει να είναι λειτουργικό και να ενταχθεί στο διάλογο με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Στα ίδια συμπεράσματα οι φορείς καλούνται να υποβάλουν σχέδια. Αλλά αυτά για του χρόνου ενώ για την ώρα διαγράφονται μόνο τα γενικότερα πλαίσια και οι πέντε τομείς. Για τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τώρα στην προώθηση της PCD θα αφήσω μερικά πράγματα γιατί κάπως έχω μακρηγορήσει. Σε μια μελέτη που κάναμε το 2007 εξετάσαμε και το τι κάνει η Επιτροπή σας και εξετάζοντας τις διάφορες αρμοδιότητες είδαμε ότι υπάρχει αύξηση του αριθμού εκθέσεων που αναφέρονται στην PCD και είδαμε επίσης ότι οι επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου διεξάγουν σημαντικό έργο σε σχέση με την πρόθεση της PCD. Τώρα για τα κοινοβούλια αυτής χωρισμένη ένα θέμα κριτικής είναι ότι οι επιτροπές συνήθως στα όσα μελετούν δεν υπερβαίνουν τα όρια των τομέων που τους έχουν ανατεθεί. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν γίνει και περισσότερο από πειράματα φτιάχνοντας κατά κάποιο τρόπο οριζόντιες επιτροπές για την ε, αλλαγή του κλίματος ανάμεσα στο 2007 και 2008 και για το χρόνο επίσης εξετάζοντας και την εντολή της Επιτροπής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπάρχει σαφής αναφορά για την προώθηση της PCD. Ορισμένοι θεωρούν ότι de facto εντάσσεται στις αρμοδιότητες της παρούσας Επιτροπής. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν το ενδεχόμενο μπορεί να θεωρηθεί και η Επιτροπή Ανάπτυξης ως οριζόντια επιτροπή και επομένω να μπορεί να προβαίνει σε κοινέ δηλώσει με άλλε ε, κοινοβουλευτικέ επιτροπέ. Κάτι τέτοιο θα ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο. Η, η Επιτροπή επίση πρέπει να προσαρμοστεί και στη νέα κατάσταση που θα προκύψει από την εφαρμογή τη συνθήκη τη ε, Λισαβόνα. Βέβαια, θα υπάρξουν και πολλές ιδέες και μία κρίσιμη είναι ότι ενδεχομένως η ευθύνη για την PCD μπορεί να μοιραστεί ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Θα μπορέσει να θεσπιστεί ένας ε, διαρκής διάλογος με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Θα έρχεται εδώ ο ύπατος εκπρόσωπος ή θα έρχεται εδώ ο Επίτροπος Ανάπτυξης για να συζητεί θέματα PCD μαζί σας. Κατά τη γνώμη μας αυτά τα θέματα παραμένουν ανοιχτά. Εξετάζοντας παλαιότερες ημερήσεις διατάξεις της ε, μικτής ε, κοινοβουλευτικής συνέλευσης, η PCD δεν, ε, έχει, εξετάσει, δεν έχει εξεταστεί πάντοτε ως τέτοιο θέμα. Απάντως εδώ νομίζω να ανοίγονται ευκαιρίες για να ζητηθεί περισσότερο και να προωθηθεί περισσότερο η PCD. Θα αρκεστώ σε αυτά. Έχω τέσσερις ε, βουλευτές που θέλουν να παρέμβουν. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Κάσμαν. Ο κύριος Κάσμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την συγκεκριά μας, τον εκπρόσωπο της Επιτροπής και τους δύο μιλητές που μας έκαναν τις παρουσιάσεις τους. Οι περισσότερες από τις ανησυχίες που παρουσίασαν οι δύο, που παρουσίασαν οι δύο μιλητές είναι και δικές μου. Να κάνω μια πρόταση λοιπόν για τις οριζόντιες επιτροπές, επιτροπές καταρχάς. Νομίζω ότι πρέπει να αποφύγουμε να επινοήσουμε ξανά τον τροχό. Πρέπει να σκεφτούμε ότι μπορεί να έχουμε ένα μόνιμο εισηγητή, διαρκή εισηγητή για θέματα πολιτικής συνοχής. Όπως για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή για τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών. Έχω και εγώ λοιπόν κάποιες ανησυχίες, τις οποίες φρόντισα να τις αναφέρω στους ηθήνοντες από τότε υπάρξει νέα θητεία. Πρώτα απ' όλα η έλλειψη δέσμευση των αναπτυσσόμενων χωρών ε, για τη συμμετοχή του στο διάλογο αυτό, διότι γνωρίζουν την πραγματικότητα τη πολιτική συνοχή ε, και μάλιστα εξαιδία πείρα. Φαίνεται ότι δεν έχουμε καταφέρει να το συμπεριλάβουμε στη διαδικασία. Κάποιε φορέ βλέπουμε τα κράτη-μέλη να παρακάμπτουν τι υποχρεώσει του και να προβλέπουν ένα 7% αναπτυξιακή βοήθεια ή να συμπεριλαμβάνουν τι κλιματικέ αλλαγέ στην ε, κατηγορία αυτή είναι σαν να προσπαθούν να αποφύγουν τις ευθύνε τους, τις υποχρεώσει τους. Δηλαδή, κάποιες φορές οι αποφάσει μπορεί να μην έχουν θετικά αποτελέσματα για τα προγράμματα, αλλά μπορεί να έχουν θετικά αποτελέσματα για τους επενδυτέ. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σαφείς και να είμαι απολύτως ειλικρινής λέγοντας ότι όλη η συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό μου φαίνεται. Ε, και θα ήθελα να είμαι εδώ διπλωματικό, διότι το έλεγα για το οροσκόπιό μου για αυτό το μήνα. Ε, η συζήτηση αυτή είναι αρκετά αδύναμη στα επιχειρήματα από την πλευρά του Επιτροπή και του Συμβουλίου. Ωραία είναι να έχουμε πολιτική συνοχή και πιστεύω ότι, ότι μπορεί να είναι πολύ καλές οι συνολικές προθέσεις αλλά εδώ το πρόβλημα είναι το ποιο θα έχει την εξουσία, ποιο θα αρπάξει την εξουσία και την αναπτυξιακό προπολογισμό και αν θα αυτό να τον αναλάβει ο το εκπρόσωπο των ε, εξωτερικών υποθέσεων. Σε καμία περίπτωση θα μπορούσα να εγκρίνω μια τέτοια επιλογή. Αυτό είναι τελείω ξένο από όσα έχει κάνει ω τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε τόσου πολλού τομεί που αφορούν την ανάπτυξη και την ε, βοήθεια. Ναι, να δούμε ε, μέσα που έχουν να κάνουμε το εμπόριο ή ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να επηρεάσουμε, για να γλιτώσουμε την Αφρική από αυτή την εξάρτησή της που κάποιες φορές ενθαρρύνεται και έχει και αναγνωριστεί ε, τι προκαλεί βοήθεια και η δική μας ε, προσέγγιση της αναπτυξιακής βοήθειας. Συμμερίζομαι την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Πρόεδρε ήθελα να επεκταθώ σε αυτά τα δύο ζητήματα ότι χρειαζόμαστε πολιτική συνοχή μεν αλλά θα μου επιτρέψετε εδώ να καταδείξω ένα κράτο μέλο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση η Γαλλία να συμφωνήσει να πάυσει και να εκριζωθεί η κοινή αγροτική πολιτική, η οποία η ίδια βελτίωσε τόσο πολύ τα δικαιώματα και τον ως, τα δικαιώματα και την ε, διαβίωση όσων ζουν στον αναπτυσσόμενο χρόνο. Δεν, κόσμο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να καταργηθούν οι επιδοτήσεις, οι εξαγωγικές ε, βοήθειε. Και ξέρετε ότι στον Ηνωμένο Βασίλειο ζητήσαμε πολλέ φορέ αυτή τη μεταρρύθμιση και ουδέποτε πετυχάμε κάτι. Και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, όπου πέρασα μια δεκαετή θητεία, κάποιοι μου λένε μια δεκαετία είναι πάρα πολύ καιρό, αλλά έχουμε πολιτικά μέσα, α τα χρησιμοποιήσουμε επιτέλου, α τα αξιοποιήσουμε για να βελτιώσουμε τι ζωέ των ανθρώπων που ζουν στον αναπτυσσόμενο κόσμο απλώς να επιβάλαμε και να εφαρμόζαμε τις συνθήκες και τις συμφωνίε που έχουμε μαζί τους, με τι τρίτε χώρε πολλά θα πετυχαίναμε. Για την ένδυα, τη φτώχεια, τα βασανιστήρια, τον πόλεμο, τις παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μόνο και μόνο αυτά, η αντιμετώπιση μόνο και μόνο αυτών των ζητημάτων, αυτά θα έδιναν τέρμα στην αιμορραγία των ίδιων των ανθρώπων που εγκαταλείπουν τι χώρε του. Μόνο και μόνο γιατί αναζητούν μια καλύτερη ζωή και ίσω και για να προσφέρουν μια καλύτερη ζωή σε αυτού που μένουν πίσω του, όχι μόνο για του εαυτού του. Δεν μπορώ να συνεχίσω νομίζω. Έχω σοβαρότατε αμφιβολίε για αυτό το PCD Plus. Ας φροντίσουμε πολιτικέ που έχουμε να λειτουργήσουν. Α βεβαιωθούμε ότι όλοι έχουμε το ίδιο επίπεδο φιλοδοξιών ότι θέλουμε να πετύχουμε τους ίδιους στόχους και κυρίως ότι έχουμε διασφαλίσει την πολιτική συνοχή προς όφελος της ανάπτυξης και ότι η ανάπτυξη δεν ωφελεί με τη σειρά της τις εξωτερικές σχέσεις ε, των επιτρόπων ή του υψηλήπα του προσώπου. Ουδέποτε αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τη μεταμελιά μου για τον ενθουσιασμό και το πάθος μου, αλλά με οδηγεί προς αυτό η ίδια Επιτροπή. Νομίζω ότι θα είναι λοιπόν ένας παθιασμένος πόλεμος αυτός, προκειμένου να πετύχουμε αυτά που επιθυμούμε. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γκέρενς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να πω ευθύς εξ αρχής ότι αυτή είναι μόνο μια αρχή των συζητήσεων για την πολιτική συνοχή και την επεξιακή βοήθεια συν. Διότι αν ήταν αρχή και το τέλος, θα χάναμε δύο σημαντικού εταίρους. Πρώτα απ' όλα εδώ το Συμβούλιο που απουσιάζει, ενώ τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν ε, καθοριστική σημασία στην αναπτυξιακή βοήθεια. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο που εκπροσωπεί μόνο 20% της συνολικής βοήθειας κρατική βοήθεια προ την ανάπτυξη. Κατά δεύτερο, θα μα έλειπε... θα έλειπαν και οι εταίροι μα, οι εταίροι μα από τον Νότο, οι εκπρόσωποι των αναπτυσσόμενων χωρών των ιδίων. Διότι αν θέλουμε να είμαστε εδώ συνεπεί πρέπει να είμαστε συνεπείς και ω προς τις αρχές μας. Αυτέ που διατηνόμαστε ότι έχουμε τουλάχιστον. Εταιρική σχέση διαφημίζουμε ότι έχουμε, η εταιρική σχέση μα επιβάλλει να ακούμε και του εταίρου μα. Ιδάλω, επιστρέφουμε στην επικαιοκρατία. Ίσως αυτό κάποιοι να το επιθυμούν, αλλά νομίζω ότι η πλειοψηφία είναι κατά της αρχής αυτής και της επιστροφής της πολιτικής στην απεικιοκρατία. Έπειτα, διακυβέρνηση συνοχή, αλλά τι σημαίνει συνοχή, πολυδιάστατη, πολυδιάστατη συνοχή, για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση πρώτα απ' όλα. Λείπει από τη συζήτησή μας ο ύπατος εκπρόσωπος. Λείπει ο μελλοντικό ύπατος εκπρόσωπος που δεν ξέρω αν θα ονομαστεί Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων, αλλά τουλάχιστον θα προεδρεύσει με όλο του το κύρο και με τη διπλή του ιδιότητα ω αντιπρόεδρο τη Επιτροπή και είπα του ε, προσώπου, που θα ασχολείται με τι εξωτερικέ σχέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λέω γιατί με ιδιαίτερη χαρά μου άκουσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λέει ότι η στρατιωτική διάσταση της ευρωπαϊκής πολιτικής πρέπει να λάβει υπόψη τις επιθυμίες και προσδοκίες της αναπτυξιακής πολιτικής. Ελπίζω ότι την ερμηνεία αυτή που μόλις κάνατε θα την συμμεριστεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σύνολό της. Ελπίζω ότι θα εισακουστεί και από τον ήπατο εκπρόσωπο. Ελπίζω ότι θα είναι η ίδια ερμηνεία και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου των Υπουργών. Εάν όλοι συμμεριζόμαστε αυτή την άποψη, γιατί όμω καταργήσαμε το Συμβούλιο των ε, Υπουργών Ανάπτυξη πριν από λίγα χρόνια. Ήμασταν λίγοι εκείνοι που αγωνίστηκαν κατά τη κατάργηση αυτού του Συμβουλίου, του σχηματισμού του Συμβουλίου. ιδίω ο Πρωθυπουργό τη χώρα μου και ο πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, ο Πατ Κόξ τότε, είχε αντιταχθεί στην κατάργηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Συμβουλίου μάλλον των Υπουργών Ανάπτυξης. Νομίζω ότι η διακυβέρνηση είναι κυρίως ε, μια κατάσταση νοητική του πώς ε, προσεγγίζουμε αυτή την πολιτική. Διότι αν δούμε την ιεραρχία της Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης, εάν βάλουμε στην δεύτερη θέση, στα καθίσματα της δεύτερης θέσης στην πολιτική της ανάπτυξης, τότε θα τις δώσουμε μια χρησιμοθυρική διάσταση. Και αν θέλουμε έτσι να την αντιμετωπίσουμε, δεν μπορούμε πια να μιλάμε για συνοχή. Εάν να δούμε χρησιμοθυρικά την αναπτυξική προσέγγιση, η πολιτική αναπτύξική βοήθειας δεν ε, δικαιολογεί τη βοήθεια που έχουμε προσφέρει στις αναπτυσσόμενες χώρες, ούτε στα πλαίσια των κλιματικών αλλαγών. Ένα τεστ λοιπόν, μια δοκιμή για την, συνοχή, την πολιτική συνοχή θα είναι η Σύνοδος της Κοπενχάγης. Εάν τα χρήματα που θα επενδυθούν προς το συμφέρον, προς το όφελος των, της καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών ε, για τις αναπτυσσόμενες χώρες, εάν τα ποσά αυτά θεωρηθούν ότι εξηγεί βοήθεια, εκεί δεν θα συμφωνώ καθόλου. Διότι αυτά τα χρήματα που θα επενδυθούν θα πρέπει να είναι πρόσθετα κονδύλια, θα πρέπει να είμαστε λοιπόν απόλυτα σαφεί ω προ τον ορισμό τη κρατική βοήθεια για την ανάπτυξη και νομίζω ότι εδώ σε αυτή τη συνεδρίαση μπορούμε να το κάνουμε, αλλά αν βγούμε από την αίθουσα σα ορκίζομαι ότι θα έχουμε όλη διαφορετική αντίληψη για το τι είναι κρατική βοήθεια για την ανάπτυξη. το ODA εντό αιθούση δεν είναι το ίδιο με αυτό που αντιλαμβανόμαστε εκτό αιθούση. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι και οι υπόλοιποι εταίροι μα σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση για την Αναπτυξική Βοήθεια θα πρέπει να συμμερίζονται την ίδια αντίληψη. Θα πρέπει επί των ενιών να μην υπάρχει καμία σύγχυση. Θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφεί. Τρίτη παρατήρηση. Δεν θέλω να παραμερίσουμε και να παραβλέψουμε ό,τι έχει να κάνει με τις συγκρούσεις, την όλη, τον όλο προβληματισμό περί συγκρούσεων. Οι συγκρούσεις προκύπτουν από την ανεπάρκη καταπολέμηση της ένδυας. Θα πρέπει η κρατική βοήθεια για την ανάπτυξη να επικεντρωθεί ακριβώς στην καταπολέμηση της ένδυας. Δεν είμαι καθόλου κατά μια ευρύτερη προσέγγιση που να συμπεριλαμβάνει και άλλα στοιχεία όπως το εμπόριο κατά κύριο λόγο ή ό,τι συμβαίνει σε επίπεδο των εσωτερικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να δούμε και τον αντίκτυπο όλων αυτών των πολιτικών εκτό Ένωση. Να τα βλέπουμε όλα αυτά σφαιρικά. Όμω σα παραπέμπω στην μελέτη που είχε γίνει στα πλαίσια της έκθεσης ε, της ευθύνης για την ανατεξική βοήθεια και είχε κάνει μια πολύ καλή ανάλυση των συγκρούσεων, των ε, μιζώνων ε, σύγχρονων συγκρούσεων που έχουν σχέση με την ένδια με την απουσία ένδυα ή την απουσία καταπολέμηση, προσπαθειών καταπολέμηση τη ένδυα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε συνετοί και επιφυλακτικοί αν θέλουμε να έχουμε μια συζήτηση σαφή που μπορεί να οδηγήσει τελικά σε συγκεκριμένα χειροπιαστά αποτελέσματα. Επιμένω στη διευκρίνηση των όρων. Θέλουμε σαφείς και διαυγείς ορισμούς όταν μιλάμε για πολιτική συνοχή ή συνοχή των πολιτικών. Και μια τελευταία παρατήρηση. Εάν διαβουλευτούμε με του εκπροσώπου των 100 μελών και συζητήσουμε μαζί του, θα δούμε ότι υπάρχουν τα νέα κράτη-μέλη που προτιμούν την, ε, προβλημα, την όλη φιλοσοφία περί σχέσεων με ανατολικές χώρες, ενώ άλλοι που προτιμούν τη Λατινική Αμερική ή τη Μεσόγειο και κάποιοι έχουν και σφαιρικότερη θεώρηση. Υπάρχουν λοιπόν τόσε διαφορετικέ απόψει για την ε, κρατική αναπτυξιακή βοήθεια, υπάρχουν τόσε απόψει όσε και τα κάτι μέλη. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να έχουμε μια συνεκτική προσέγγιση και μια ενιαία άποψη. Δεν λέω να έχουμε μία ενιαία φιλοσοφία μόνον, αλλά να είμαστε συνεπεί. Αν θέλουμε να είμαστε συνεπεί, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη να δεσμευτεί και να λάβει μέρο στον ίδιο αγώνα. Δεν θα πρέπει να έχουμε κατακαιρματισμό των ε, πεπιθήσεων και των απόψεων. Υπάρχουν λοιπόν ε, πολλά που πρέπει να γίνουν. Σας εύχομαι πολύ και καλή δουλειά κυρία Κέλλερ. <clears throat> Είχαμε μια πρώτη εικόνα, ένα το για για το περιεχόμενο της εκθεσής σας, για τη διάσταση της συνοχής, αλλά θα πρέπει να επικεντρωθούμε αυτής εξ αρχής ε, στην εκκίνηση αυτής της στο θέμα των ορισμών να είμαστε βέβαιοι όταν μιλάμε για κάτι, ότι μιλάμε για τα ίδια πράγματα. Ότι καταλαβαίνουμε όλοι το ίδιο. Ανατρέχοντας μάλιστα σε όρους, ιδίως στον, ε, όταν ανατρέχουμε σε όρους, ιδίως στον τομέα των συνεχής των πολιτικών. Ευχαριστούμε. Το λόγο και ο κύριος Μπέρμαν. Και θα συνεχίσω στα γαλλικά όπως και ο προλαλής σας. Αυτό που κάπως με ξαφνιάζει σε αυτή τη συζήτηση είναι ότι εδώ και χρόνια αγωνιζόμαστε για μια συνοχή όλων των ευρωπαϊκών ε, πολιτικών. Οι επιδοτήσεις εισαγωγών στη Γεωργία, οι αλληλευτικές συμφωνίες και το καθεξής. Τώρα έχουμε μπροστά μας μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει να μας προτείνει νέα θέματα, αγώνες σε νέους τόπους. Όμως, νομίζω ότι η απόπειρα αυτή, παρόλο που είναι ειλικρινής και ευφύης, δεν θα πρέπει να μας αφήσει να παραδεχτούμε ότι είμαστε καχύποπτοι. Παρόλο που η ανάλυση είναι πολύ καλή, εύστοχη, δεν πάβει να ακυρώνει την εγκυρότητα της, δεν πάει να μην ε, την εγκυρότητα της ανάλυσης της ε, Φραντσίσκα Κέλλερ. Και τα δικά της επιχειρήματα είναι εύστοχα. Και για τον επιπλέον λόγο ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αύξηση των ε, εξαγωγικών επιδοτήσεων για τα γαλακτοκομικά προϊόντα γιατί υπάρχει ελληνική συμφωνία που έχει ανασταλεί βέβαια με τη Γουινέα, αλλά δεν ήταν ούτως ή άλλως εξ αρχής ε, συνεκτική. Γιατί στη συμφωνία TRIPS υπάρχουν διαπραγματεύσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση με, την κεντρική, με τι χώρε τη Κεντρική Αμερική. Και αν σωστά είμαι πληροφορημένο, έχει σκοπό να παρατείνει την περίοδο κατά την οποία θα προστατεύει τα διπλώματα ευρεσιτεχνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε και πάλι θα εμπλακούν εδώ και τα ιατρικά προϊόντα και η πρόσβαση στα φάρμακα για αυτέ τι χώρε. Όλα αυτά δείχνουν μια φρικτή ασυνέπεια εκ μέρους μας, αδικαιολόγητη, απαράδεκτη. Όταν μειώνουμε την προβολή της, ε, την παρουσία της Γεωργίας όλη αυτή την ανάλυση, μιλάμε για επισητιστική ασφάλεια, πολύ ωραίο είναι αυτό, μου αρέσει, αλλά υπάρχει ένας κίνδυνος εδώ να παραμελήσουμε τη Γεωργία ως πεδίο δράσης. Και εδώ μπορεί να δώσουμε και μεγαλύτερη έμφαση στο ίδιο συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ότι στο όφελος των ε, αναπτυσσόμενων χωρών. Ο κίνδυνος αυτός λοιπόν πρέπει να αποφευχθεί. Δεν θα πρέπει να αποφευχθεί μόνο με, το, με τη συμβολή του Ombudsman, του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή όχι, εμεί πρέπει να είμαστε διαμεσολαβητέ μετά την θέση σε ισχύ τη ε, συνθήκη τη Λισαβόνα. Εμεί αναλαμβάνουμε το καθήκον να υλοποιήσουμε τι συνθήκε και όλε τι συνθήκε. Αυτό είναι ο στόχο τη συνοχή που τόσο πολύ επιδιώκουμε. Εμεί πρέπει να προσφύγουμε στο ΔΕΚ. Εμεί πρέπει να παρουσιάσουμε μια υπόθεση. Όχι ο διαμεσολαβητή. Είναι πολιτική δράση κι αυτή. Είμαι λοιπόν ε, μάλλον ε, άφωνο με όλα αυτά, διότι δεν έχω καταλάβει πώ θα προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλε αυτέ τι δράσει. Παρά τι καλέ προθέσει που ανακοινώνει το κείμενό σα, μου φαίνεται ότι δείχνεται αρκετή καχυποψία. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Κύριε Σαργεντίνη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν πρώτα αυτή η ή όταν το είδα εγώ πρώτη φορά στην ημερήσια διάταξη αυτή τη συνοχή για την αναπτυξιακή βοήθεια, ενθουσιάστηκα. Διότι αυτό αποτελεί το συνολικό κάλυμα. Εγώ γι' αυτό έχω έρθει σε αυτή την Επιτροπή. Συνοχή, δηλαδή συνεκτικές πολιτικές που να επιτρέψουν την ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών ή πάντως να μην ανακόψουν την ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών. Ε, με, την, με, με εφαρμογή εσφαλμένων πολιτικών. Εξετάζοντα την ατζέντα αυτή, περιλαμβάνονται ορισμένα πράγματα τα οποία δεν είναι απαραίτητο να συζητηθούν εάν όντω θέλουμε να μιλήσουμε για συνεκτικέ πολιτικέ. Οι συνέπειε τη οικονομική και χρηματοδοτική κρίση για την ασφάλεια των τροφίμων, η Συμφωνία ΑΚΕ Ευρωπαϊκή Ένωση για την η Συμφωνία Κοτονού. Αυτά μπορούν να φύγουν από την ατζέντα. Εμεί να εμείνουμε σε ένα θέμα, συνοχή δηλαδή των πολιτικών ανάπτυξης. Ο κ. Γιώργος σωστά είπε ότι πρόκειται για θέμα ορισμών. Ακούγοντας ε, ε, συνοχή πολιτικής ανάπτυξης, μου φαίνεται ότι είναι ένας διαφορετικός, δεν είναι ένα διαφορετικός τρόπος για να μην ξεχάσουμε μονάχα την ανάπτυξη όταν θα αρχίσει η ευρωπαϊκή εξωτερική δράση. Είναι ένας τρόπος για να διασφαλίσουμε ώστε όλες οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι τέτοιες που να μην βλάπτουν τις αναπτυσσόμενες χώρες ή, πάντως, ε, ή, και, ή και να τις βοηθούν, να ενισχύουν την ανάπτυξη. Αυτά σκέφτομαι. Αφενός θεωρώ ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε το έργο της Γενικής Διεύθυνσης τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί πράγματι ε, ε, εργάζεται σκληρά και πράγματι κάνει βήματα προ τα εμπρό και πράγματι το μπουκάλι είναι μισογεμάτο. Από την άλλη μεριά όμω, η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξη πρέπει να αρχίσει τη μάχη αυτή με τη, μέσα στην όρκο του Κομισιόν και με το Συμβούλιο, γιατί αν δεν το κάνει αυτό, πώ θα προχωρήσουμε. Δηλαδή, τι να κάνω, να επενέσω το έργο που έχει επιτευχθεί, να ε, επικρίνω το ότι δεν έχει προχωρήσει αρκετά. Και αυτό το δεύτερο συνέστημα αρχίζει και κερδίζει μέσα στο μυαλό μου. Και η ερώτηση μου προς την Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι γιατί. Γιατί δεν επανεξετάζουμε τον ορισμό της συνοχής πολιτικής ανάπτυξης. Ας ζυγίσουμε τις λέξεις αυτές, να δούμε τι ε, ακριβώς αξία έχουν. Και μετά μπορούμε να προχωρήσουμε στον αγώνα με αυτές. Δεν μπορείς να κάνεις συνοχή πολιτικής ανάπτυξης χωρίς εμπόριο. Και όταν μιλούμε για ασφάλεια τροφίμων πρέπει πάλι να μιλήσουμε για εμπόριο. Αυτά όμως είναι ανοησίες διότι το εμπόριο δίνει τη δυνατότητα στις ε, χώρες να ε, κάνουν συναλλαγές μαζί μας. Πρόσφατα ο αρμόδιος υπουργός της ε, Νότιας Αφρικής μου εξήγησε σε μια διάλεξη με ποιο τρόπο με ε, με ποιο τρόπο διεξάγεται το εμπόριο αυτό. Και εγώ τράπηκα και ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί ε, επιλέγουμε τον, την οδό της ε, ελάχιστης αντίδρασης και δεν κάνουμε μια πιο έντονη προσπάθεια. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω τους διερμηνείς αν μπορούν να μείνουν μαζί μας 10 λεπτά παραπάνω γιατί είναι σημαντικό το θέμα και θα ήθελα να μεταφράζονται όλοι. Κυρία Λεβίν, παρακαλώ, ευχαριστώ πολύ. Απόλυτα συμφωνώ με την κυρία Αζεντίνη. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια κυρία Κέλλερ για την εξαιρετική δουλειά που έκανε. Ανησυχώ έντονα, πολύ έντονα για αυτή τη συζήτηση για το ODA Plus και το νέο ορισμό του ODA. τι θα μπορούσε να σημαίνει η συνεκτικότητα και συνοχή πολιτικής στην πρακτική εφαρμογή και σε ποιους τομείς θα μπορούσε να αποκληθεί ODA στο εμπόριο ή σε κάτι άλλο. Θα ήθελα λοιπόν απλά και μόνο να αναφέρω τις ε, συμφωνίες εταιρικής σχέσης αλλίας, Αποκαλούνται συμφωνίες ή συμβάσεις εταιρικής σχέσης ε, και θα έλεγα μια και αυτή η πολιτική για την συνεκτικότητα ξεκίνησε την εξέταση αυτών των θεμάτων το αποτέλεσμα τώρα είναι ότι προκαθορίζουμε ένα συγκεκριμένο ποσοστό των συμφωνιών αλίας για να καλύπτουν κάποιους τομείς και λέμε στις αναπτυσσόμενες χώρες ότι πρέπει να χρησιμοποιούν 50% των κονδυλίων που πληρώνουμε εμείς για την αλία στα χωρικά τους ύδατα για να αναπτύξουν την, ε, ε, το λιμενική, την ε, λιμενική τους υπηρεσία, την ακτοφυλακή ή για την εσωτερική πολιτική και την πολιτική αλλιευμάτων από πλευρά τους. Το πρόβλημα όμω είναι, λοιπόν, πρώτον, εμείς κάνουμε αυτές τις συμφωνίες με πολύ διεφθαρμένες κυβερνήσεις και χώρες. Και όταν κάνει την αποτίμηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδεικνύεται το αντίθετο μάλιστα συμβαίνει ότι τα χρήματα αυτά δεν πάνε για τους τομείς και δράσεις που προβλέπονται από τις συμφωνίες μια και είναι διεφθαρμένες αυτές τι κυβερνήσεις και χώρες και σε σχέση με την βοήθεια όταν θα δίνουμε μόνο τα χρήματα αυτά αν μπορούμε να αλλιεύουμε στα χωρικά ύδατα αυτών των χωρών ε, υπάρχει όρος και προπόθεση λοιπόν που ε, εμπνέει αυτές τις συμφωνίες σε σχέση με την υποστήριξη λοιπόν της ε, αλλιευτικής τους ε, ε, βιομηχανίας και της ασφάλειας τροφίμων και της επάρκειάς τους σε τρόφιμα. Αυτό θα ήταν αυτό το οποίο θα αποκαλούσαμε βοήθεια. Έχουμε όμως εμείς ισχυρά επιδοτούμενα μεγάλα σκάφη που αλλιεύουν στα χωρικά ιδέα αυτών των χωρών και αυτό με ανησυχεί πάρα πολύ εμένα. Και τι γίνεται με τον ορισμό της βοήθειας. Βοήθειας. Θα πρέπει να είναι πολύ αυστηρός και όταν πρόκειται για συμφωνίες αλληλείας, ε, δεν, δεν πρέπει να κάνουμε λόγο για ανάπτυξη και βοήθεια μέσω αυτών των συμφωνιών. Είναι εμπορικέ συμφωνίε αυτέ Και τελεία και παύλα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω προσπαθώντας να απαντήσω στα πέντε ερωτήματα της κυρία Κέλλερ όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση. Πώς επιλέχθησαν οι πέντε προτεραιότητες, οι τέσσερις συνολικές προκλήσεις. Νομίζω στην ανακοίνωσή μας ε, πενισόμαστε ποιε είναι και τους λόγους που τις επιλέξαμε. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για σφαιρικές προκλήσεις που είναι σημαντικές από την άποψη της ανάπτυξης. Και το κάναμε αυτό μελετώντας τις εκθέσεις που μας φτάνουν από τις αντιπροσωπείες μας. Ξέρετε, τα στρατηγικά έγγραφα αναχώρα έχουν πλέον ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο για την πολιτική συνοχή. Έχουμε λοιπόν αναλύσεις που μας οδηγούν απευθεία σε κάθε αναλυόμενη χώρα εταίρο. Και βεβαίω υπήρξαν και διαβουλεύσει που έγιναν με, σε συνεργασία με ομάδε αναπτυσσόμενων χωρών. Υπάρχουν δύο τέτοιε εκθέσει και υπάρχουν και οι μελέτε συγκεκριμένων περιπτώσεων, όπω και αυτέ που έγιναν από τι μη κυβερνητικέ οργανώσει και ενημερώνουν για το ποιοι είναι οι πιο σημαντικότεροι προβληματισμοί σε σχέση με την ανάπτυξη. Δεύτερο κριτήριο ήταν βεβαίως η όλη, όλος προβληματισμός αυτός να έχει πολιτική προτεραιότητα ούτως ή άλλως στην ατζέντα, στη σειρά προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να υπάρχει και περιθώριο ελιγμών για να είμαστε πραγματικά ενεργοί στα πλαίσια της ε, ατζέντα της συνοχής. Έπρεπε λοιπόν να επιλέξουμε θέματα τα οποία να είναι προτεραιότητας έτσι κι αλλιώς για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τρίτο κριτήριο ήταν να υπάρχει κάποια διάρκεια ε, ως προς την ε, σημασία των ε, προκλήσεων αυτών. Τώρα, οι παραπομπέ στην τελευταία έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου, η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για τη συνοχή αφορούσε εξ όσων γνωρίζω, συγκεκριμένα ζητήματα, έχει το σύνολο της έκθεσης 2007 που έχει υποβάλει τον Σεπτέμβριο του 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα συγκεκριμένα αυτά ζητήματα ήταν η αλία και η ξυλία η υλοτομία εκεί σε συγκεκριμένο κεφάλαιο αναφερθήκαμε σε μηχανισμούς για βελτίωση της συνοχής και στην έκθεση του 2009 και ιδιαίτερως στο κεφάλαιο που αφοσιώθηκε στην αλληλευτική πολιτική. Τρίτον, για το screening, την ανάλυση και τον έλεγχο του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής και τον σχεδιασμό των προτάσεων για την ερχόμενη χρονιά, εντοπίσαμε πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να είναι εύστοχες για σκοπούς πολιτικής συνοχής και να έχουν και κάποιο όφελος για την ανάπτυξη. Ακολουθούμε το πρόγραμμα εργασιών τη Επιτροπή. Είναι εγκεκριμένο το πρόγραμμα αυτό. Συνεργαζόμαστε με τη διπρεσιακή ομάδα ε, στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής και ε, διαλέγουμε κάποιε πρωτοβουλίε προσπαθώντα να καταρτήσουμε και ένα κατάλογο προτεραιότητα. Διότι δεν μπορούμε να διαλέξουμε 500 πρωτοβουλίε και να πούμε ότι θα είμαστε ενεργοί και στι 500 ταυτόχρονα. Θελήσαμε λοιπόν να εντοπίσουμε πρωτοβουλίε που πραγματικά να έχουν σημαντικότατο αντίκτυπο για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Και προσπαθήσαμε να προβλέψουμε δράσεις για όλες αυτές τις προτεραιότητες και για τις τεχνικές αναλύσεις και τις αναλύσεις αντικτύπου. Επίσης, για τον τρόπο που θα κάνουμε τους εταίρους μας στην ανάπτυξη να συμμετάσχουν σε όλες αυτές τις μελέτες αντικτύπου. Από τον Ιανουάριο 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβλεψε καθημερινέ γραμμές για την μεθοδολογία των μελετών αντικτύπου και εισαγάγαμε ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο αντίκτυπω για την ανάπτυξη ιδιαίτερο κεφάλαιο πολύ πιο εξελιγμένο από ό,τι στο παρελθόν. Ιδίω με το να ζητούμε οι μελέτε αντικτύπου να εξετάζουν τις ενδεχόμενες επιπτώσεις μιας προτινόμενη πολιτικής για τις δυνατότητες των ε, χωρών που επιδιώκουν το στόχο της ανάπτυξη, αλλά κάνοντα και διαφοροποίηση ανάλογα με τις κατηγορίες ανάπτυξη των χωρών. Μια πρόταση στον ένα ή τον άλλο τομέα δεν θα έχει τον ίδιο αντίκτυπο στη Βραζιλία που ακόμη θεωρείται αναπτυσσόμενη χώρα ή στο Μαλί ή στο Μπαγκλαντέ. Έπρεπε λοιπόν να γίνει διαφοροποίηση των επιπτώσεων, είτε ανα κατηγορία χώρας, είτε ανα γεωγραφική περιοχή. Για κάθε πρωτοβουλία που προτείνατε. Οι κατευθυντήριε γραμμέ για τι μελέτε αντικτύπου επιβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να οργανώσει διαβουλεύσει με του ε, ενδεχόμενους εταίρους. Στο κεφάλαιο λοιπόν αυτό περί ανάπτυξης έχουμε συγκεκριμένη βάση για να κάνουμε τους εταίρους μα της ανάπτυξης να συμμετάσχουν ενεργότερα. Και για το επόμενο σημείο νομίζω ότι εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση πραγματικά. Πώς να βελτιώσουμε τη στάθμιση των πρόοδων σε σχέση με την ανάπτυξη. Αν διαβάσατε την έκθεση του 2009 θα διαπιστώσατε ότι σε σχέση με το 2007 προσθέσαμε ένα ακόμη κεφάλαιο κεφάλαιο που αποπειράται ουσιαστικά να μελετήσει κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις. Εξετάσαμε εκεί πώς επιτόπου σε κάποιες χώρες της Αφρικής μπορούμε να αποτιμήσουμε τις, συνέ... επιπτώσεις ε, των ευρωπαϊκών πολιτικών πέραν των αναπτυξιακών ε, για τις δυνατότητες ε, σε σχέση με συγκεκριμένους στόχους της χιλιετίας, συγκεκριμένα προγράμματα και σχέδια. Από την πρώτη μας ανάλυση διεξεγάγαμε κάποια πρώτα συμπεράσματα για το μέλλον. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα μεθοδολογίας σε πρώτη φάση, ιδίω πρόβλημα δεδομένων. Είναι δύσκολο να συλλεχθούν τα δεδομένα για τις επιπτώσεις των πολιτικών αυτών, αλλά είναι μια δουλειά που θα την ε, συνεχίσουμε. Σε συνεργασία πάντοτε με τον ΟΣΑ ο ΣΑ που έχει και αυτός ε, δυνατότητες ε, ανάλυσης και έρευνας ε, και σε ό,τι αφορά τη συνοχή, ιδιαίτερα ανεπτυγμένες. Θα συνεργαστούμε στενά λοιπόν για αυτούς τους σκοπούς. Τώρα, η μέτρηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων ως προς τη συνοχή, η έκθεση είναι ένα από αυτά τα εργαλεία που θα επέτρεπαν να τονώσουμε την όλη συζήτηση. Ελπίζουμε λοιπόν να εξυπηρετήσει αυτό το σκοπό. Για το μέλλον ωστόσο, το να εντοπίσουμε δείκτες προόδου είναι κάτι που το επιθυμούμε. Ιδίω βάσει της νέας μας προσέγγισης που θα επιτρέψει να έχουμε ένα κατάλογο πολύ πιο αυστηρό για τους στόχους που θα επιδιώκουμε βάσει της ατζέντα της συνοχής. Αντί λοιπόν να εργαζόμαστε περιγραφικά για τα πολιτικά μέσα και να εξετάζουμε το ενδεχόμενο αντίκτυπό τους, κάτι που ούτως ή άλλως το κάνουμε, εφαρμόζοντας τους υπάρχοντες τους μηχανισμούς, αυτό που τώρα προσπαθούμε να κάνουμε είναι να έχουμε στόχους. Στόχους συνοχής, αυξημένη συνοχής, για συγκεκριμένα εντοπισμένα εκ των προτέρων προβλήματα και εκεί ελπίζουμε να αναπτύξουμε πραγματικά δείκτε προόδου και να επιτύχουμε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Συνολικά ελπίζουμε να έχουμε ένα καλύτερο εργαλείο στα χέρια μας. Ως προς τις υπόλοιπες παρεμβάσεις, με ένα-δυο σχόλια αν με επιτρέπετε, θα προσπαθήσω να μην επεκταθώ. Για την καχυποψία, κύριε Μπέρμαν, εσείς το είπατε. Καχυποψία αντί των προτάσεών μα Θα πρέπει να έχουμε υπόψη το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο συζητούμε. Θα Αναφέρω απλώ δύο πτυχέ εδώ. Πρώτα απ' όλα την γενικότερη συζήτηση που ούτω ή άλλω ε, εκτελήσεται στου ακαδημαϊκού κύκλου και του πολιτικού για τον τερματισμό τη βοήθεια. Νέα αντίληψη τη βοήθεια. Όλα αυτά είναι συζητήσει θεωρητικέ που γίνονται. Γίνονται ταυτόχρονα και πρέπει να προσπαθήσουμε να τι ακούσουμε και να συμμετάσχουμε ενεργά. Ξέρω ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε, αλλά και εμείς ε, συμμετέχουμε σε αυτή τη συζήτηση, δεν είμαστε στο περιθώριο. Έπειτα το άλλο σημείο που θέλω να τονίσω είναι ότι υπάρχει και η χρηματοπιστωτική και η οικονομική κρίση που απλώς οξύνει τις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών ιδιαιτέρως. Για το ότι η εμπορική πολιτική είναι καθοριστική σημασία σε κάθε ατζέντα συνοχής, ε, προφανώς. Ναι, η ατζέντα της Ντόχα, οι συμφωνίες και οι διαπραγματεύσεις και όλα αυτά είναι σημαντικότατα. Οι εμπορικέ μα σχέσει αυτέ μα απασχολούν, δεν θα τι εγκαταλείψουμε. Δεν σημαίνει ότι η νέα προσέγγιση θα μα οδηγήσει σε εγκατάλειψη των παλιών μηχανισμών. Ελπίζω ότι ήμουν σαφή ω προ αυτό. Και η τελευταία παρέμβαση για τι αλληλευτικέ συμφωνίε. Κοιτάξτε, διαπιστώνουμε ότι η τοποθέτηση της Επιτροπής είναι πολύ, απέχει μακριά, από, απέχει πολύ από την ε, όλη αντίληψη της δικής μας Επιτροπής. Σίγουρα δεν εξαντλήσαμε το θέμα αυτό. Θα έλεγα λοιπόν να συνεχίσουμε τη συζήτηση σε μια άλλη περίσταση. Έχει περάσει ώρα και για τους διερμηνείς μας. Θα έλεγα αύριο στην συνεδρία των συντονιστών να προβλέψουμε μια επόμενη συνεδρίαση για να συνεχιστεί αυτή τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο νομίζω <clears throat> που πρέπει να μας απασχολήσει. Σας εύχομαι λοιπόν καλό βράδυ και θα τα πούμε αύριο. Είναι και αύριο πολύ φορτωμένη ημέρα, πολύ σημαντική, ελπίζω να σας δω όλου.